Otwieram posiedzenie. Στα πολωνικά. Το πρώτο σημείο στην διάταξη τη σημερινή συνεδριάσεω είναι αυτή η κοινή συζήτηση που αφορά την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Ε, które mamy przed sobą. Wysłuchamy oświadczenia pani wiceprzewodniczącej, wysoki przedstawiciel. Θα ακούσουμε βεβαίω για το πρώτο μας θέμα και τη δήλωση της Λέδης Άστον, της ε, υπάλληλη εκπροσώπου τη Ένωσης για θέματα εξωτερική πολιτικής και θα συζητήσουμε κάποιες πτυχές αυτής της πολιτικής και της πολιτικής Άμυνα. Θα συζητήσουμε επίσης στη συνέχεια την κατάσταση στην Συρία και το στρατόπεδο Ασράφ. Επίση θα συζητήσουμε και την κατάσταση των χριστιανών της Αιγύπτου. Επίσης θέματα άλλα εξωτερική πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σε σχέση με την συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στους διεθνείς οργανισμούς. Τη Δευτέρα ήταν η γιορτή της Ευρώπης, η μέρα της Ευρώπης. Σήμερα δε θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, μια που έχουμε το με κάποιες προκλήσεις, διότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την κρίση, αλλά θα πρέπει και να προετοιμαστούμε και για το μέλλον της μέλουσες κρίσης. Όλες τις κρίσεις που σοβούν και εκτός της Ευρώπης. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις ταραχές σε Συρία και Μπαχρέιν σε την Ισία και Αίγυπτος έγιναν και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε επίσης και ε, τους ε, ε, τέρους μας προς Ανατολάς μια που ξε, μόλις τώρα ξεκίνησε και αυτή η πολιτική Euronest και θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αποτελεσματική η ευρωπαϊκή διπλωματία που να είναι ένα εργαλείο αποτελεσματικό για αυτή την εξωτερική μας πολιτική. Να δούμε πώ θα λύσουμε τα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα μπορεί να γίνει μόνο εάν λάβουμε υπόψη στα σοβαρά τα όσα γίνονται εκτό Ένωση. Επομένως θα πρέπει να δούμε και το θέμα της εκπροσώπησής μας και πώς θα γίνουμε και πολιτική και όχι μόνο οικονομική δυναμική. Και τότε σκητάλη θα πάρει η αντιπρόεδρος της Επιτροπής και είπατε εκπρόσωπος η Λέδη Άστον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα συζητήσουμε τρία θέματα σήμερα και θα αρχίσω εξηγώντα στα αξιότιμα μέλη πώ βλέπω τα πράγματα όσον αφορά τι προκλήσει που αντιμετωπίσουμε και να θίξουμε και κάποιε άλλες ε, πτυχέ όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία ζητήσατε να συζητηθούν ε, σήμερα. Αυτά ακριβώ που σα απασχολούν που θεωρείτε σημαντικά. Καταιγίδε φερίζουν τους ε, γείτονές μας στις χώρες, τις γειτονικές και όπω όπως και με ό,τι εικόνα και να το δούμε όλα αυτά είναι ε, πάρα πολύ ε, ξαφνικά, πάρα πολύ σημαντικά και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Βεβαίω και υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές ε, προσδοκίες για αυτές τις επαναστάσει για το κατά πόσον επομένως κάτι θα γίνει κατόπιν όλου αυτού του αίματο το οποίο ηχήθηκε, κατόπιν όλα αυτά τα προβλήματα και οικονομικά και πολιτικά που επί δεκαετίε σοβούν στην ε, Βόρεια Αφρική και στον αραβικό κόσμο. Όλα αυτά είναι και προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για μας. Αυτές οι ευκαιρίες δεν πρέπει να χαθούν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις πράξεις μας, τις ενεργειές μας. Πρώτα-πρώτα ότι εμείς από πλευράς ε, Ευρώπης ξέρουμε πόσο οδυνηρός, πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος για την ε, ελευθερία, γιατί και ε, εμείς ακολουθήσαμε αυτόν τον αργό και βασανιστικό δρόμο προς την δημοκρατία και την ελευθερία στον 20ο αιώνα και επομένως θα πρέπει να δούμε κατόπιν αυτών των συγκρούσεων το πόσο δυσάρεστο είναι όταν δεν υπάρχει δημοκρατία. Για όταν πάει να δημοκρατία δημοκρατία. Ε, γι' αυτό το, είδαμε με τι ε, ε αυτοκρατορίε. άρα χρειάζεται με ταπεινότητα να δούμε τα πράγματα και να διαπιστώσουμε ότι για την ε, πρόοδο του ανθρώπου είναι βασικό θεμέλιο η δημοκρατία. Επίση. δεν είναι μόνο πολιτική, δεν είναι μόνο εκλογές η δημοκρατία. Είναι παραπάνω. Χρειάζεται επομένως κάτι βαθύτερο. Ελευθερία λόγου, ε, κράτος δικαίου, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελεύθερη δικαιοσύνη και επίσης μια αμερόληπτη ε, διοίκηση. Επίσης χρειάζεται να υπάρχουν πράγματα δικαιώματα τα οποία να ισχύουν στην πράξη, χρειάζεται να υπάρχει συνδικαλισμό και επομένω αυτό το οποίο χρειάζεται να υπάρχουν τα κατάλληλα θεσμικά όργανα και κατάλληλη νοοτροπία. Οπότε μακρόβουνα, μακροπρόθεσμα, αυτό είναι η δημοκρατία και να υπάρχουν επομένω ελεύθερε εκλογέ, να υπάρχει ελεύθερη επιλογή του ποιο θα κυβερνήσει αλλά όλα αυτά είναι τα, τα, τα, τα κατεπίφαση φαινόμενα της δημοκρατίας και για να υπάρχουν αυτά πρέπει να υπάρχει βαθύτερη δημοκρατία. Επομένως μόνο αυτό γίνεται, ε, δεν υπάρχει κανένας είδους ε, εύκολη, έτοιμη, γρήγορη λύση ε, που να οδηγήσει αυτή τη λύση στη δημοκρατία που τόσοι υποθούν. Οπότε από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε το, το ότι θα πρέπει να υπάρχει ανοχή ελευθερία θρησκευτικής πίστης είδαμε τι έγινε στην, στην Αίγυπτο ε, το, η έλλειψη αυτής της ε, ελευθερίας ε, οδήγησε σε, σε, φόβο, οδήγησε σε εγκλήματα. Αυτό θα πρέπει επομένω να ισχύσει παντού και θα πρέπει να κα, ε, καταδικάσουμε όσου θέλουν να χρησιμοποιήσουν σαν μέσο καταστολή τη θρησκευτική πίστη. Θέλουμε ανοχή, ανεκτικότητα και στη Συρία αλλά και στο Πακιστάν, όπω στην Αίγυπτο, όπω και παντού θα πρέπει να προβεί σε κάποιε επιλογέ η Ευρώπη και επομένω να ρίξουμε μια ματιά στο τι γίνεται στη γειτονιά μα. Θα πρέπει να ετοιμαστούμε ώστε να ε, είμαστε στο ύψο των περιστάσεων. Προβαίνουμε σε όλε αυτέ τι ε, δηλώσει και καταδικάζουμε, απευθύνουμε εκκλήσει, παρακαλούμε. Όμω θα πρέπει επίση να λάβουμε και δράση και αυτή η δράση θα πρέπει να λάβει διαφορετικέ μορφέ. Πρώτα πρώτα, όσον αφορά τι ε, κυρώσεις τις οποίε εμεί επιβάλλουμε, ανακοινώνουμε κατά κάποιων καθεστώτων που ε, δεν δίνουν καμία αξία στη ζωή των πολιτών, όταν ε, οι αρχές αρχέ κατόπιν διαταγών σκοτώνουν τον κόσμο. Χθε, γι' αυτό το λόγο, επιβάλαμε κάποιες κυρώσεις στη Συρία, εμπάργκο όσον αφορά το εμπόριο όπλων, ε, περιορισμοί ε, στα ταξίδια εις βάρος αυτού του καθεστώτος και παγώσαμε επίσης και τις συμφωνίες σύνδεσης με τη χώρα αυτή και θα πρέπει να το, το θέσουμε ομά ακριβώς όπως το έθεσα ομά και στον, ε, στον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας. Αυτό το οποίο γίνεται στη Συρία είναι ότι ο κόσμος θέλει κράτος δικαίου, θέλει δημοκρατία. Δεν υπάρχει κανένας είδους συνωμοσία από τα έξω. Όποιος δεν μπορεί να διαπιστώσει αυτό το οποίο σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι θα χάσει την δημοκρατική του νομιμότητα. Και αυτό παθαίνει το καθεστώς της Συρία ε, αμαυρώνεται και προς τα έξω και επομένως όλες αυτές οι απειλές αυτά είναι, είναι πράγματα τα οποία αφορούν το μακρινό παρελθόν που έχει περάσει. Επομένως αυτό μας καίει εδώ πέρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε διάφορες πόλεις της Συρίας ε, εκεί έχουμε ε, αντιπαραθέσεις ε, κατέβηκαν τα τάγκς οπότε και εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αλλάξει η ρότα η κυβέρνηση της Συρίας. Τώρα. Χθε μίλησε επομένω με τον Υπουργό Εξωτερικών και του είπα ότι θα πρέπει άμεσα να ανοίξει τη χώρα στην ανθρωπιστική βοήθεια και μόνο τότε είναι δυνατόν να δώσουμε βάση σε αυτά τα οποία ισχυρίζονται. Τώρα, να δούμε τι γίνεται προς Ανατολάς, τι γίνεται εκεί που ο πρόεδρος Λουκασέγκο στην ε, ε, στην Λευκορωσία ε, παρά τις εκλογές που έγιναν δεν μπόρεσε να ανοίξει την κοινωνία του στη δημοκρατία και στην Ευρώπη και επομένως δεν εκμεταλλεύτηκε την εκλογική του Νίκη όχι μόνο αυτό αλλά και χρησιμοποιεί την βία κατά των ε, διαδηλωτών των ειρηνικών φυλακίζει όλο και περισσότερο κόσμο για πολιτικά αίτια και εμεί έχουμε έρθει σε επαφή με τις οικογένειες αυτών που έχουν φυλακιστούν πολιτικών κρατουμένων και επομένως η μόνη μας λύση είναι και προς την Λευκορωσία να επιβάλλουμε κάποιες κυρώσεις και επομένως ε, και όπως Λουκασέγκο και οι άλλοι από το καθεστώς του επίσης να, να καταλάβουν τι θα πει οι κυρώσεις αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον κόσμο εκεί και την ε, κοινωνία. Τώρα, όσον αφορά το Ασράφ. Στις 8 Απριλίου, είναι τρομερό αυτό το οποίο έγινε. Το καταδικάσαμε ανεπιφύλακτα. Είμαστε κατηγορηματικοί ότι χρειάζεται δυναμική απάντηση ε, και μίλησε επίσης και με την κυβέρνηση του Ιράκ. Φυσικά και δεν είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας, αλλά θα πρέπει ε, να αποστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο στρατόπεδο του Ασράφ. Επόμενο να ε, αναλυθούν ενέργειες, να γίνει μια έρευνα αμερόληπτη, αντικειμενική και έτσι να καταλάβουμε το, ακριβώ το τι έγινε. Όπω όμω γνωρίζετε, αξιόν κύριοι βουλευτέ, από όλε αυτέ τι επιστολέ, τι ατομικέ και τι ε, ομαδικέ που έλαβα από εσά αλλά και από αλλού, η λύση εδώ δεν θα είναι απλή. Έχουμε ένα σωρό σενάρια για μια μακρόπνοη λύση και ε, υπό την ίδια του ΟΗΕ που θα δούμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις και επομένως ε, σας ευχαριστώ όλους όσους πήγατε εκεί, όλους όσους με βοήθησαν ε, θα πρέπει αυτό να το συζητήσουμε και στο Συμβούλιο Εξωτερικών. Θα πρέπει να τα δούμε και με τον είπα εκπρόσωπο για τους πρόσφυγες και με τον ΟΗΕ. Σήμερα έρχεται να έχουμε συνάντηση η, η πρέσβυρα του Ιράκ και ξέρουμε πόσο μας ενδιαφέρει το θέμα και θέλουμε ακριβώς να γίνει μια έρευνα και να υπάρξει ανεπιφύλακτη καταδίκη. Στην Εμένη επίσης Εκεί το Συμβούλιο συνεργασία, κατέβασε κάποιε προτάσει, ο πρώτο Αλέχ επίση ε, ε, ήρθε σε επαφή μαζί μου πρόσφατα και συζητήσαμε για το τι γίνεται με την αντιπολίτευση, τι επαφέ είχε, για το τι προτάσει ε, υπάρχουν στο τραπέζι και του είπα τι, τι πρέπει να γίνει, του είπα ότι όλα αυτά εξυπηρετούν τα δικέ τη δική του χώρα και ότι θα πρέπει να προχωρήσει προ εκείνη την κατεύθυνση. Επίση, συνάντησα στον, ε, στην αποστολή μου στον κόλπο τον βασιλέα του Μπαχρέν και είπαμε ε, και εκεί τα, τα όσα ισχύουν είπαμε για το διάλογο που πρέπει να ανοίξει στη χώρα, στον Παχρέν Όπω είναι τώρα τα πράγματα κύριε Πρόεδρε δεν υπάρχουν απλέ απαντήσει. θέλουμε στον Παχρέν να υπάρξουν δίκες δίκες και θέλουμε να αποφευθούν οι θανατικές καταδίκε. σε όλε αυτέ τι περιπτώσει Πρόεδρε αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρξει κάποια τέτοια άμεση εμπλοκή από πλευρά μα. ασκούμε πιέσει, έχουμε μια ε, ξεκάθαρη προσέγγιση και δεν θα πρέπει να έχουν ψευδεστήσει και με όλου όσου ε, μίλησα ήμουνα επίση ε, ξεκάθαρη για το τι θέλουμε να γίνει και επομένω ε, είμαι στο πλευρό σας και το, το ίδιο θα ισχύσει και για το τι θα κάνουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τη Λιβύη τώρα. Έχουμε κάποιους εδώ στο Κοινοβούλιο που θα ήθελαν βεβαίω να έχουμε πιο δυναμική πολιτική ασφάλειας και άμυνας και έχω να τους πω ότι τελευταίες εβδομάδες αλλά και μήνες εξετάσαμε την διαδρομή που έχουμε κάνει και επίσης διαπιστώσαμε ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πάντως έχουμε δεσμευτεί όσον αφορά τη, την ανθρωπιστική τραγωδία σε συνεργασία με τον ΟΗΕ ε, όλη η Ευρώπη να βοηθήσει τον κόσμο εκεί που έχει ανάγκη ακριβώς όπως κάναμε και για εκείνο τον φοβερό σεισμό στην ε, ΑΙΤ όπου είχαμε πολίτες, στρατιωτικούς ε, ε, το πλοίο του πολεμικού που βοήθησαν και, και ξέρουμε ότι είναι κάτι πάνω από την πολιτική το θέμα αυτής της ανθρωπιστικής βοήθειας όμως δεν θα πρέπει να κινδυνεύουν τη ζωή τους ε, οι, οι ακτιβιστές για, για, την ανθρωπιστική βοήθεια όμως τελικά ε, ο στρατός μπορεί να, να, να, καταφέρει αυτό το οποίο θέλει για να τα κάνει αρκετά γρήγορα ώστε να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και γι' αυτό και ε, μόλις ε, ο ΙΑ αναλάβει ενέργειες και εμείς θα βοηθήσουμε. Πάντως θα πρέπει να κινηθούμε ε, ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά. Και εγώ πρώτη θα παραδεχτώ ότι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Και θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή στη σημερινή συνεδρίαση περισσότερο. Επίσης έχουμε καλύτερη συνεργασία με το ΝΑΤΟ αν έχουν ανταλλαγή πληροφοριών στις επιχειρήσεις, οπότε έτσι εξελίσσονται, βελτιώνονται οι σχέσεις μας και την Παρασκευή τα είπαμε με τον ε, κύριο Γενικό, τον κύριο Ράσμουσεν για να δούμε τι θα γίνει με το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο και επίση ε, συζητήσαμε και για την Λιβύη. Ε, επίση συνεργαζόμαστε με την Αφρικανική Ένωση, την, τον Αραβικό Σύνδεσμο, κύριο Μούσο και τον κύριο Σανόπλου και, και με άλλους παράγοντες. Επίσης και σε σχέση με τον κύριο Βανκιμούν ε, συζητήσαμε για το τι θα γίνει στο Κάιρο και για την συνέχιση που θα δοθούν σε επαφές μας στην Ρώμη και να εξετάσουμε ε, τι θα γίνει, ποιο είναι το μέλλον της Λιβύης, πώς θα υπάρξει διάλογος, σύνταγμα, ε, προετοιμασία για εκλογές. Επίσης έχουμε δύο αποστολές στη Λιβύη κατά τις οποίες συναντήσαμε νέους, συναντήσαμε γυναίκες και όπως είπε ο επικεφαλής του επιτελείου μου είπε ότι για πρώτη φορά συζητήθηκε το θέμα του συντάγματος, ε, συζητήθηκαν κάποια επιχειρήματα, κάποια θέματα τα οποία ποτέ δεν είχαν συζητηθεί και τώρα που πλησιάζει το τέλος του καθεστώτος του Καντάφη θα πρέπει ξεκάθαρα να πούμε ότι πρέπει να φύγει. στην εργασία επίση θα πρέπει να ανοίξουμε ένα γραφείο και να έχουμε άμεση επαφή με τον κόσμο. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία των πολιτών, ε, την προσωρινή κυβέρνηση, τον κύριο Τζεμπρίλ και ε, θα συνεχίσουμε τις επαφές μαζί του ώστε να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που ζητάει εκεί ο κόσμος. Θέλω να τους βοηθήσουμε και όσον αφορά θέματα παιδείας, ε, υγείας, ε, και όσον αφορά τη φύλαξη των συνόρων να τους βοηθήσουμε όπως μπορούμε και επομένως θα πρέπει κυρίως ό,τι και να κάνουμε να βάλουμε υπόψη μας την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια νέα πολιτική γειτονίασης με όραμα, με φιλοδοξίες. Και να είμαστε υπεύθυνοι να δεσμευόμαστε προς ε, τις χώρες αυτές, προς τις γειτονιάζουσες χώρες, αλλά επίσης να είμαστε υπεύθυνοι και όσον αφορά τους Ευρωπαίους. Θα πρέπει να συνεχίσουμε πάνω στις βάσεις που έχουμε βάλει και υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν απαραίτητοι πόροι, όμως υπάρχει κάτι πάρα πολύ βασικό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να βαθίσουν το μέλλον ε, να υπάρχει κινητικότητα των νέων. Πρόκειται για κοινωνίες που έχουν πάρα πολλούς νέους που ποθούν να τους δοθούν κάποιες ε, ευκαιρίες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο να βοηθήσει ε, αυτόν τον κόσμο αυτούς τους νέους και αυτό θα πρέπει να το δούμε με τα κρατημέλη θέλουν ευκαιρίες για να μπορέσουν να πάνε να σπουδάσουν θέλουν και οι γυναίκες ε, επίσης να βοηθηθούν χρειάζονται αγορές για τα προϊόντα τους είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και επίσης Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο ότι με αυτές τις χώρες ε, ε, πάρα πολλά κρατημέλη έχουν ε, ιστορικέ και ιστορικού δεσμού θα πρέπει να αναβαθμιστούν αυτοί οι δεσμοί και για την προσβασιμότητα στι αγορέ και εδώ μπορούμε κάτι να κάνουμε για να του βοηθήσουμε στην οικονομική του ανασυγκρότηση, οικονομική ανάπτυξη γιατί ξέρουμε ακριβώ πόσο αυτέ οι ταραχέ είναι καταστροφικέ για την οικονομία. Κάποιε από αυτέ τι χώρε μόνο εμά έχουν για τι εξαγωγέ του. Οπότε Εάν τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις αγορές τους, αυτό θα κάνει τη διαφορά και έτσι θα υπάρχει εμπιστοσύνη, έτσι θα υπάρχουν αυθεντικές ευκαιρίες και αυτό κυρίως αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να γίνουν όλα αυτά όμως θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη πολιτική βούληση και επομένως έτσι να δεσμευτούμε ότι θα ανοίξουν σε αυτές τις χώρες οι αγορές μας. Να μια πρόκληση, αξιότιμοι βουλευτές, και ε, κυρίω όσον αφορά τη σημερινή οικονομική συγκυρία θα πρέπει να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό τότε ε, και εμείς θα υποστούμε τις συνέπειε ε, τις αποτυχία αυτών των οικονομιών Επίση. Ε, δεν λέω να κάνουμε ενίσχυση οικονομική απευθείας άμεση αλλά κάποιο είδου μόχλευση να υπάρχει υπέρ αυτών των χωρών και αυτό και έχουμε προσχεθεί να κάνουμε. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Αυτό αφορά πάρα πολύ την, την Ισία και 24 Ιουλίου, όπως ανήκει ο Πρωθυπουργός της χώρας, θα τελεστούν εκεί εκλογές. Ε, δεκαδικά ψηφία είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, άρα θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο, να βοηθήσουμε την κοινωνία τους και επομένως να έχουμε υπόψη και μακρόπνους στόχους και τι στρατηγική θα χαράξουμε, αλλά και το τι θα κάνουμε και πώς θα βοηθήσουμε τώρα την Αίγυπτο, την Τινησία και τις άλλες χώρες. Εδώ και τώρα. Γιατί έχουν πολύ σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα και γι' αυτό ήδη αρχίσαμε επαφές με κράτη-μέλη, με χρηματοοικονομικά ε, ιδρύματα για το πώς είναι δυνατόν να βοηθούν αυτές οι χώρες, τι θα γίνει με τα ελλείμματά τους. Ε, δεν έχουν τουρισμό, η οικονομία τους δεν ε, λειτουργεί. Είναι θέματα που καίνε τώρα. Επομένως θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλα αυτά πήγουν τώρα και θα πρέπει ταυτόχρονα και παράλληλα να υπάρχει μακρόπνοη στρατηγική. Αυτά ισχύουν και για την Αίγυπτο, στην οποία μετέβην στις τελευταίες εβδομάδε τρει φορές και συνάντησα του νεαρού ηγέτε τη επανάσταση, συνάντησα και ε, αντιπροσώπους του γυναικείου κινήματο και κυρίω οι γυναίκες ε, θέλουν να δουν του καρπούς των υποσχέσεων που έχουν λάβει, να ακούγεται τη φωνή του. Ε, επίσης ε, συνάντησα την υποψήφιο της, για την προεδρία τη χώρα που και θέλει αυτό να ακούγεται τη φωνή των γυναικών, συνάντησα υπουργού. Ε, τον κύριο συνάντησα και τον ε, Υπουργό Χωροταξίας Ανάπτυξης που έχει όραμα σε σχέση με το, με το, με το θέμα της ε, στέγασης, πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη χώρα και θα πρέπει επομένως με όραμα να δούμε πώς τις υποσχέσεις μας θα τις υλοποιήσουμε προς αυτές τις χώρες και επομένως να υπάρχει κατάρτιση, να υπάρχει παιδεία, ε, υποδομές, να δοθούν ευκαιρίες στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δούμε πώς θα υπάρχει και ασφάλεια στα, στα, σπίτια τα οποία χτίζονται οπότε να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτά που θέλει ο λαός της ε, Αιγύπτου μίλησα και με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας και είπαμε ότι θα συνεργαστούμε όσον αφορά τις προσπάθειες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή να συνεχίσουμε στον τρόπο που έχουμε και να αναπτύξουμε τις σχέσεις με τους ε, συνομιλητές μας θα πρέπει αυτό να κάνουμε του επόμενου μήνες, τα επόμενα χρόνια να βοηθήσουμε και τον κόσμο στις τι ε, προκλήσεις και να λάβουμε υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη μας, τις επαφές μας, τους πόρους μας και όλα αυτά να τα συστρατεύσουμε υπέρ της Αιγύπτου πάντα έλεγα ε, εδώ ότι η υπηρεσία ε, εξωτερικών σχέσεων πρέπει να βοηθάει στην ειρήνη, στην επίλυση των κρίσεων. Αυτό ισχύει για Κωσυφοπέδιο, για Σερβία. Έχουμε την, την ψηφοφορία ε, στον ΟΗΕ. τώρα ακούγεται η φωνή μας. Θέλουμε να δουν τα πράγματα αλλιώς οι ηγέτες στη Βοσνία να ενεργήσουν για το συμφέρον της χώρας και για τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε καλά ότι για την, για την Μέση Ανατολή θα ε, πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες για την ειρήνευση. Έχουμε τόσες δεκαετίες ε, κρίσης και σύγκρουσης, αλλά εμείς με το κουαρτέτο νομίζω ότι δώσαμε κάποια όθηση στα πράγματα. Έγινε η συνάντηση του Φεβρουαρίου και έχουν τους διαπραγματευτές ε, και από τις δύο πλευρές ε, που για πρώτη φορά κάτσαν στο ίδιο τραπέζι στο κουαρτέτο. Είχαμε τη συνάντηση του Απριλίου επίσης όπου και προέβημεν σε κάποια δήλωση για τις θέσεις μας και συνεχίζω να πιστεύω ότι κατόπιν διαπραγματεύσεις θα βρεθεί μια λύση και επίσης θα υπάρξει και μια συνάντηση αυτόν το μήνα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους Παλαιστινίους να αποκτήσουν ένα κράτος ε, και στις 13 Απριλίου ε, συγχαρήγαμε τον Σαγιάτ για, την, ε, για τόσο έχει πετύχει για παιδεία, για υγεία και είπαμε ότι αυτά χρειάζονται τόσο ώστε να λειτουργεί η κυβέρνηση της χώρας και επίσης χαιρετήσαμε τις προσπάθειες συμφιλίωσης. Τα είπαμε τον πρόεδρο Αμπάς. Πρόκειται για μια ευκαιρία τώρα για την ειρήνη αυτό το οποίο χρόνια προσπαθούμε να βοηθήσουμε που και τώρα γίνονται κάποιες σοβαρές προσπάθειες να υπάρξει ενότητα στη χώρα που και αυτή βοηθάει ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια λύση δύο κρατών. Επαφές με είπα με Ισραήλ και λέμε ότι θέλουμε να σταματήσει η βία, να τηρηθούν οι δεσμεύσεις μας και τελικά θα κρυθεί εκ του αποτελέσματος το τι προσπάθειες καταβάλλονται. Επίσης, να δούμε τι θα γίνει με τη φορολογία που βάλει το Ισραήλ στους Παλαιστινίους. Οι χθες της Χαμάς δεν έχουν αλλάξει. Ε, οπότε ένα βασικό θέμα μας προβληματίζει είναι και η ασφάλεια του Ισραήλ. Επίσης, Δεν θεωρώ ότι ο αποκλεισμό της ε, Γάζας και ότι ε, ο ανθρωπιστικός αυτός στόλος είναι η καλύτερη λύση. Χρειάζεται περισσότερη καλύτερη πρόσβαση και να αρχίσει να αναπτύσσεται η οικονομία στη Γάζα. Διότι εκεί η κατάσταση είναι τραγική, ιδίω για τα παιδιά. Έχουμε προτείνει στο Ισραήλ στο πώς μπορεί να υπάρχει από πρόσβαση να δώσουμε ένα μέλλον στην Γάζα και θα πρέπει ο Χαλίτ να μπορέσει να πάει να δει τους δικούς του μετά από τόσα χρόνια. Χρειάζεται πραγματική δημοκρατία, ειρήνη και ευημερία. Και μόνο με θεμελίωση της Δημοκρατία, μπορούμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Έχουμε την εμπειρία αυτές τις χώρε που μα ζητούν βοήθεια να τις βοηθήσουμε. Και οι προτάσει. Προ τα εκεί κατατείνουν με χρήση των πόρων που έχουμε και να δοθούν ευκαιρίες ιδίω στους νέους να ασχοληθούν με τον πολιτικό βίο της χώρας να, να δημιουργηθούν κόμματα, να λειτουργήσουν ακριβώς ό,τι έχουμε κάνει οι χώρες που εκπροσωπούμεθα σήμερα εδώ. Να υπάρχει μια πολιτική διαδικασία, ούτως ώστε να λειτουργήσουν τα κόμματα, η κοινότητα των πολιτών και έτσι να ανθίσει και στις χώρες αυτές η δημοκρατία και είπαμε δεν είναι θέμα εκλογών και ανάδειξη μιας κυβέρνησης. να μπορεί κανείς να μπορεί να λειτουργήσει ένα καθεστώς ε, μια, ένα, ένα πολίτευμα να ανεβαίνει μια κυβέρνηση και να μπορεί να αποχωρεί μια κυβέρνηση όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και όλα αυτά λειτουργούν μόνο όταν υπάρχει δημοκρατία που έχει βαθιές ρίζες γι' αυτό είναι σημαντικό το ότι γίνεται στην ακτή του ελεφαντοστού βοηθήσαμε εμείς όσον αφορά την ανάληψη καθηκόντων του Προέδρου, τον στηρίξαμε σε αυτή τη διαδικασία ανάδειξης και επίσης είναι πάρα πολύ καλό το ότι εύρυθμα διενεργήθηκαν εκλογές στην Νιγηρία και εκεί επομένως θα πρέπει να δούμε ε, μια καλή θετική διαδρομή για, την, για τον κοινωνισμό της χώρας. Πρόοδος σημαίνει αλλαγές. Χρειάζεται όμως για να γίνει αυτό και αποφασιστικότητα. Ζητούνται ενέργειες από την Επιτροπή και από τα κρατημέλη. Άρα και εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε να παίξουμε το ρόλο που μας αναλογεί. Τα φώτα είναι πάνω μας και θα πρέπει να ενεργήσουμε έχοντας κατά νου το μέλλον. και να πείσουμε τους γείτονες όχι μόνο να αρχίσουν τη διαδρομή προς τον εκδημοκρατισμό αλλά και να ολοκληρώσουν αυτό το ταξίδι. Με γρηγόρης, αλλά πάντως θα πρέπει να ευχαριστήσω τους εισηγητές σας και εν κατακλείδη σας αναφέρω ότι είπε μία ανθρωπολόγος, η Μάργαρετ Μίτ, η οποία έχει πει και τη θαυμάζω ότι ποτέ κανείς δεν πρέπει να έχει επιφυλάξεις για το πόσο οι λίγοι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Thank you. Thank you, Lady Ashton. Ευχαριστώ, Lady Ashton. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδελφούς ότι πέραν της εισαγωγικής δήλωσης της Lady Ashton έχουμε να συστήσουμε και συγκεκριμένα τρεις εκθέσεις των συναδελφών, του κ. Αλμπερτίνη, του κ. Γκουαλτιέρη και της κυρίας Μουνίας του Υπενθυμίζω δε ότι προσθέσαμε τη Δευτέρα με την προσαρμογή τη ημερήσια διάταξη και το θέμα τη βία τη βαρό των χριστιανών στην ε, κοινή αυτή συζήτηση. Εκ μέρου των πολιτικών ομάδων τώρα θα λάβει το λόγο ο κύριο ε, Ντόνο, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία είπατε εκπρόσωπε Λίδια Ειρηνικές ήταν οι εξελίξεις ε, ευτυχώ στι περισσότερες ε, χώρες της ε, γειτονική μα περιοχής στην Μεσόγειο και πιο πρόσφατα μέσω μια συμβολικής πράξης το τέλος της περίοδου της εποχής Μπεν Λάντεν διαπιστώσαμε. Εμείς θέλουμε να δεσμευτούμε με καλή βούληση χωρίς αμφιβολία οι δράσει του ΟΗΕ στην Λιβύη μετά από πρωτοβουλία κάποιων κρατών, αρχικών κρατών και ε, ηγετών τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξαν ότι η Ευρώπη μπορεί να ενεργήσει στι δύσκολε στιγμές όταν το επιθυμεί. Είμαστε ωστόσο ένα ε, απαραίτητο διεθνής φορέας ε, με επιρροή στο ύψο του οικονομικού μα κύρου. Η απάντηση είναι αρνητική. Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ο κοντορεβιθούλης τη πολιτική και τη γεωστρατηγική παρά τι μεγαλύτερε προσδοκίε τη Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Εμεί έχουμε στοιχηματίσει σταθερότητα και στην αναπτυξιακή βοήθεια στην Μεσόγειο. Οι λαοί όμω ε, διεκδικούν την πολιτική του ελευθερία και αυτό είναι θεμητό και φεύγουν από τις χώρε τους γιατί δεν μπορούν να περιμένουν για τους ίδιου και για τα παιδιά τους ένα βιώσιμο και αξιοπρεπέ μέλλον. Η ανθρωπιστική βοήθεια που δίνουμε εδώ και κάποιου μήνε είναι χρήσιμη βέβαια όμως, κυρία Αντιπρόεδρε, κύριε, κυρία είπατε εκπρόσωπος, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Αρχίσαμε να βγάζουμε τα διδάγματα από αυτή την εμπειρία. Ελπίζω μετά από τα κύματα μεταναστών που έρχονται στις ακτές μας και που πεθαίνουν στη θάλασσα και ούτε καν ξέρουμε πόσοι πνίγονται, οι χώρες μας πολύ συχνά αντιδρούν ε, μέσω ε, συγκρούσεων, ε, κλεισίματος των συνόρων και αφισβητώντας την τόσο ουσιαστική συνθήκη του Σέγγεν. Όλα αυτά είναι στο ύψος της Ευρώπης, των αξιών της Ευρώπης, ε, των ιδιωδών της. Όχι, δεν το πιστεύω. Το, η ομάδα μου, το ΕΛΚΑ, δεν το πιστεύει και είμαι βέβαιος πως η πλειοψηφία των συναδέλφων σε αυτό το ημικύκλιο δεν το πιστεύει. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα το πρωί συζητάμε με την ΥΠΑ το εκπρόσωπο, διότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, της δώσαμε μια, δώσαμε μια φωνή και ένα πρόσωπο στην Ευρώπη και είναι πλέον καιρός όμως να κάνουμε πιο πρακτικά πράγματα. Αυτό σημαίνει επιλογές και τήρηση αυτών των επιλογών. Ποιε είναι οι προτεραιότητες της Ευρώπης, οι σχέσεις με την Ανατολική και Μεσογειακή της γειτονία, η καταπολέμηση τρομοκρατίας, η λύση των ε, συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή και όλα αυτά ταυτόχρονα δεν είναι εύκολα. Ποιοι είναι οι προνομιακοί μας εταίροι, οι ΙΠΑ, ΕΕ, οι αναδυόμενες χώρες ή και άλλοι. Πώς να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα αφήνοντας το πολιτικό πεδίο στα κράτη-μέλη μεμονωμένα ή μιλώ, ε, όπως εδώ και 60 χρόνια μιλώντας με μια ε, δυνατή και ενωμένη φωνή. Στις εξωτερικές υποθέσεις όπως στην άμυνα και στην ασφάλεια η λύση δεν είναι περισσότερο διακυβερνητική, είναι περισσότερη Ευρώπη. Δεν πρόκειται για περισσότερους, ε, περισσότερη ισότητα σε εθνικό επίπεδο αλλά περισσότερη ενότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μια στερεή πολιτική, εξωτερική πολιτική, μόνο αν, μπορέ, αν επιδιώξουμε με όλο μας το βάρος και το κύρος κάποιους κοινού στόχους θα το επιτύχουμε. Θα πρέπει αυτή η χρονιά να είναι η χρονιά της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ε, ανάπτυξης της Μεσογείου. Αν η Ευρώπη και τα καταφέρει θα, οδηγήσει στην ε, λησμονιά στη λύθη των περασμένων ε, της λαθών. Κυρία Άστον, μη φοβάστε να σας πω τα λόγια του Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου. Έχουμε τέσσερα δις ε, που έχουμε εξοικονομήσει. Μην τα στείλετε πίσω στα κράτη, κάντε ό,τι μπορείτε για να τα χρησιμοποιήσετε για αυτούς τους στόχους. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος Μάρτιν Σούλτς για τους σοσιαλιστές. Κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε κάποιε τάσει για επανεθνικοποίηση πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έπρεπε η συνθήκη τη Λισαβόνα να αποτελέσει. Ε, το βασικό γνώμονα για μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ε, άμυνα και ασφάλεια ότι η συζήτηση λοιπόν αυτή που διεξάγουμε με την υπατή εκπρόσωπο μας υπερθυμίζει για άλλη μια φορά ποιες ήταν οι απαρχές αυτές της προσπάθειας. Και υπήρχαν συγκεκριμένε κυβερνήσει τότε, οι οποίε, σε παραδείγματι, δεν ήθελαν πουδενή τον τίτλο Υπουργό Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και ο όρο ύπατο εκπρόσωπο ή ύπατη εκπρόσωπο. Μαζί με τη φορολογική πολιτική, μαζί με την εσωτερική πολιτική βέβαια και είναι κατανοητό αυτό, η εξωτερική πολιτική είναι ένα από τα ε, στοιχεία του πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας, εθνικής κρατικής κυριαρχίας. Και η μεταφορά της, η εκχώρηση της σε ένα υπερεθνικό οργανισμό ακριβώς αποτελεί ένα θαραλέο αλλά και δύσκολο βήμα. Πάντως εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μαζί με την ύπατη εκπρόσωπο θα πρέπει να διερωτηθούμε ως προς το εξής. Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος είναι ο ρόλος αυτής της Ένωσης ως μεμονωμένου οργάνου στο ε, διεθνές πλέγμα της πολιτικής. Ένα άρθρο της έπατη εκπροσώπου που διάβασα πρόσφατα με εξέπληξε διότι πάνω απ' όλα μάλλον ένα άρθρο σχετικά με την υπατή εκπρόσωπο που επικρίνει την απουσία της υπατής εκπροσώπου από τη διεθνή σκηνή και αυτό το άρθρο προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι πάνω απ' όλα θέλουν να προβάλλουν την εθνική τους κυριαρχία, την εθνική δηλαδή, την, την εθνικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Μονομερός, χωρίς ε, ε, συνεννόηση με κάποιον από τους εταίρους κάποια κράτη λαμβάνουν αποφάσεις τα, οι οποίες ουσιαστικά διαλύουν την Ευρώπη. Λιβύη Φερρυπίν. Δεν υπήρξε πιο ορατή διέρεση της Ευρώπης στην εξωτερική της πολιτική σε μια διεθνή ε, δράση όσο αυτή της περίπτωσης στην περίοδο της Λιβύης. Στις πρωτεύουσες, στις μεγάλες πρωτεύουσες των κρατών της Ευρώπης υπάρχει μια τάση η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεωρείται ως μια ε, συνέχεια με ευρωπαϊκά κονδύλια της εθνικής εξωτερικής πολιτικής. Είτε πρόκειται για Κέντοχσε, είτε πρόκειται για Foreign Office, είτε πρόκειται για Υπουργείο Εξωτερικών τη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανία, η ίδια τάση εκφράζεται. Και εσείς κυρία εδώ, ε, κυρία Άστον, μπορείτε να στηρίσετε στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου εάν σε αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους πείτε ότι ναι, σεβόμεθα τα μονομερή σας συμφέροντα αλλά δεν μπορούν αυτά να ορίζουν την κατεύθυνση εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον δεν εκφράζονται μέσα από τη δική μου και συνενετική βέβαια μαζί σας ε, τοποθέτηση. Ναι, να ανοίξετε γραφείο στη Λιβύη. Διότι εσείς ως είπατε εκπρόσωπος εκφράζετε, εκπροσωπείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μεμονωμένη οντότητα και ε, θα έχετε ως εκ τούτου, ως εκπρόσωπος αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υψηλότερη αναγνώριση και αποδοχή και κύρος από ότι οι μεμονωμένες κυβερνήσεις. Όταν είχαμε πέρσι το φινόπορο Φερρυπίν παρουσία στην μεγαλύτερη έκθεση όπλων της Λιβύης, διεθνή έκθεση όπλων, την παρουσία με μεγάλα στάντ της Ιταλίας, της Γερμανίας, της, Βρετανία, της ε, Βρετανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, όλοι αυτοί πήγαν να πουλήσαν όπλα στον Καντάφη. Στο στρατό του Καντάφη που τώρα βομβαρδίζει τους ίδιους του πολίτες. Επομένως, την αξιοπιστία που χρειάζεται η Ευρώπη θα την εξασφαλίσουμε μόνο με εκείνους οι οποίοι θέλουν να προαγάγουν τη δημοκρατία, οι οποίοι πάνε και ανοίγουν ένα γραφείο αντιπροσωπείας για να στηρίξουν τις προσπάθειες για τον εκδημοκρατισμό, οι οποίοι προσφέρουν τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι όμως με την έννοια της υπαγωγής στην εξουσία των ευρωπαϊκών κρατών κάποιων άλλων κρατών και της προβολής των μονομερών του συμφερόντων, αλλά μέσα από μια συνθήκη, σχέση διμερούς ή πολυμερούς ε, συνεννόηση συμφωνιών διμερών ή πολυμερών σε σχέσεις ισότιμες και σεβασμού. Εταιρικέ σχέσεις δηλαδή. Αυτό σημαίνει η πολυμερων σε σχέσει ισοτιμε και σεβασμου εταιρικε σχέσει, δηλαδη αυτο Αναφερθήκατε στα 3M, Money, Mobility, Market Access, χρήματα, κινητικότητα, πρόσβαση σε αγορές. Θα σας θυμίσω ότι χρειάζεται να συμπληρώσετε και 3C, Coherence, Completeness και Community Method ε, συνοχή, ολοκληρωμένη προσέγγιση και κοινοτική μέθοδος. Αυτά λοιπόν πιστεύω χρειάζονται να χρειάζεται να προβάλλεται και σας διαβεβαιώ για την αμέριστη υποστήριξη της σοσιαλδημοκρατικής ομάδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλά πράγματα μένουν να βελτιωθούν. Για άλλη μια φορά λοιπόν θα ήθελα να επαναλάβω την, την πρότασή μου, πιστεύω και προ όλου του συναδέλφους ε, το απευθύνω αυτό, θα συμφωνήσουμε όλοι. Για τα οράματά σα, για μια κυρία εξωτερική πολιτική εδώ μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχετε πολύ περισσότερου, εταίρου και υποστηρικτέ από ότι στη Σύνοδο των 27 Υπουργών των Εξωτερικών για του οποίου έχω κάθε σεβασμό φυσικά, αλλά βεβαίω έχουν άλλα προβλήματα. Εσεί είστε διπλωματική αντιπρόσωπος μια ολόκληρη υπήρου. Ευχαριστώ, λίγο, Πρόεδρος. Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες τώρα με τον κύριο Κίφερ Χόφστατ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Άστον το Σάββατο είχα μια μακρά συνάντηση με τον νέο Πρωθυπουργό κύριο, της Αιγύπτου, κύριο Σεράφ. Τα συμπεράσματά μου μετά από αυτή τη συνεδρίαση, γιατί ήταν το δεύτερο μου ταξίδι στο Κάιρο τους τελευταίους μήνες, ε, είναι όπως είπατε και εσείς ότι χρειάζεται να βοηθήσουμε μαζικά τις επαναστάσεις αυτές στη Βόρεια Αφρική και κυρίως ε, μετά τα όσα έγιναν στην Αίγυπτο. Πρέπει να σταματήσουμε με τις μικρές μας πατερναλιστικές ε, προσαρμογές τις οποίες έχουμε ανακοινώσει μέχρι τώρα. Μία σύντομη σύγκριση. Το σχέδιο Μάρσαλ τον είπα. Θυμάστε, ξέρετε πόσα χρήματα. 1% του ΑΕΠ ετησίως 162 δις ε, δολάρια. Και εμείς μιλάμε γιατί στην Ευρώπη, τι τους υποσχόμαστε, ένα δις. Όχι 162 δις το 2011, το 2012, όχι ούτε καν το, τώρα θα τους τα δώσουμε, το 2013 λέμε ένα δις όταν θα μπορούμε να τους τα δώσουμε. Νομίζω πως αυτό δεν είναι ε, αξιοπρεπές. Και αυτό που περιμένω εγώ από εσά και από την Κομισιόν, γιατί μιλάμε για χρήματα της Κομισιόν βασικά, δεν είναι τα μεγάλα σχέδια για να αλλάξουμε την πολιτική κοινωνία. Σα. Ναι, αυτό χρειάζεται να το κάνουμε στο μέλλον, αλλά αυτό που εγώ περιμένω είναι όσο γίνεται πιο σύντομα να υπάρξει άμεσα δημοσιονομική βοήθεια προ την Αίγυπτο, γιατί μέχρι το τέλο του έτου δεν έχουν φράγκο και αυτό μπορεί να ε, σημάνει την αρχή μιας αντιεπανάστασης στην, Αίγυπτο. Ε, να ακυρώσουμε το χρέος είτε άμεση βοήθεια δημοσιονομική. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και μια τέτοια είδου ανακοίνωση σήμερα θα ήταν σίγουρα βοηθητική για τους Αιγύπτιους και για την Αίγυπτο. Το Δεύτερο μου μήνυμα αφορά την Συρία. Ας είμαστε ειλικρινεί κυρία Άστον. Η Συρία είναι καταστροφή. Αυτό που συμβαίνει εκεί δεν μπορούμε να το περιγράψουμε άλλως. Είναι η αραβική μεν που γίνεται εκεί. Τους σπάζουν ε, τα τάγκς και οι ελεύθεροι σκοπευτές καθημερινά. 800 έχουν ε, ε, σκοτωθεί μέχρι στιγμής, 8.000 έχουν συλληφθεί. Πολλοί βασανίζονται με τον πιο βίαιο τρόπο για να μαρτυρήσουν τους κωδικούς τους στο Facebook και τις επαφές τους στο Facebook και οι στρατιώτες που δεν θέλουν να πυροβολήσουν τους δικούς τους, το λαό τους, πυροβολούνται οι ίδιοι από τις ε, μυστικές υπηρεσίες και από το, ε, το μυστικό στρατό του Μπασέρ Λασάρφ. Τα όσα συμβαίνουν στη Συρία λοιπόν σήμερα είναι ο Μπασάρ Λασάρφ είναι ο πιο βίος δικτάτορας του κόσμου αν δεν κανείς τα όσα συμβαίνουν στη Συρία. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε σήμερα. Τι να κάνουμε λοιπόν με αυτόν. Όταν βλέπουμε 800 σήμερα, 8.000 άνθρωποι που έχουν φυλακιστεί και εμείς τι κάνουμε. Τι κάνουμε, τους παγώνουμε τις καταθέσεις 13 ανθρώπων και όχι του ίδιου του Ασάντ, παγώνουμε τα περιουσιακά στοιχεία. Μα αυτό είναι γελίο και καθόλου ισορροπημένο και δεν βοηθά να πιεστεί ε, το καθεστώς αυτό για να αλλάξει την ε, πορεία του. 10, τι λέμε, 13, 30 ε, τι είναι ο αδερφός και ο ξάδερφο και ο αρνηψιο του ΑΣΑΦ που είναι στον κατάλογο. Όχι. Εκατοντάδε ανθρώπους πρέπει να βάλουμε στο λίστα όσο γίνεται πιο γρήγορα για να ασκηθεί πραγματική πίεση. Εντάξει, καταλαβαίνω την προσέγγιση σα. Λέτε, ναι, ίσω να αφήσω τον Ασάφ από έξω, απ έξω από το κατάλογο και ίσω αυτό να τον βοηθήσει αργότερα να αλλάξει την πορεία. Εντάξει. Ναι, αλλά πείτε το ξεκάθαρα εδώ πέρα στη συζήτηση. Θέλω να πείτε ότι δίνετε διορία στον ΑΣΑΒ για λίγε μέρε. Αν σε αυτέ τι μέρε δεν σταματήσουν τα όσα γίνονται για την ώρα, επαγώστε τότε τα περιουσιακά στοιχεία το όχι μόνο των 13, αλλά ολόκληρη οικογένεια ΑΣΑΒ. Και όλη την οικογένεια ΑΣΑΔ και να πείτε ε, ε, ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το περιμένω. Χθε είχαμε άμεσα ε, επαφή με τον λαό στη Συρία. Πρέπει να ενισχύσετε τις ποινές, τις κυρώσεις, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να το βάλει κάτω. Να δηλώσετε πως η οικογένεια ΣΑΤ ποτέ δεν θα θεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πραγματικός εκπρόσωπος του Συριακού λαού και ότι θα απολογηθεί για τη συμπεριφορά της. Ο πρόεδρος διακόπτη έχει τελειώσει η ώρα σας. Εσείς αυτό πρέπει να κάνετε, να σταματήσετε αυτήν την αραβική τι Δεν είναι αλήθεια πως δεν παίζουμε ρόλο, παίζουμε πολύ σημαντικό ρόλο και ο λαός της Συρίας περιμένει αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα σήμερα, όχι αύριο, σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Τσόλς Τάνοκ, μεταρρυθμιστές, συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ. Η κύρια εξέλιξη στην εξωτερική πολιτική ήταν η ανάπτυξη τη λειτουργία τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Πρόσφατα, εσεί, κυρία Υπατή, εκπρόσωποι, υποστήκατε πιέσει ω προ τι επιδόσει σα. Ωστόσο, βαρώνει Άστον, δεν θα μπορούσατε παρά να είσαστε όσο. Ε, τόσο μάλλον αποδοτική και αποτελεσματική δουλειά όσο θα το επιτρέπουν τα κράτη-μέλη. Σε αυτό ε, ορίζεται η δική σα εντολή και συμφωνώ απολύτω. Δεν μπορείτε λοιπόν ε, να έχετε ειδική βαρύτητα στο διεθνή, ε, στη διεθνή σκηνή όπως απαιτεί η έννοια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης εφόσον πρέπει να έχετε και την ομόφωνη συμφωνία, την ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών που θα σας στηρίζει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η υπονόμευση εθνικής κυριαρχίας από τις ευρωπαϊκές ε, φιλοδοξίες της, Ευρω... Ε, της διεθνείς φιλοδοξίες Ευρωπαϊκής στην εξωτερική πολιτική. Ενώ τώρα κάποιοι καταγγέλνουν ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή η ευρωπαϊκή πολιτική κινδυνεύει λόγω των εθνικών προτιμήσεων ή φιλοδοξιών. Όπως βλέπουμε σε περιπτώσεις όπως αυτή της Λιβύας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας δεσμεύει Κλείνοντα τον κρουνό των πόρων σε θέματα όπως αυτά της εξωτερικής πολιτικής, όπου θα μπορούσαμε και τον Ευρωπαίο πολίτη να υπηρετήσουμε κάνοντας κάτι το αποτελεσματικό και να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων. Στην περίπτωση της... Ε, ε, Τη ε, Γάζα και των πλοίων που κατευθύνονταν για βοήθεια. Μπορούμε να πείσουμε την Τουρκία ή να πιέσουμε την Τουρκία να σταματήσει να παρεμβαίνει στην υπόθεση αυτή και να προξενεί με υποστήριξη προ του τρομοκράτε. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την ε, Χαμά την ίδια. Πρέπει να περιορίσουμε τη δράση τη. Για δε το στρατόπεδο Ασράφ στο Ιράκ. Τι έχετε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα και τελευταίο μπορείτε να καταδικάσετε τον νόμο Μπαχάρτη ο οποίος ε, ποινικοποιεί την ομοφιλοφιλία την Ουγκάντα. Και κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι βεβαίω και υποστηρίζω τι προσπάθειέ σα για σταθεροποίηση στην ε, Μέση Ανατολή και την Αφρική. Γιατί όμω, όπω υπόθηκε και νωρίτερα, δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο κυρώσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ασάντ, εφόσον δικέ του δυνάμει είναι αυτέ οι οποίε καταστέλουν τι ειρηνικέ διαμαρτυρίε των πολιτών. Ευχαριστώ, Κονβεντήτ. Πράσινη. Mm. Κυρία Υπάτη εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ ήθελα να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις, ε, κυρία Υπάτη ε, εκπρόσωπε. Ε, καταρχήν ο Γκίφερ Χόφστατ το είπε για τη Συρία. Ποιος εμποδίζει στην Ευρώπη να βάλουμε τον Ασάντα στο κατάλογο. Ποια είναι χώρα, ποιες είναι οι χώρες που σήμερα ε, εμποδίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει την μόνη απαραίτητη απόφαση. Μα πείτε το, αν δεν είναι δυνατόν γιατί είναι ο κύριος Βεστεβέλε, ε, πείτε το. Πείτε το, ο κύριος Βεστεβέλε δεν θέλει. Να ξέρουμε δηλαδή πού βασίζονται και πού ασκούνται οι πολιτικές των μένων και των ΔΕ. Γιατί είναι απίστευτο. Δεν θα πούμε όπως το πιστεύει το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι η λύση στα προβλήματα του δεκτάτορα Ασάντ είναι ο Ασάντ. Άμα δεν μας κάνουν να το πιστέψουμε αυτό, είναι απίστευτο. Η λύση στη Συρία θα υπάρξει μόνο άμα ο Ασάντ θα έχει φύγει από την εξουσία εκεί. Αυτή πρέπει να είναι η θέση της Ευρώπης και είναι σαφές ότι ο Ασάντ και όλη την οικογένεια να μπουν σε αυτό το κατάλογο από σήμερα, και αν αυτό είναι, αυτό είναι αδύνατο γιατί χρειάζεται η ομοφωνία, ε, πρέπει να μα πείτε ποιο την εμποδίζει αυτή τη λύση. Πρέπει να το πείτε δημόσια για να γίνει πραγματική συζήτηση στην Ευρώπη. Δεύτερον, ποιο εμποδίζει σήμερα και πώ εμποδίζει το Ισραήλ να πληρώσει του απαραίτητου φόρου στους Παλαιστινίους. Ναι, πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του Ισραήλ, αλλά αυτή δεν εξασφαλίζεται μέσω της δυστυχίας των Παλαιστινίων. Δεν μπορεί να είναι αυτή η λύση. Και τελευταία ερώτηση. 600 νεκροί στις ε, λιβικές ακτές πριν από λίγες μέρες. Ένα σκάφος ήταν κοντά. Είπατε ότι δεν, υπόθηκε ότι δεν ήταν του ΝΑΤΟ. Δεν ήταν το Charles Ήταν υποτίθεται ένα μαλτέζικο σκάφος. Σας ρωτώ, ποιο ήταν το σκάφος και ποιες είναι οι πληροφορίες. Γιατί δεν τους πήγε να τους πάρει, γιατί δεν πήγε να τους σώσει τους 600 πρόσφυγες που έφευγαν από τη Λιβύη. Υπήρχε δίπλα ένα σκάφος. Ε, μην πείτε τώρα ότι τον 21ο αιώνα δεν μπορεί να γνωρίζουμε ποιο σκάφος ήταν, γιατί είναι έγκλημα αυτό. Δεν προσφέραν τη βοήθεια στα άτομα αυτά που κινδύνευαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Λόταρ Μπίσκι. Ενωμένη ε, αριστερά, ο Πρόεδρος. Είπατε εκπρόσωπε. Από τη συζήτηση αυτή θα αποκομίσετε βέβαια και επένους, αλλά και επικρίσεις για τις ορισμένους τομείς. Η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποτύχει έναντι των αραβικών κρατών στο Αφγανιστάν, στο, στην προσπάθεια για επίλυση του Παλαιστινιακού και στις επαφές μας στην ε, άμεση μας γειτονία στη Μέση Ανατολή. Γιατί αποτύχαμε, αποτύχαμε διότι έχουμε την ε, αδυναμία να ε, ενώσουμε 27 διαφορετικές γραμμές ε, εθνικές σε μια κοινή εξωτερική πολιτική, σε μια πολιτική για την ασφάλεια και την άμυνα. Εξωτερική πολιτική λοιπόν σημαίνει εγκατάλειψη της παλαιάς πολιτικής όπου τα κράτη κοιτούσαν μόνο τα συμφέροντά τους και καταπίεζαν μάλλον τα κράτη εταίρους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανοίξει μια πολιτική της εξίσωσης των ίσων δηλαδή συμφερόντων όχι με διπλά μέτρα και σταθμά όχι με στρατιωτικές επιλογές οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τέτοια μεγάλη αποτυχία αυτές τις ε, πολιτικές όταν αποφάσισε το Συμβούλιο Ασφαλείας την ε, στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη, στη Λιβύη, το Κοινοβούλιο σχεδόν πανηγύρισε. Ενώ τώρα βρισκόμαστε όλοι σε αμηχανία, όλοι υπογραμμίζουν σε αμηχανία, εν των εξελίξεων που παρατηρούμε. Τι γίνεται στη σχέση με τις εξελίξεις στη Γάζα, στο Δαρφούρ, πώς προστατεύουμε το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή διαβίωση του κάθε ενός από τους 1,4 δισεκατομμύρια συμπολίτες μας στον κόσμο που έχουν να επιβιώσουν με ένα μόνο δολάριο την ημέρα. Πρόκειται για ένα ερώτημα το οποίο ανησυχεί βαθύτατα την ομάδα μου. Ε, επαναστάσεις στον αραβικό κόσμο έχουν ένα κοινό αίτημα, το αίτημα για δικαιοσύνη, δικαιοσύνη στην κατανομή του πλούτου μέσα στις ίδιες αυτές κοινωνίες, με δημοκρατική συμμετοχή στις πολιτικές αποφάσεις και στις διεθνείς σχέσεις. Η απέτηση αυτή είναι μια απέτηση την οποία θα πρέπει να ικανοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σημαίνει ταυτόχρονα μια κοινή εξέλιξη στο δημόσιο δίκαιο και όχι μία μονομερή και συμφεροντολογική μόνο ερμηνεία του. Ευχαριστώ κύριο Μπέλντερ, Ελευθερία και Δημοκρατία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Ήπατη εκπρόσωπε, θα χρειαστεί να σε δώσω, θέσω κάποιες ερωτήσεις προς την ε, Ισραηλ, Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύραξη. Τι στάση σκοπεύει να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το Σεπτέμβριο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι Παλαιστίνοι από ό,τι φαίνεται θέλουν πλέον να κηρύξουν κράτος. Τη δε προηγούμενη εβδομάδα διαπιστώσαμε ότι η Χαμάς δεν θέλησε να ε, υποκύψει στις απαιτήσει ε, που είχε ορίσει η τετραμέρης. Θα ήθελα λοιπόν πολύ ξεκάθαρα να πω ότι η Χαμάς έχει θέση μόνο σε έναν κατάλογο, στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί είναι εγγεγραμμένη και εκεί θα πρέπει να μείνει. Πώ σκοπεύει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να, να, χειριστεί την υπόθεση αυτή. Δεν μπορούμε μόνο με μορομερεί εκφράσει ε, ευχολογίων να λύσουμε τα προβλήματα. Μόνο μεγάλη ζημιά στι Ισραηλινοευρωπαϊκέ σχέσει μπορούμε να προκαλέσουμε και δεν πρόκειται να βοηθήσουμε βέβαια καθόλου στην ειρηνευτική διαδικασία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο συνάδελφο Αλμπερτίνη. Γκαμπριέλα Λεμπερντίνη. Εγώ προτείνω να μοιράσετε το ομιλία σας σε δύο τμήματα. Τέσσερα λεπτά στην αρχή και δύο λεπτά στο τέλος της συζήτηση. Για να ολοκληρώσετε. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε είπατε τι εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα της εξωτερική πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας είναι ακόμα πιο σημαντική σε αυτή την ιστορική στιγμή που χαρακτηρίζεται από ε, μια εξαιρετική περίοδο διαμαρτυριών που ξεκίνησε από την Μεσόγειο, την Νότια Μεσόγειο και έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την ε, Ανατολή. Ε, αυτή επεκτείνεται και στη ζώνη της Αραβικής Χερσονήσου. Για όλα αυτά εμείς θα πρέπει να αποτελέσουμε το αντιχείο για όλες τις δημόσιες φωνές που κραυγαλαία ζητούν και με τον κίνδυνο της ίδιας της ζωής τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την έναρξη δημοκρατικών διαδικασιών που θα ε, αποσυνθέσουν τα σημερινά καθεστώτα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να υποτελέσουμε έναν πρώτη τάξη συνομιλητή μέσω της Λέδης Άστον αλλά και για την ε, διαδικασία ελέγχου των ε, δημοσιονομικών σχέσεων μέσα στο πλαίσιο της, της ΚΕΠΑ. Ε, στην πρώτη φάση θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι σχέσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ξεκινώντας ε, μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής μετά την Λισαβόνα. Πολύ σημαντικό είναι και το θέμα της ε, πολυμερούς εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινώντας με το νέα υπεξυπηρεσία ε, εξωτερικών υποθέσεων που επιτέλους έχει γίνει πραγματικότητα. Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ικανοποίησή μου μετά από τις εξελίξεις της τελευταίας συνέλευσης ε, του Ηνωμένων Εθνών που δεχόμενη τα όσα ορίζει η συνθήκη της ε, Λισαβόνας δέχτηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέλος μέσα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Προσπαθούμε να δώσουμε όσο γίνεται καλύτερη θέση στην Ένωση, ε, τονίζοντας την έκθεση, όπως είναι σωστό, το μεγάλο κύμα ε, λαϊκής διαμαρτυρίας στην την Ισία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, τον Μπαχρέιν, την Ιεμένη, που λαοί που ζητούν πολύ συγκεκριμένο συγκεκριμένα πράγματα και επιπλέον είδαμε την ισχυρή διατλαντική συμμαχία και τις ε, τεράστια σημασία σχέσεις μας με τη Ρωσία. Διεύρυνση όσον αφορά την στήριξη των ε, δικαιωμάτων του πολίτη, διπλωματικές σχέσεις με τις ε, χώρες BRIC, Αραβοϊσραηλινή σύραξη. Είναι κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα της έκθεσης τα οποία υποβάλλω στην προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Επόμενος συζητητής είναι ο συνάδελφος Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη και σας κάνω την ίδια πρόταση κύριε Γκουαλτιέρη να κρατήσετε δύο λεπτά για το τέλος της συζήτησης. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, αντιπρόεδρε. Ε, η πολιτική ασφάλειας ε, και κοινή άμυνας ε, διανύει πολύ, πολύ ευαίσθητη κατάσταση. Ακριβώ τη στιγμή που το διεθνές σύστημα επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ένα αξιόπιστο ρόλο για την ασφάλεια, ακριβώ όταν η ευρωπαϊκή κίνηση στηρίζει τη δημοκρατία και, όχι, και δεν εξάγει δημοκρατία, αυτό είναι η πιο κατάλληλη στάση που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε. Ακριβώ στη φάση που η οικονομική κρίση καθιστά δύσκολη την πορεία προς μια κοινή άμυνα και όταν ε, την ίδια στιγμή η συνθήκη της Λισαβόνα προσφέρει νέα μέσα για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ακριβώς δηλαδή τη στιγμή που θέλουμε να κάνουμε ένα άλμα ποιοτικό και που αυτό είναι απαραίτητο αλλά και δυνατό να γίνει, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα φαίνεται να τρίζει επικίνδυνα και κινδυνεύει ε, να περιορίσει την ε, υλοποίηση των προσδοκιών μας και των φιλοδοξιών μας για την ΚΕΠΑ. Ε, εμείς ε, προσπαθούμε να δώσουμε πιθανές λύσεις και απαντήσεις. Για την λιβική κρίση δεν περιοριζόμαστε στο να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας για την αδυναμία της Ένωσης να ορίσει μια κοινή θέση και να προβεί σε κοινέ δράσεις και να περιορίσει την εντολή προς την είπατε εκπρόσωπο. Εμείς θεωρούμε πως είναι η στιγμή για μια ευρωπαϊκή πολιτική κοινωνική πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει πάυση του πυρός και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια δημοκρατική μετάβαση στην οποία θα συμμετέχουν όλοι. Είναι προφανές ότι η στρατιωτική παρέμβαση του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα και είναι, συχνο... Ε, και είναι σημαντικό το να γίνει σεβαστή η εντολή του ΟΗΕ χωρίς να γίνει δυσανάλογη χρήση της, ε, των δυνάμεων και της ε, βίας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες για να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους ε, πολίτες που είναι υποεπίθεση, που τελούν υποεπίθεση, καλά και να βοηθήσουμε στην ε, ανάπτυξη της δημοκρατίας στη Λιβύη. Ωστόσο, η υπόθεση της Λιβύης απαιτεί πιο βαθύ προβληματισμό. Είναι σαφές ότι η βασική ευθύνη για το μέλλον της Ευρώπης για την ασφάλεια και την άμυνα είναι ε, βαραίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου και ο πρόεδρος του οποίου είναι υπεύθυνοι για την εκπροσώπησή μας. Ε, εγώ θέλω να τους πω ότι η διμερή συνεργασία και ο εθελοντισμός δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ε, ε, το, τον πυρήνα, τον πολιτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο δεν μας πείθει, όχι μόνο γιατί είμαστε υπέρ της απόλυτης στήρισης της συνθήκης, αλλά και γιατί μια τέτοια επανεθνικοποιημένη πολιτική δεν είναι κατάλληλη ενώπιον των προκλήσεων που έχουμε ενώπιον μας. Εμείς ζητάμε στρατηγικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, του ζητάμε να ακούσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, να επεξεργαστεί μια γνήσια στρατηγική εξωτερικής πολιτικής, να συγκαλέσει έκτακτη συνάντηση, ε, διάσκεψη κορυφή για την ασφάλεια και την άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί σα ζητάμε, κυρία Άστονα, να οδηγήσετε τα κράτη-μέλη στη συνεργασία και να χρησιμοποιήσετε τι διάφορε αρμοδιότητέ σα για να ενισχύσετε το ρόλο τη ΚΕΠΑ και τη εξωτερική πολιτική τη Ένωση. Ε, γι' αυτό και η υπηρεσία εξωτερική δράση είναι πολύ σημαντική ε, για το ρόλο τη. Έχουμε υποβάλει διάφορα διάφορες ε, προτάσεις με βάση το Crisis Management Board και αυτό βλέπουμε πως ήδη δημιουργείται. Ε, η υπόθεση της Λιβύης ε, αποδεικνύει επίσης ε, την ακαταλληλότητα των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνατοτήτων πέρα από την, παρά την γενική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών όλων των κρατών μελών. Η, ενω, η αυτό είναι γνωστό. Θα πρέπει να υπάρξει μόνιμη συνεργασία, ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς της άμυνας, ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης, ενίσχυση των κοινών δυνατοτήτων των ελέγχου ε, ε, και και διαχείρισης ξεκινώντας με τη δημιουργία ενός ε, μόνιμου επιχειρησιακού γενικού επιτελείου. Ε, όλα αυτά τα θέματα για την, πολιτική, την εξωτερική πολιτική ασφάλειας αλλά και εσωτερικής ασφάλειας εμείς διατυπώνουμε διάφορες συγκεκριμένες προτάσεις και θεωρούμε ότι από αυτή τη βάση οι βασικέ ευρωπαϊκέ ομάδε είναι ενωμένε και για αυτή τη συνεργασία θέλω να ευχαριστήσω του και ηγητέ και του συντονιστέ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να υποστηρίξει την ανάπτυξη μια ε, ΚΕΠΑ που θα, που θα συνδέεται με την ε, εξωτερική δράση της Ένωσης ε, και ελπίζουμε κυρία Άστρο να μας δώσετε πιστικές απαντήσεις με τα λόγια αλλά κυρίως με τις πράξεις. Ο πρώτος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε συνάδελφε. Σας υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για αυτή την έκθεση του κύριου στον την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας και έχουμε επίση και την έκθεση ε, Γκουαλτιέρη. Ε, για την ε, πολιτική αυτή σχέση με την Λισαβόνα και έχουμε επίσης και την τελευταία ε, έκθεση που την έχει συντάξει η κυρία Μαρία Διορκήθα για την Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμιο παράγοντα σε πολεμικούς οργανισμούς. Έχετε το λόγο κύριε Συγήτρια, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Από πλευράς στρατιωτική, είναι πολικό ο κόσμος ε, από άλλη πλευρά είναι, είναι μονοπολικός ε, και από, και από μια άλλη όψη να τα δει κανείς τα πράγματα είναι πολύ, πολύ γιατί πρόκειται για μια παγκοσμιοποίηση η οποία ε, έχει δημιουργήσει διάφορα κέντρα εξουσίας και έχουμε επομένως γι' αυτό ένα σωρό οργανισμούς, διεθνείς θεσμούς ε, έχουμε το, το G20, το G8, G7 κλπ, κλπ. Οπότε το θέμα είναι τώρα τι μεταρρυθμίσεις θα γίνουν για αυτούς του διεθνείς ε, οργανισμούς, τους παραδοσιακού. Έχουμε αυτό το πλαίσιο επομένω όπου όλα αλλάζουν και έχουμε και την ε, μεταβαλλόμενη νομική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι σε, σε αυτό το τοπίο ο ρόλος μας. Ποιο είναι ο χώρο που πρέπει και καλείται να καταλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τι πολυμερεί επαφέ για να μπορέσει να ασκήσει τον ρόλο που τη απονέμουν οι συνθήκε και ε, ε, αυτά τα οποία προσδοκούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι Ευρωπαίοι. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ε, σχετικό ψήφισμα του, του, του ΟΗΕ που επιτρέπει να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εργασίες της Γενικής Ελεύσεω του ΟΗΕ. Αυτό ήταν μια επιτυχία. Αυτό είναι ένα γεγονός ιστορικό. Μπράβο σας κυρία στον συγχαρητήρια. Όμως έχουμε τις σχετικές διαπραγματεύσεις σε σχέση με το ψήφισμα του 1973 και θα πρέπει να δούμε πώς θα ε, επικαιροποιήσουμε την εκπροσώπησή μας η οποία είναι προς το, προς παρόν ε, κατετμημένη ε, και κάθε φορά άλλα πράγματα κάνουμε όσον αφορά τις διάφορες συμφωνίες τις οποίες έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι 250 περίπου οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στα διάφορα διεθνή φόρα και θα πρέπει να δούμε στους, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς θα είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί στην εκπροσώπηση ε, σε σχέση με ε, το πώς εσείς και η εξωτερική υπηρεσία θα συνοείται με την Προεδρία της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Και επίσης με την, την ε, κυκλικά ανασώμενη κάθε φορά Προεδρία ούτω ώστε να μπορέσει να αναδειχθεί ο διεθνής ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς. Εκεί που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την συνάντηση κορυφής της Κοπενχάγης. Εκεί δόθηκε ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Εκεί υπήρχε κακοφωνία. Εκεί δεν βγήκε τίποτα καλό όσον αφορά την εκπροσώπηση. Όμως στον ΠΟΕ και στον ΦΑΟ εκεί η εκπροσώπησή μας είναι παράδειγμα προς έχουμε επίσης ε, κάποια δυσλειτουργική συμμετοχή των ε, Προεδριών. Έχουμε και το άρθρο 34 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον συντονισμό ε, για το Συμβούλιο Ασφαλείας, για τον ΟΗΕ, όσον αφορά την παρουσίαση των θέσεων της Ένωσης. Εκεί επομένως είναι εντυπωσιακή δυσλειτουργία όπως ακριβώς τα είπε και ο κύριος Σουλς. Επίσης ε, μας αναφέρατε το πώς προσπαθείτε να πείσετε τα κράτη-μέλη για να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τον ρόλο που της αρμόζει για να ασκεί μια αυθεντική εξωτερική πολιτική. Να μπορέσουμε ε, να, να, να καταφέρουμε το σωστό ποτάμι να μην γυρίσει πίσω και να πάμε προς επανεθνικοποίηση εξωτερικής πολιτικής. Πάντως, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να λάβουν τις ευθύνε του τα κράτη-μέλη ε, και εσείς επίσης να ε, μπορέσετε να στρατευτείτε με την υπηρεσία σας για να μπορέσετε να καταφέρετε να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης, να μπορέσει να υπάρχει εκλογήκευση ε, σε αυτόν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια που τώρα ζούμε ιστορικές στιγμές, μια που θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πρωτοπόρα. Στη Βεγγάζη είπαμε ότι θα ανοίξουμε ένα γραφείο εκπροσώπηση. Ε, το Κοινοβούλιο συμφωνεί, θα σας ε, στηρίξει και θα πρέπει το νωρίτερο δυνατόν να καταφέρουμε να υπάρχει μια εκπροσώπηση ε, η οποία είναι σωστά διαρθρωμένη και εκλογικευμένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Το ρόλο τώρα έχει η Λέδη Άστον, η Αντιπρόεδρος και η Πατήκη Πρόσωπος. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Κύριε Πρόεδρε, ένα από τα στοιχεία που προβάλλονται σε όλες τις ομιλίες των αρχηγών ομάδων και ότι ο κύριο Στάνοκ υποστήριξε ότι ποτέ δεν ήταν υπέρ της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, ζήτησαν όλοι λοιπόν μια ενοποιημένη δράση. Συμφωνώ. Δεν υπολείπομαι φιλοδοξιών ως προς το τι μπορεί να γίνει η Ευρώπη. Εκεί που έχω πρόβλημα είναι το τι είμαστε τώρα έχω ένα αστείο που συνήθω λέω ότι όταν ε, πέρασε η συνθήκη μου έδωσαν το χαρτί της συνθήκης, το, το κείμενο και ένα μολύβι και με αυτού του πόρου ξεκίνησα τη δουλειά μου. Αλλά έστω και αν είναι αστείο αυτό δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Πάντω βλέπω εδώ να εκφράζονται φιλοδοξίε με μεγάλο ενθουσιασμό να υποστηρίζετε μια κοινή εξωτερική πολιτική. Πλην όμω πρέπει να πείσουμε και το Συμβούλιο, το Συμβούλιο των Υπουργών Αμήνη, των Υπουργών Εξωτερικών, όλα αυτά πιστεύω ότι προχωρούν, δείχνουν ότι προχωρούν όλοι με την ίδια φιλοδοξία και αυτό δεν εκπλήσει κανέναν είτε ε, ε, σε κάθε κράτος μέλος είτε σε επίπεδο υπουργών βλέπουμε ότι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί περισσότερο αποτελεσματική, όπως θα θέλατε εσείς, όπως θα ήθελα και εγώ, και αυτό κυρίως με περισσότερη φιλοδοξία. Είτε πρόκειται για κυρώσεις, όπου χρειάζονται 27, ομοφωνία δηλαδή, είτε με, ως προς την προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε για να υποστηρίξουμε χώρες όπως η Αίγυπτος, την Ισία κτλ. Όπου όπως είπε και ο κύριος Φιωρχόφστατ χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση, να κινηθεί, να αλλάξει στρατηγική και να χαράξει μια νέα φιλοδοξία μακροπρόθεσμα αλλά και πρόθεσμα να μας επιτρέψει να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν αλλαγή νοοτροπία. Ουσιαστικέ αλλαγέ. Είμαστε στο δρόμο. Δεν έχουμε φτάσει. Χωρί να παραπονιέμαι, λοιπόν, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ε, βλέπω τα πράγματα ρεαλιστικά. Ε, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα και μπορείτε να με πιέσετε όσο θέλετε να κάνω περισσότερη δουλειά πιο γρήγορα. Πολύ ευχαρίστω να ε, υποκύψω σε αυτές τις πιέσεις αλλά μην με κατηγορήσετε για απουσία φιλοδοξίας, για απουσία οράματος μην με κατηγορείτε ότι δεν λέω ξεκάθαρα στο Συμβούλιο των Υπουργών ε, ή στον τύπο ακόμη ποιε είναι οι προθέσεις μου, οι φιλοδοξίες μου, το όραμά μου γιατί θεωρώ πράγματι ότι μπορεί η Ευρώπη να είναι πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι είναι τώρα αλλά πρόκειται για ένα δρόμο τον οποίο πρέπει όλοι μαζί να χαράξουμε και είναι δύσκολο πράγματι τα επιμέρους κράτη-μέλη και οι επιμέρους, ε, τα εκλογικά σώματα τα επιμέρους να δεχθούν να δουν αυτή την πραγματικότητα με το φακό του ευρωπαϊκού συμφέροντος και όχι μέσα από το εθνικό πρίσμα. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Ντόλ ε, ότι η τρομοκρατία, η γειτονία, η διαδικασία για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή είναι ένας κύριος στόχος για την τρέχουσα χρονιά και, πρέπει, και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να πούμε ότι η προσπάθειά μας στη Λιβύη είναι ακριβώς να φέρουμε μαζί και την αραβική, ε, τον Οργανισμό Αναβικής Ενότητας και τα Ενωμένα Έθνη και τις περιφερειακές οργανώσεις ώστε να συμπράξουν όλοι αυτοί. Εκείνη η δυσκολία όμως. Πώς θα φτάσουμε μέχρι το σημείο όπου θα αποχωρήσει ο κατάφυκιο, που θα γίνει διάλογος δημόσιος και θα δει ο κόσμος ξεκάθαρα μια εικόνα να διαμορφώνεται. Είναι δύσκολα όλα αυτά και χρειάζεται να έχουμε εμείς ενωμένο μέτωπο. Ο κύριος Σούλτς είπε ότι θα είναι μακρύς ο δρόμος. Συμφωνώ. Πολλά ακόμα μένουν να γίνουν. Και θα πρέπει η ε, οικοδόμηση αυτής της δημοκρατίας, αυτών των δημοκρατιών να πραγματοποιηθεί. Ομολογώ βεβαίω ότι θα είναι ένα μακρόπνο όραμα. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Χρειάζεται ακόμη περισσότερη συνοχή, ακόμη καλύτερη συνεργασία, διαφανή, ε, προσδιορισμό των στόχων που ξέρω ότι απαιτεί το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ σε όλα αυτά. Λοιπόν, συνεχίστε να μου ασκείτε πίεση, αλλά να ασκείτε πίεση και στα κράτη-μέλη. Ένα Marshall Plan, λοιπόν, ένα σχέδιο Marshall. Ε, αυτό που είχε γίνει με τα αρχικά 13 δισεκατομμύρια δολάρια το 1948 που εξασφάνισε ο Μάρσαλ από το Κογκρέσο ήταν ένα καλό πρότυπο. Πρότυπο διότι μπορούμε να πούμε ακριβώς τι έγινε. Είτε ήταν δάνεια, είτε ήταν υπηρεσίες, είτε ήταν επιστηστική βοήθεια. Ο Μάρσαλ μπόρεσε αυτό να το, ποσό να το κατανείμει σε διαφορετικές ε, υπηρεσίες ε, που μπορούσε να προσφέρει. Ε, δεν μπορούμε βέβαια να ακολουθήσουμε ακριβώ το ίδιο μοντέλο, αλλά μπορούμε να το παρακολουθήσουμε κατά κάποιο τρόπο και να εμπνευστούμε από αυτό. Και ιδιαίτερα πρέπει να συζητήσουμε τι χώρε με τι οποίε έχουμε αυτέ τι ιδιαίτερε σχέσει και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ επίση με την έκταση τη βία στη Συρία φιλοδοξίες, οι φιλοδοξίες δεν μας λείπουν ως προς την αντιμετώπιση του προβλήματος Συρίας. Η λίστα αυτή του ε, παγώματος των λογαριασμών ξεκίνησε με 13 άτομα. Είπατε και εσείς κύριε Κονπεντήτ γιατί δεν είναι ο Ασάντ. Ε, δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος ήταν υπέρ ή όχι και κατά. Πρέπει ό,τι κάνουμε να καταλάβετε ότι το έχουμε κάνει με δεδομένη την κατάσταση μέσα στην οποία κινούμεθα. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να ξεπεράσουμε κάποια όρια. Πάντως είμαι πεπισμένη και από αποφασισμένα στους ότι μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση στη Συρία και με τον κύριο Μουαλάμ, τον Υπουργό των Εξωτερικών που συνομίλησε χθε, προσπάθησα να του εξηγήσω ότι η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο και κλείνει πλέον το παράθυρο τη ευκαιρία. να αλλάξει πορεία η κυβέρνηση και να μετατρέψει την πολιτική της, να αλλάξει πολιτική. Κύριε Τάνοκ, μιλήσατε εσείς για την υποστήριξη του 27, για το πόσο θα θέλατε να υπάρχει ε, να υπάρχει μια απελευθέρωση στις δυνατότητές μας να αναλάβουμε δράση, πως η Επιτροπή μας δεσμεύει και δεν μας δίνει αρκετούς πόρους. Ναι, δεν υπάρχει όμως αυτό ζήτημα. Το θέμα είναι οι φιλοδοξίες μας να υλοποιηθούν στην πράξη. Για να ανοίξω μια υπηρεσία, μια αντιπροσωπεία στις, στην Μπεγκάζη ή το Ιράκ που συστήθηκε νωρίτερα σήμερα, χρειάζομαι τους σχετικούς πόρους και πρέπει κάπου να τους αναζητήσω. Και βέβαια με πιο αποτελεσματική και ουσιαστική ε, αποτελεσματική χρήση αυτών των πόρων που έχουμε στη θέσή μου, αλλά και ε, αναζητώντας νέους σπόρους. Μιλήσαμε επίσης για τα πλοία της βοήθειας προς τη Γάζα. Το κλείσαμε το θέμα αυτό, όπως μιλήσαμε και για τις συνομιλίες μεταξύ Φατάχ και Χαμάς. Έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει αποχαρακτηριστεί η Χαμάς, δεν έχει αλλάξει χαρακτηρισμό δηλαδή απλώς. Υποστηρίζουμε την πρόοδο με βάση την οποία θα μπορούσε ο πρόεδρος Αμπάς να, βοήθει, να βοηθήσει η κυβέρνηση αυτής της Χαμάς να ε, ενωθεί με την Φατάχ και να συμπράξει για το καλό του Παλαιστινιακού λαού με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα όχι υπερβολική ισοδεξία. Παρακολουθούμε την κατάσταση. Θα ήθελα επίση να κάνω κάποιε παραπομπέ στι παρατηρήσει του κύριου Μπίσκη, ο οποίο μίλησε για του πιο φτωχού του κόσμου. Μιλήσατε για μια διαβίωση συνθήκε αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι με του στόχου για τη χιλιετία, αν του στόχου τη χιλιετία, προσπαθούμε και με τη λυπή βοήθεια να βοηθήσουμε ακριβώ την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Και χωρί να θέλω να σα καθυστερήσω περισσότερο, θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Αλμπερτίνη και την έκθεσή του. Παραθέτω λοιπόν από το κείμενο αυτό, γιατί ο κύριος Αλμπερτίνη μιλάει για συνοχή και λέει ότι η συνοχή απαιτεί πρώτα απ' όλα πολιτική βούληση εκ μέρου των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των διαφόρων ε, προβλημάτων. Ναι βεβαίως ξέρουμε ότι αν πρόκειται να υλοποιηθεί 100% η συνθήκη τη Λισαβόνα χρειάζεται, αυτό το λέει και ο κ. Αλμπερτζίνη, ουσιαστική χρηματοδότηση αυτών των στόχων. Και συμφωνώ λοιπόν με τον εισηγητή σε πολλά σημεία, αλλά ιδιαίτερω ω προ το ότι πρέπει με αποφασιστικότητα να προβάλλουμε τι αξίε μα και να διαθέσουμε και τα σχετικά μέσα για την υλοποίηση αυτών των αξιών. Και θα ήθελα να ενισχύσουμε το διάλογο που έχουμε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι το ζήτημα του χρόνου. Πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε κατά το βέλτιστο δυνατό ε, σημείο το χρόνο που έχουμε να συνομιλούμε μαζί. Για τον κύριο Γουαλτιέρη, συζητήσαμε χθε νομίζω πολύ καλά μαζί. Ε, ιδιαίτερα συμφωνήσαμε ω προ το pooling and sharing, ω προ την διάθεση, συλλογή και διάθεση πόρων. Θα πρέπει γι' αυτό να το δούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πω μπορούμε του πόρου Ευρωπαϊκή Ένωση να του αξιοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά. Είναι μια πολύ απλή ιδέα αυτό το pool and share, αλλά είναι μια πολύ, ένα πολύ γερό μέσα, ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Έχουμε, επί παραδείγματι, δει την ε, ε, χρησιμότητα του pooling and sharing στους στρατιωτικούς πόρους. Πιστεύω ότι με, βάση, με έμπνευση αυτό το δεδομένο μπορούμε να προχωρήσουμε και αλλού. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα, σε παραδείγματι, που μπορεί και πόρους να εξοικονομήσει και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις σε κάποια από τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει από τις πρόσφατες εβδομάδες γιατί στη Λιβύη. Την ε, κυρία Μουνής Δεουρκουίζα θα ήθελα να πω ευχαριστώ πολύ για την έκθεση, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και σας διαβεβαιώνω για άλλη μια φορά πως είμαι ε, αμέριστη υποστηρίκτρια της, δράση ε, δράσης αυτής της παρουσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οργανισμού, οργανισμούς της αποφασιστικής μας ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τους ομιλητές που έλαβαν το λόγο στον πρώτο αυτό γύρο της συζήτησης και περιμένω να ακούσω και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε. Έχουμε επίσης και μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Ο κύριος ε, Γιούρκ Λάχτφρετ ήταν ο εισηγητής, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω να προ... τα είπα καλά στα πολωνικά. Όταν ε, μιλούμε για την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης και δει το ρόλο της Ευρώπης στο διεθνή σκηνικό, στη διεθνή σκηνή, ε, βλέπουμε νομίζω ότι πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα. Αλλά θα μπορούσαμε να επενθυμίσουμε και μια αντίστοιχη άλλη πολιτική, όπου το έχουμε καταφέρει αρκετά καλά, την εξωτερική πολιτική εμπορίου. Η εξωτερική πολιτική, η πολιτική εξωτερικού εμπορίου, λοιπόν, είναι μια πολιτική στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει ε, μεμονωμένα δράση και εκπροσώπηση των κρατών μελών στι διεθνεί σχέσει Χωρί να ε, βρίσκεται μέσα αυτή τη διαλκυστίνδα των διαφορετικών και αντικρουωμένων ε, συμφουρώντων. Και εκεί που είμαστε ενωμένοι λοιπόν είμαστε και ισχυροί στην εξωτερική μας, ε, στο εξωτερικό μας εμπόριο. Έχουμε μπορέσει να πείσουμε πιστεύω και τους εταίρους μας ότι και εκείνοι υποφελούνται από τα στοιχεία και τα ιδεώδη τα οποία γνωρίζουμε εμείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελεύθερο εμπόριο, την ελεύθερη οικονομία της αγοράς, την ε, τις του κράτους δικαίου. Αυτά σημαίνουν ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στη, μέσω των εξωτερικών μας εμπορικών ε, σχέσεων να βοηθήσουμε και άλλα κράτη να γίνουν πιο δημοκρατικά, να προχωρήσει το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ πολύ και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στον κύριο Λισεκ. Για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να απευθυνθώ στον κύριο Γκουαλτιέρη καταρχήν για να τον ευχαριστήσω για τη σκληρή δουλειά που έκανε. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του και με τους υπόλοιπους σκιώδης συζητητές ε, και ε, να σας πω ότι ήταν μια δύσκολη έκθεση στρατιωτική, αλλά η δική μας συνεργασία ήταν πολύ ειρηνική. Κυρία, είπατε εκπρόσωπε, στην πρώτη σας παρέμβαση μιλήσατε για τις συγκρούσεις που ξέσπασαν στην Βόρεια Αφρική και είπατε πως δεν γνωρίζουμε πώς θα, πού θα καταλήξουν τα πράγματα. Η πολιτική ασφάλειας και κοινή άμυνας δεν μπορούν να, μπορεί να αποτελέσει πανάκια για όλα τα στραβά που συμβαίνουν στον κόσμο. Ωστόσο θα μπορούσε να μας επιτρέψει να γνωρίσουμε καλύτερα αυτέ τις συγκρούσει, να μπορέσουμε να τι προλάβουμε στο μέλλον αλλά και να τις επιλύσουμε. Ε, και για τις συγκρούσει που έχουν ξεσπάσει στην, ε, στην ε, Ανατολική Αφρική αλλά και σε άλλες συγκρούσεις όπως στην υπερνηστερία, στην Γεωργία και αλλού στον Αγκόρνο Κάραμπαχ. Ε, ε, τώρα για την εν λόγω έκθεση είναι πολύ ογκώδης, δεν μπορώ να αναφέρω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά θέλω να μιλήσω για δύο θέματα. Η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τώρα στην Επιτροπή Άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να, ανασύρουμε τα διδάγματα από τα σφάλματα και τις ελλείψεις του παρελθόντος ώστε στο μέλλον να λειτουργήσουμε καλύτερα το θέμα του σχεδιασμού και της διαχείρισης των ευρωπαϊκών ε, επιχειρήσεων. Στείλαμε, μάλλον η ομάδα της Βαϊμάρης έστειλε μια μια πρόταση για την αντιμετώπιση αυτού του, συστη... του, θέματος και επιτά όσον αφορά τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα σε εσά και την... το ΝΑΤΟ και θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις αλλά αντίθετα εξοικονομήσεις. Ε, δεν περιμένουμε επαναστάσεις αλλά σε εξελίξεις και βασιζόμαστε σε εσά. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Ντεκεζέρ για 1,5 λεπτό. Ακούσατε πάρα πολλέ επικρίσει αυτέ τι μέρε. Και εμεί τι καταδικάσαμε. Ε, ήταν πάρα πολύ εμβόλια όλα αυτά, τα οποία ελέγχθησαν. Ε, πολλέ φορέ τα πράγματα δεν είναι ασπρομαύρο να την εξωτερική πολιτική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίση θα πρέπει να έχουμε υπόψη ποιο είναι ο επόμενο στόχο. Ε, γιατί ε, πολλές φορές ε, είσαστε συγκρατημένοι, πολλές φορές έχετε μινιμαλιστικές θέσεις ανακοινώσεις φεύγει μήνυμα πολλές φορές, στέλνετε μήνυμα αλλά πολλές φορές είναι αρνητικό και εσείς κινείστε, τηλεφωνάτε και κάνετε ό,τι μπορείτε αλλά πολλές φορές το αποτέλεσμα των ενεργειών τελικά ε, χάνεται μέσα στο, στο χάος της ε, καθημερινότητας επικαιρότητας οπότε θα πρέπει να δούμε το ότι πολλές φορές η πολιτική εντυπωσιασμό αυτή που ασκούν κάποιοι ηγέτε. Επομένω, επομένως θα πρέπει να δείτε ότι τώρα υπάρχει χώρος για διπλωματία, για πολιτική λόγω της ε, Αραβικής Επανάστασης. Θα πρέπει να διακριτώσει ο ρόλος μας διότι ε, πέραν των ε, ιδιωτικών κάθε χώρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι, ήταν η συμφιλίωση με τη Χαμάση ήταν κάτι το, το απίστευτο και όμως έγινε ε, λόγω της ε, επανάστασης στην Αίγυπτο, λόγω ε, της καταστολής στην Συρία. Και εσείς θα πρέπει τελικά την τελευταία στιγμή να συνομιλήσετε και στο Κατάρ και στο Κάιρο. Επομένως τελικά τι γίνεται με τη Συρία, τι γίνεται με τη Μέση Ανατολή, τι πολιτική ασκείται. Και εγώ σας το είπα ότι αυτό το οποίο κάνετε δεν είναι αρκετό. Συμφωνώ με την αγανάκτηση των Ρημένου Συναδέλφων σε σχέση με την Συριακή εξαίρεση για τον Πασόρα Λάσαντο, ο οποίος επίσης δεν ε, ε, έχει τίποτε κυρώσεις βάρος του και δεν υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Όντως, ε, είχαμε το, το Κουβέιτ, το Νεπάλ, ε, και η Συρία παραλίγο από τις 20 ε, Μαΐου να προεδρεύει το Συμβουλίο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μα το φαντάζεστε κυρία Άστον, ε, οι κυρώσεις είναι ανεπαρκείς. Εσείς τι κάνατε τόσο ώστε να μην αναλάβουν την Προεδρία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον ΟΗΕ, η Συρία; Τι κάνατε για τις σφαγές. Ακόμα και δεν καταφέρετε να τους πείσετε, να τους το πείτε όπως είπε ο κύριος Κομπεντίτ. Μην ε, έχετε τέτοια στάση θολή. Και για την Μέση Ανατολή επίσης εγώ είμαι ευθυγραμμισμένη μαζί σας. Ε, Φαντάχ και αμάς θα πρέπει να συμφιλειωθούν όντως, όμως θα πρέπει να μην επαναλάβουμε τα λάθη του 2007. Όντως η κατάσταση είναι περίπλοκη. Όμως θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία. Η Χαμάς ε, είναι υπέρ της ειρήνευσης και επομένως τα δύο κόμματα του κοινωνικού συνασπισμού κάνανε παραχωρήσεις ε, απίστευτες. Αυτά όλα διατυπώθηκαν ε, εγγράφως και σε ένα μήνα αυτά θα είναι, θα ήταν η κυβέρνηση του συνασπισμός και η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να καταλάβει ότι έχουμε τώρα την ε, διαπραγμάτευση των συνόρων του 2007. Άρα και εσείς να μην λέτε ότι δεν άλλαξε τίποτα και ότι ξαναγυρίζουμε ε, στα γεγονότα που έγιναν δύο, χρόνια πριν. Επομένως, είναι κατεπήγον κυρία είπατε εκπρόσωπος ότι χρειάζεται τόλμη στην εξωτερική πολιτική. Εμείς πάντοτε σας ε, στηρίζουμε εάν έχετε το φάρος και το όραμα. Πρόεδρος, ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Λάμς Ντορφιέ. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Απέχουμε πολύ, Βαρόνια, Άστον, από μια ουσιαστική κυρία εξωτερική πολιτική. Και ακούτε τις σχετικές επικρίσεις. Αλλά νομίζω ότι μερικέ φορέ μετατρέπεστε στον αποδιοπομπαίο τράγο μιας κατάστασης την οποία δεν ελέγχεται στη τελευταία ανάλυση. Διότι δεν έχουν τα κράτη, οι κυβερνήσει στην πολιτική βούληση να συμφωνήσουν σε μια κοινή πολιτική γραμμή. Λιβύα, για παραδείγματι. Πρώτα παρεμποδίζει την ε, ανάληψη δράσεως και κυρώσεων η Ιταλία, μετά αναλαμβάνει μονομερή δράση η Γαλλία, μετά παρεμβαίνει η Γερμανία. Η κατάσταση είναι πολύ συγκεκριμένη. Για τη Συρία, ναι, θα χρειαζόμασταν ε, κυρώσεις, αλλά υπάρχουν κράτη, ακούγεται από τον τύπο ότι πρόκειται για την Ιταλία, την Ελλάδα, ίσως να είναι και η Γερμανία μεταξύ εκείνων που δεν θέλουν να θέσουν τον Χαφεζελάστατ στην ε, λίστα εκείνων των οποίων θα παγώσουν οι λογαριασμοί. Χρειάζεται λοιπόν η βούληση για να προχωρήσουμε στο επόμενο κβαντικό βήμα τη εξωτερική πολιτική. Και αυτό νομίζω μπορεί ο κύριο Τάνοκ να το μεταφέρει στου ε, συντηρητικού φίλου του στη Βρετανία. Αυτό μπορείτε να κάνετε εσεί να αξιοποιήσετε τα κοινοτικά μέσα. Η προαγωγή τη δημοκρατία, η παραδείγματι και με έπλησα ή άκουσα την παρατήρηση σας σχετικά με την επαλήθευση των όρων της δημοκρατίας στην οποία αναφέρατε εσείς γιατί κάνουμε μαζί με την κυρία Ντακεζέρ που είναι η κύρια εισηγήτρια μία έκθεση ακριβώς για το θέμα αυτό για μία δηλαδή ταχεία πολι... μη πολιτικά στιγματισμένη και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική που θα ελέγχει και τους όρους της τήρησης δημοκρατίας. Ευχαριστώ Καμίνσκι. Ένα λεπτό. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, ένα από τα πιο συγκινητικά, μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές στη ζωή μου ήταν το Δεκέμβριο του 2007 όταν με τον πρόεδρο Κατσίνσκι συμμετείχα στη Αγγένεια μάλλον στο άνοιγμα των συνόρων ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία. Εμείς που ζήσαμε πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα είμαστε ε, πραγματικά συγκινηθήκαμε από το άνοιγμα των συνόρων που είναι ένα σύμβολο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε λοιπόν πίσω στα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης. Δεν μπορεί αυτό να αποτελέσει πολιτικό μέσο ε, ή λαϊκιστικό μέσο για να αντιμετωπίσουμε πραγματικά προβλήματα. Η ζώνη του Σέγγεν είναι μια επιτυχία πολύ μεγάλη που πρέπει να την υπερασπιστούμε. Και σας ευχαριστώ για τα λόγια σας. Είπατε ότι η θέση μας απέναντι στην Χαμάς δεν αλλάζει, όμως έχει αλλάξει η θέση του Προέδρου Αμπάς και των Παλαιστινίων απέναντι στην Χαμάς. Θα ήθελα να ρωτήσω, η βοήθεια που στέλνουμε στην αυτόνομη Παλαιστινιακή Αρχή χρησιμοποιούνται από αυτούς τους ε, εχθρούς απέναντι στη μοναδική δημοκρατία της περιοχής, δηλαδή εναντίον του Ισραήλ που είναι η μόνη χώρα στην Μέση Ανατολή όπου οι Άραβες μπορούν να ελέγξουν τους δικούς τους εκπροσώπους στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπραντνερ για δύο λεπτά. Η κυρία Μπνάντρα, με συγχωρείτε. Καλώς ήρθατε, κυρία είπατε εκπρόσωπε. Η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινοτική μέθοδο, μια εξωτερική πολιτική. Και τώρα που έχει περισσότερες, ε, περισσότερα μέσα στη διάθεση ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να περιμένουν τα κράτη-μέλη να διαμορφώσουν τα ίδια μια κατάσταση και μετά να διαμορφώσουν ένα κοινό παρονομαστή ε, ελάχιστο για να παρεμποδίσουν ουσιαστικά την ανάληψη δράση. Όπω η παραδείγματι στην ε, Συρία, θα έπρεπε να δούμε τι δικέ σα απόψει. Μην μα λέτε τι λένε τα κράτη-μέλη. Πείτε μα εσεί τι θέλετε. Θέλετε κυρώσει νέου. Μα λέτε να ε, ασκήσουμε πιέσει στα κράτη-μέλη. Τότε, ναι, καταδείξτε μα ποια κράτη χρειάζεται, σε ποια κράτη πρέπει να ασκήσουμε πιέσει. Ξεκινήστε τον ανοιχτό διάλογο. Ναι, ξέρουμε ότι μερικέ φορέ χρειάζεται να ομολογήσουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να αναλάβουν αποφασιστική δράση ή δεν θέλουν να σα δουν ισχυροί επιβεβαιώνω όμω, κυρία Άστον, δεν πρόκειται ούτε να σα στηρίξουν ούτε να σα σώσουν τη ζωή την ώρα που θα χρειαστείτε βοήθεια. Δεν θα σα εγγυηθούν την παραμονή στη θέση σα. Ε, και σα διαβεβαιώ ότι και η συνθήκη τη Λισαβόνα έχει προβλέψει πολύ ισχυρότερο ρόλο για εσά. Γιατί εσεί ουσιαστικά αντικαθιστάτε την ε, εναλλασσόμενη Προεδρία, είστε Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή. Εσεί μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα, την λεγόμενη ατζέντα, μπορείτε να προβάλλετε τι θέσει σα και τι αποφάσει σα και να ε, αφήσετε εκ των υστέρων να αντιδράσουν τα κράτη-μέλη. Και, εν περιπτώσει, αν δεν θέλετε να ορίσετε τι δικέ σα θέσει, αφήστε του άλλου να ε, προχωρήσουν στην αναθεώρηση του προγράμματος Gothenburg που ξεκίνησε από την Άννα και που τώρα ξεκίνησε να αναθεωρεί η Ουγγρική Προεδρία με σκοπό να σας το αναθέσει σε εσάς. Εσείς όμως το ε, παρεμποδίσατε αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πρέπει να τολμήσετε περισσότερο, να αναθέτετε περισσότερες αρμοδιότητες να αποτελέσετε εσείς τον παράγοντα της αλλογής που χρειαζόμαστε. Μόνο αυτό και μόνο αυτό σας υπόσχομαι πρόκειται να οδηγήσει σε αλλαγή στάσης και νοοτροπιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Χατζηγεωργίου για 1,5 λεπτό. Κυρία Άστον, εγώ νομίζω ότι έχετε δίκιο να αισθάνεστε αδικημένοι από την κριτική που σας ασκείτε τι φταίτε εσεί όταν είναι φανερό ότι είστε δέσμια των αποφάσεων των μεγάλων κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω έχω ακόμα ένα ερώτημα. Όσοι κριτικάρουν εδώ τι κυβερνήσει του, θα κάνουν μήπω κάτι διαφορετικό από αυτό που καταγγέλνουν όταν αύριο θα είναι κυβερνήσει στι χώρε του. Εγώ συμφωνώ και με αυτό που είπε ο κύριο Σούλτ, ότι μέχρι χτε ευρωπαϊκά κράτη πουλούσαν όπλα σε αυτού που ανακαλύψαμε σήμερα ότι είναι δικτάτορε. Όμω πολιτική σημαίνει πρόβλεψη, σημαίνει έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων. Αλλιώτικα απλώ κάνουμε νεκροψία. Ευρωπαϊκά κράτη βομβαρδίζουν του χτεσινού εταίρου του, την ίδια ώρα όμω βομβαρδίζουν και καταστρέφουν τα όπλα που ήδη πούλησαν. Προφανώ δεν μπορεί να πουλήσει καινούρια όπλα αν δεν βομβαρδίσει τα παλιά. Για μα, για να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει μια πολιτική βασισμένη σε ειρηνικέ αρχέ απεγκλωβισμένη από στρατιωτικά μέσα και παρεμβάσεις και να προωθήσει την αποστρατιωκοποίηση των διεθνών σχέσεων να απελευθερωθεί η ίδια από τα πυρηνικά όπλα και να συμβάλει στην αποπυρηνικοποίηση του πλανήτη. αυτό θα είναι μια θέση στιγμής μια δόξα στιγμής για την ευρωπαϊκή ένωση. μια φράση για τη μια γείτονα χώρα της μέσης ανατολής την τουρκία. στη χώρα αυτή βρίσκονται στη φυλακή σήμερα δεκάδες δημοσιογράφοι και συνεχίζει να κατέχει με 40.000 στρατό την μισή Κύπρο και παραβιάζει τα δικαιώματα τουρκοκυπρίων και ελληνοκυπρίων. Εδώ είναι που καλώ την κυρία Άστον να δει έγκαιρα στην Κύπρο αυτό που δεν είδαμε αργά στην Αραβική Χερσόνησο. Προβέρα για ένα λεπτό τώρα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είπα ότι εκπρόσωπε Άστον. Οι επιθέσεις της Εκκλησίας Κοπτών στην Αίγυπτο και οι δολοφονίες πιστών δείχνουν μια επιδείνωση της θρησκευτικής δυσανοχής ε, και που προδίδει το πνεύμα της ε, πλατείας ε, Ταρέκο που κόπτες και μουσουλμάνοι επαναστάτησαν. Αυτό καθιστά δύνατη την κοινωνική σταθερότητα που είναι απαραίτητη για μια ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη δέσμευση από τις αρχές του Καΐρου για την προστασία των μειονοτήτων και κατά των ακροτήτων των των ε, σαλαφτών και να ε, ε, είναι απαραίτητη η οικονομική ανάπτυξη, εξωτερικέ επενδύσει μάλλον από το εξωτερικό και σίγουρα ο τουρισμό, Αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν χωρί την ανοχή, την τάξη και την ασφάλεια. Σημαντικό να δώσει γενναιόδορες γενναιόδορη βοήθεια η Ευρώπη, αλλά αυτό θα πρέπει να καθορίζεται από μια αποτελεσματική πολιτική προστασία των μειονοτήτων σύμφωνα με την αρχή more for more που εσεί είπατε εκπρόσωποι προτείνετε μετά από τον, μαζί με τον Επίτροπο Φίλε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Μόλτζερ για δύο λεπτά. Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε. Βλέπουμε με παράδειγμα τη Συρία σε τι προβλήματα έχει λεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε ότι ο Ασάτ, ο δικτάτορας, συνεχίζει να βομβαρδίζει το λαό του και να ε, καταστέλει βία τις διαδηλώσεις. Χρειάζονται λοιπόν σαφείς κυρώσεις. Η δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα για τον ανθρώπινο κόσμο, από ό,τι φαίνεται, δεν σημαίνουν τίποτα άλλο παρά κενά λόγια. Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες, δίνει προτεραιότητα στα γεωπολιτικά συμφέροντα των Αμερικανών όταν αναλαμβάνει δράση στην, στην περιοχή αυτή. Η κοινή ανάπτυξη του κοινού χώρου της Νότιας Μεσογείου μάλλον έχει πληγεί από τις εξελίξεις αυτές και ενώ έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το χάος στην Τινησία μια κυβέρνηση που διαθέχτηκε την άλλη φαίνεται ότι ετοιμάζεται να πέσει. Βλέπουμε τις εξελίξεις ε, στην Αίγυπτο να μετατρέπουν την κυβέρνηση σε μια στρατιωτική δικτατορία όπου κινδυνεύουν η ζωή ίδια των χριστιανών ε, κοπτών και μια πολύ χλιαρή αντίδραση από τις διεθνείς ε, δυνάμεις. Για δε τη Συρία, ο Άσαντ ξέρει ότι μπορεί να στηρίσει στην ε, ε, υποστήριξη του στρατού του και ίσως εκεί μπορούμε να προβλέψουμε ένα πολύ μεγάλο κύμα μεταναστών γιατί ήδη είναι πολλές εκατοντάδες ε, πολιτών της Συρίας που έχουν διαφύγει μέσω των σύνορων της Τουρκίας στο εξωτερικό. Η κατάσταση λοιπόν αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη δεν είναι τόσο μακριά από την Μέση Ανατολή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες και δεν μπορούμε να αφήσουμε ε, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να μας εμπλέξουν σε ένα κικαιώνα βίας και τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. Κουκάν. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Άστον, αγαπητοί συνάδελφοι. Όσον αφορά την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην διεθνή σκηνή, οι εξελίξει έχουν καταδείξει ότι θα πρέπει ταχύτερα να ενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τι παγκόσμιε προκλήσει. Η συνθήκη τη Λισαβόνα μα έχει δώσει το πλαίσιο και τα μέσα ούτως ώστε να αναλάβουμε τέτοιου είδου ενέργειες. Επομένως ε, έτσι θα πρέπει να αρχίσουμε να αναέρουμε κάποια κενά που έχει η διεθνής τάξη παρά την συνάντηση της Κοπενχάγης έχουμε ε, το, το ψήφισμα της, ε, του του ΟΗΕ μας επιτρέπει τώρα να εμπλακούμε πλήρως συγχαρητήρια κυρία Άστον και επομένως θα, θα πρέπει να μπορέσουμε να χαράξουμε μια κοινή στρατηγική ε, έχουμε αυτή την έκθεση που λέει το πού θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπαθειές μας και πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα. Το, το πώς δηλαδή θα έχουμε καλύτερο συντονισμό ε, στο σύστημα του ΟΗΕ. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τους διεθνείς οικονομικούς ε, οργανισμούς, τις πολυμε τους πολυμερείς οργανισμούς, όλα αυτά βεβαίως απαιτούν χρόνο και απαιτούν συνεπεί ενέργειες και συντονισμένες από πλευρά μας. Επομένως χρειάζεται μια μακρόπνοη στρατηγική. Αυτή να έχει ξεκάθαρα στάδια, ε, να γίνεται ό,τι πρέπει, ούτω ώστε να μπορέσουμε να δρεώσουμε την παρουσία μας στη παγκόσμια σκηνή και ελπίζω ότι μια τέτοια στρατηγική ε, θα, θα την διαμορφώσετε ταχαίως κυρία Άστον και επίσης θα μας δοθεί ευκαιρία να τη ζητήσουμε σε αυτό το ημικύκλιο την εκκλησία ε, Αλμπερτίνη έχω να πω ότι στην Αλβανία ε, είχε εκλογές και εγώ είχα πάει εκεί στις εκλογές ε, ως αποστολή παρατηρητών και το μήνυμα είναι το εξής η Αλβανία και δεν μιλάω για τους πολιτικούς μιλάω για τον Κοσμάκη αυτοί σε εμά προσβλέπουν με εμπιστοσύνη, με ελπίδα, με προσδοκία για να τους βοηθήσουμε να εξεύρουν λύσεις σε αυτό το πολιτικό αδιέξοδο. Ε, που τους οδήγησαν η πολιτική τους. Επομένως, ε, ένα μικρό βήμα που κάναμε νομίζω ότι οδήγησε σε αυτή την επιτυχία. Ε, δίνουμε εξετάσεις σε αυτά εκεί και επομένως θα πρέπει με αξιοπρέπεια να ανταποκριθούμε. Ο ευχαριστούμε πολύ και τώρα το λόγο κύριε για τρία λεπτά, τρεις λεπτά. Πρόεδρε, κύριε Άστον, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Αλμπερτίνη για τη συνεργασία στην έκθεση του εγώ Σκιώδης της. Ήταν πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και προφανώς χάρη με την ευκαιρία αυτή τη έκθεση, αλλά και χάρη στη συζήτηση που έχουμε σήμερα στρέψαμε το βλέμμα προς τη Μέση Ανατολή, προς τον Νότο και θα ήθελα να επανέλθω, όπω και η κυρία Ντεκεζέρ, για άλλη μια φορά στην κατάσταση στην Παλαιστίνη. Διότι διαβλέπω μεγάλη ευκαιρία στη συμφωνία μεταξύ Χάμά και Φατάχ και την ευκαιρία ακόμη για ίδρυση ενό κράτου. Εάν ιδρυθεί λοιπόν το κράτο, με την ίδρυση ενό κράτου, συνδέονται και ευθύνε. Αυτό πρέπει να το καταστήσουμε σαφέ. Η ευθύνη είναι τι αναγνώριση του Ισραήλ, εγκατάλειψη της βίας αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να αναγνωρίσει και το Ισραήλ το νέο αυτό κράτος. Όπως θα πρέπει Χαμάς να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Μόνο τότε μπορούμε να έχουμε μια λύση δύο κρατών, δηλαδή ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και δεν θέλω να μιλήσω μόνο με το βλέμμα προς τον Νότο, αλλά και προς Ανατολάς καθώς είχα την ευκαιρία να ηγηθώ μια αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου του Τουρκμενιστάν ε, και ανέλαβα εχθές και μια εισήγηση για τη σχέση μας με τη Ρωσία. Θα ήθελα να πω ότι επικεντρωνόμενοι στα προβλήματά μα, ε, τα προβλήματα στα νότια μα σύνορα δεν πρέπει να λησμονούμε την ανατολική μα γειτονία. Και εδώ έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει η Τουρκία. Δεν μπορούμε την Τουρκία να την εξετάσουμε μόνο με την προοπτική τη ε, προσχώρηση και το ναι ή όχι στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είναι εταίρο και βέβαια στι σχέσει μα στη Μέση Ανατολή αλλά και στι σχέσει μα με τα κράτη τη Μαύρη Θάλασσα, του Εύξηνου Πόντου. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε μέσα σε μια ευρύτερη εξωτερική πολιτική ε, και πολιτική ασφάλεια Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό χωρί να έχει δηλαδή άμεσα σχέση και διασύνδεση με την προοπτική τη Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ρωσία δεν θέλω να πω ότι θέλουμε εταιρική σχέση με τη Ρωσία, αλλά αυτό το, διαπραγματευόμαστε από θέση ισχύω και με αυτοπεποίθηση. Μερικές φορές βλέπουμε ότι ε, μπορεί η Ρωσία να κάνει πολλά και εμείς να κάνουμε λιγότερα. Λοιπόν, θα πρέπει μια σχέση εταιρική να είναι πραγματικά σχέση ισότιμη, να προσφέρουν και οι δύο το ίδιο. Και θα ήθελα να ε, εκφράσω την έκπληξή μου ως προς το, τις εξελίξεις των πιέσεων που ασκεί η Ρωσία στην Ουκρανία παραδείγματι. Τον τελευταίο καιρό ασκεί πολλές και ισχυρές πιέσεις εις βάρος της Ουκρανίας, πράγμα το οποίο δεν θεωρούμε δίκαιο. Το ίδιο βλέπουμε και εν μέρη σε σχέση με το Τουρκμενιστάν. Θέλουμε λοιπόν να απευθύνουμε το μήνυμα ότι ναι, θέλουμε μια εταιρική σχέση, θέλουμε μια ισότιμη ε, σχέση, θέλουμε να αναπτύξουμε προστερέ σχέσεις, αλλά οι συνθήκες θα πρέπει να είναι σωστές. Για δε τις ε, υπόλοιπες χώρες ε, της ε, περιοχής αυτής της Κεντρικής Ασίας θέλουμε να αναλάβουμε δράση, θέλουμε να έχουμε εταιρικέ σχέσεις, αλλά δεν έχουμε αντιπροσωπείες, δεν έχουμε χρήματα για να στήσουμε αντιπροσωπείες. Θέλουμε την ενέργειά τους, θέλουμε να αναπτύξουμε τις εμπορικές σχέσεις, θέλουμε να προαγάγουμε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στην πράξη. Πρόκειται για κράτη τη Κεντρική Ασία, τα οποία είναι ουσιαστικά οι γείτονέ μα. Ή θα στραφούν προ την Κίνα, ή θα στραφούν προ τη Ρωσία, ή, εάν του δώσουμε την ευκαιρία, θα αναπτύξουν τι σχέσει του με την Ευρώπη. Και επειδή έχουμε πει ξεκάθαρο ότι θέλουμε να τα υποστηρίξουμε και είναι απόλυτα σωστό, πιστεύω, ε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να το πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα, λίγο πιο απερίφραστα και λίγο πιο ουσιαστικά για να βοηθήσουμε την Ευρώπη αλλά και τα κράτη αυτά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριο Νταφ για ένα μισή λεπτό. Καθιάστον. Μίλησες ξεκάθαρα όσον αφορά το πρόβλημα του να αποσπά κανείς συμφωνίες από 27 υπουργού εξωτερικών. Η συνθήκη της Λισαβόνα. δίνει την ευχαίρεια προ κάτι τέτοιο. Συμφωνία και δημιουργία των προποθέσεων για ενισχυμένη συνεργασία. Η ομοφωνία αφορά αυτές τις κυρώσεις κατά της Συρίας ε, όμως θα πρέπει να καταργηθεί και αυτό το οποίο έχω να προτείνω είναι να αναζητηθεί η πρωτοπορία να υπάρχει έτσι ένας σκληρός πυρήνα των ε, όσων έχουν την πολιτική βούληση των όσων κρατών την πολιτική βούληση και να συνεργαστείς μαζί τους, ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια τέτοια κοινή πολιτική. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φανόρντεν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βαρονιάστον δεν θα σας εκπλήξω εάν ε, σας εκφράσω την απογοήτευσή μου. Όχι όσον αφορά τα όσα έχετε πετύχει με την ε, κοινή σας πολιτική αλλά και το ότι ακόμα επιμένετε ε, να, ε, να, να, να, να σπαταλάτε τις προσπάθειές σας σε κάτι το οποίο δεν πιάνει τόπο. Έχουμε αυτές όλες τις περίφημες αποστολές. Αυτές οι αποστολές δεν σημαίνουν τίποτα. Καλύτερα να τις έκανε το ΝΑΤΟ. Πρόκειται για πολιτικές αποστολές ή πρόκειται τέλο πάντων για κάποιες μη επιχειρησιακές προσπάθειες στρατιωτικών και ουσιαστικά σε αυτές τις ε, αποστολές ε, γονατιστεί παρακαλά ενώ πετύχει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αποσπαστεί μια εντολή ούτως ώστε να ισχύσει το θαλάσσιο εμπάργο, ο θαλάσσιος αποκλεισμός και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας. Το θέμα είναι πάντως ότι ούτε ο ΙΕ ούτε το ΝΑΤΟ θεωρούν ότι εμείς πρέπει να εμπλακούμε στα δίκαιο. Φυσικά και χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια και θα μπορούσε βεβαίω να είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω όχι με ε, τρόπο που να εκφράζει κάποιες τέτοιες άστοχες στρατιωτικές φιλοδοξίες. Αυτό διαιρεί του συμμάχους. Έχουμε επικάλυψη ενεργειών και έτσι και υπονομεύουμε άλλωστε και τον ρόλο του ΝΑΤΟ, το εκθέτουμε στους ίδιους τους συμμάχους. Πρόεδρος. Βλέπω μια μπλε κάρτα υψωμένη. Δέχεστε. Ε, επερώτηση. Κυρία Σινκλέρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα συμφωνούσε ο συνάδελφος. Κατ' όμως είπε για τον ΟΗΕ ότι εάν είχαμε ένα βήμα έκφρασης για το ότι θα είχαμε επομένω ε, μεταφορά της ε, εθνικής κυριαρχίας από Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο προς τον ε, ΟΗΕ. Θα σας ευχαριστώ για την ερώτηση του κ. Φανόρντεν. Ναι, και αυτό αποτελεί ακόμα μια τραγική συνέπεια στην κρίση της Λισαβόνας. Ότι δηλαδή η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εκχωρήσουν την ε, θέση τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στη θέση τους να συμμετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι αυτό θέλει να το κάνει καμία χώρα. Αυτό όμως το διατυπώνει η Συνήθεια Λισαβόνας και γι' αυτό και εμείς αντιτιθέμενο. Δύο λεπτά κύριε Λούνατσεκ. Η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει Άστον, υπάτη εκπρόσωπο. Πάρα πολύ θετικά όλα όσα είπατε στην πρώτη σας εισήγηση όσον αφορά ε, την πολιτική τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι γίνεται με την Βόρεια Αφρική, την Ισία, Λιβύη και ε, ιδίως όσα μας είπατε για του νέου και όσα είπατε για τις ε, γυναίκε. Συμφωνούμε για την δική σα προσέγγιση, για την ε, βαθιά δημοκρατία και είναι πράγματα τα οποία φαντάζομαι βρίσκουν τους πάντες εδώ συμφώνου και επομένω πιστεύουμε θα τα καταφέρετε. Όμω από την άλλη μεριά πρέπει να συμφωνήσουμε με του περισσότερου συναδέλφου ότι δηλαδή ο Ασάντ θα έπρεπε και αυτό να έχει υποστεί κάποιε κυρώσει και όπω είπε ο Ντανιέλ Κομπεντίτ, πέστε μα, ποιοι ε, έφεραν την εμπλοκή στο Συμβούλιο, ο κύριο Βέστελφελτ ή ποιο άλλο. Οπότε ε, θα... παρακαλώ να έχετε διαφάνεια στι σχέσει μαζί μα και τότε εμεί θα σα στηρίξουμε αυτό και για την ε, εντολή σα. Όσο πιο πολλά μα πείτε για το γίνεται το Συμβούλιο, τόσο πιο πολύ θα σα ε, στηρίξουμε. Παρακαλώ, πέστε μα. Και όπω είπατε και εσεί, ε, αυτό θα σημαίνει συνέπεια και συνοχή. Στην έκθεση Αλμπερτίνη που αυτή τη εβδομάδα θα ψηφίσουμε, ζητούμε οι εθνικέ πολιτικέ να στηρίζουν τι θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσον αφορά τους αδέλφου εδώ, στο Κοινοβούλιο, παρακαλώ, όσοι προέρχεστε από κόμματα εξουσίας να τα πείτε αυτά στους υπουργού εξωτερικών και στους πρωθυπουργούς να στηρίξουν την κοινή εξωτερική πολιτική. Μην φροντίζετε μόνο τα του οίκου σας όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Αλλιώ δεν θα αποκτήσουμε ποτέ μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Ε, Επομένω, να δείξετε φιλοσοφία, να είσαστε κυρία στον τολμηρή τη φιλοδοξία σα, διότι μιλούμε για 61 χρόνια μετά την ε, διακήρυξη Σούμα, την οποία και τιμήσαμε την Δευτέρα, διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ συγκεκριμένα χρειάζεται αποτροπή κρίσεων, τη κρίση ε, και διαχείρισή του. Επομένω, ε, θέλουμε αυτή την εξωτερική υπηρεσία για να υπάρξει μια ανεξάρτητη μελέτη επιπτώσεων όσον αφορά ε, τα κοινωνικά, όσον αφορά τι συνέπειε τέτοιων αποστολών και χρειάζεται περισσότερο προσωπικό επίσης σε αυτές τις ε, αποστολές. Πρόεδρος. Επερώτηση. Μπλε κάρτα βλέπω. Δέχεστε, ναι. Κύριε Συγκλέρα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σωστά αυτά τα οποία είπατε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, αυτό που είπατε για την κοινή πολιτική, αλλά συμφωνείτε ότι είναι φαρισαϊκά αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την θανατική ποινή. Γιατί έχουμε αυτή την κοινή δήλωση. Μπαρόσο και φουνερόν πάει. Όσον αφορά το θάνατο του Μπιν Λάντεν. Τι γίνεται η θανατική ποινή αποτελεί κύρωση Αυτό το οποίο μας είπατε για τον θάνατο του Μπιν Λάντεν, όχι δεν ήταν κανένα του θανατική καταδίκη. Ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να συλληφθεί και να συρθεί στη δικαιοσύνη. Όχι, δεν είναι ε, υποκριτικό αυτό που είπε ο κύριος Μπαρόσο. Πρόεδρε μια δήλωση κύριος Φανουροπέ. Και εγώ θα προτιμούσα να έχει δικαστεί από κάποιο διεθνές δικαστήριο ο Μπιν Λάντεν. Δεν έγινε αυτό. Όμως μην τους κατηγορείτε για υποκρισία γιατί τη χρειαζόμασταν αυτή την κοινή θέση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Λιγαρίκα για 1,5 λεπτό. Κυρία, είπατε εκπρόσωπε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ πως τα όσα είπατε στην πρώτη σας παρέμβαση όσον αφορά την επιθυμία σας για ύπαρξη Παλαιστινιακού κράτους μετά από την ε, Παλαιστινιακή Συμφιλίωση είναι πάρα σημαντικά. Αυτή η Παλαιστινιακή συνεννόηση, η συμφιλίωση είναι πολύ σημαντική και όπως είπατε το μάλλον αντίθετα με το αυτό που είπατε, για ΑΜΑΣ για πρώτη φορά δέχτηκε την ε, την ε, ΟΑΠ και την ΦΑΤΑΧ για ως υπαρκτούς εταίρους και συνομιλητές. Ε, γι' αυτό και, μάλιστα θα δημιουργηθεί μια κατάλληλη ομάδα για την προετοιμασία εκλογών. Ε, έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως ανεξάρτητου κράτους με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα με τα σύνορα του 67 στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον επόμενο Σεπτέμβριο. Πέρα από αυτά, είπατε πριν από λίγο, κυρία, είπατε εκπρόσωπε, ποιο νέα πράξη θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γνωρίσει το Παλαιστινικό κράτος και να υπερασπιστεί αυτή την ιδέα στον ΟΗΕ. Ε, επιπλέον μπορείτε να μας ε, γνωστοποιήσετε τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς η ίδια ώστε η Ισραηλινή κυβέρνηση να αποκαταστήσει, μάλλον να επιστρέψει τα, τους φόρους και τους δασμούς που θα πρέπει να που ανήκουν στο Παλαιστινιακό κράτος. Ευχαριστώ. Ε, do you accept... Δέχεστε περώτηση, μπλε <coughs> Yes. Yes, please. Παρακαλώ. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι. Συμφωνώ. Η συμφωνία μεταξύ Φατάχ και Χαμάς αποτελεί ένα ιστορικό βήμα στη διαδικασία της συμφωνίωση μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραήλ και μόνο βήματα πρόοδου μπορούν να πραγματοποιηθούν από εδώ και μπρος. Όπως είπε όμως η κυρία Άστον αυτή η δεύτερη αποστολή βοήθειας ε, προξενεί μάλλον ζημιά. Δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα θετικό. Εσείς συμφωνείτε στην καταδίκη αυτής της δεύτερης αποστολής πλοίων. Euh, Όχι, κοιτάξτε, αυτά τα πλοία είναι πρωτοβουλία ε, της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης για να προξενήσουν άρση ενός οικονομικού αποκλεισμού, ενός αποκλεισμού περιτού και άχρηστου. Μόνο εάν, εμείς, ε, μόνο εάν τα κράτη είχαν ε, μπορέσει να επιβάλλουν το διεθνές δίκαιο όπως όφυλαν, δεν θα χρειαζόταν να παρέμβουμε εμείς. Γιατί έχουν μείνει αποκλεισμένοι οι Παλαιστίνοι για πάρα πολύ καιρό. Το λόγο έχει ο κύριος Σολαβράκος, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, συγχαίρω τον κύριο αλμπερτίνη για την έκθεσή του και την αναφορά που κάνει στις αρχές και τις προτεραιότητες της ε, κέπα της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. βεβαίως ο κόσμος αλλάζει και η ευρωπαϊκή ένωση καλείται να αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις που είναι απαραίτητο να λάβει δράσεις ουσιαστικές για την αντιμετώπιση τους. απειλές από τη συνεχιζόμενη φτώχεια τον κοινωνικό αποκλεισμό ευρέων μαζών τη διόγκωση της ενεργείας τις γεωπολιτικές μεταβολές στον αραβικό κόσμο σημειώστε το ιδιαίτερα αυτό τις φυσικές καταστροφές και τη μετανάστευση αποτελούν βασικό πρόβλημα του παρόντος και προεικονίζουν εντάξει το μέλλον. ειδικότερα το θέμα της μετανάστευσης που αποτελεί σημείο τριβής πρόσφατα μεταξύ ιταλίας και γαλλίας έθεσε σε αμφισβήτηση τη συνθήκη κατά την άποψή μου το μεταναστευτικό πρόβλημα δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε πρέπει όμως να το διαχειριστούμε με συνέση και αποφασιστικότητα ναι στην αλληλεγγύη αλλά ναι και στη διατήρηση των κοινωνικών δομών και οποιαδήποτε συζήτηση για τη συνθήκη σέγγεν κατά την άποψή μου πρέπει να συνδυαστεί με τροποποίηση της συνθήκης δουβλίνο 2. ευχαριστώ πάρα πολύ. E Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Σίνκλερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέδη Άστον, εγώ ε, θα πω κάποια πράγματα συμπάθεια και στήριξης προ εσά. Παρακολουθούσα ένα πρόγραμμα του BBC το οποίο συζητούσε ο Τζέρεμι Πάξμαν και εσεί βρεθήκατε σε πολύ δύσκολη θέση. Σας ρώτησε από ποιον παίρνετε τις διαταγές σας. Ποια από τις, ποιο από τις 27 χώρε είναι αυτή με την οποία συνομιλείτε. Δεν, και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει μία κοινή πολιτική. Το είδαμε αυτό με το ψήφισμα του ΟΗΕ για την ε, ε, ε η απαγόρηση πτήσεων στη Λιβύη. Ε, πώς μπορούμε να έχουμε κοινή πολιτική όταν μία από τις μεγαλύτερες ε, χώρες της Ένωσης είναι αντίθετη με δύο άλλες ε, μεγάλες χώρες της Ένωσης. Έχετε πραγματικά πολύ δύσκολη αποστολή. Εγώ λοιπόν σας υποστήριξα και διάβασα στην Κυριακάτικη εφημερίδα ότι δεν θα εγκαταλείψετε τη θέση σας. Είναι πολύ σημαντική η θέση σας για την ευρωπαϊκή πολιτική και είναι πολύ σημαντικό επίσης ε, να μείνετε όσο γίνεται περισσότερο στη θέση σας και για τη χώρα μας, γιατί ε, Όσο είσαστε εσεί σε αυτή τη θέση, δεν θα έχουμε πρόβλημα να χάσουμε την κυριαρχία μα. Εμεί, μιλώ για τη χώρα μου βέβαια. Τώρα, εσείς μιλήσατε για παίρνετε ένα σωρό χρήματα στην θέση σας και έχετε πει επανειλημμένως πως αυτό ήταν ε, ένα πολύ μικρή, μια πολύ μικρή υπόθεση ότι δεν υπήρχε σημαντική μεταφορά και, ε, κυριαρχίας. Το είπατε επανειλημμένως, ήταν ανοιχτές ερωτήσεις. Μπορούμε να έχουμε μια ειλικρινή απάντηση από πλευρά σας. Το λόγο έχει ο κύριος Σαλαφράγκα για δύο λεπτά. Κυρία Αντιπρόεδρε, κύριε Υπάρχει εκπρόσωπε, συνάδελφοι, το βασικό σημείο της κουβέντας είναι το κατά πόσον θα πρέπει να προστατευτούμε προς την πολιτική που θα ασκήσουμε για την Βόρεια Αφρική, τη Μέση τα είπε η κυρία Άστον. Θα πρέπει να μην υπάρχουν σκιά στις σχέσεις μας ο Τζόζιο Ναπολιτάνο μας τα επενθύμησε αυτά, ο πρώην συνάδελφο. Παρά τι προσπαθίε σα, κύριε Άστον, έχουμε κάποιε ε, σκιέ και επομένω θα έπρεπε να έχουμε πιο ξεκάθαρα κριτήρια για το τι θα κάνουμε στο Συμβούλιο ασφαλεία. και στο Συμβούλιο επίση. Τι γίνεται επίση και με το στρατόπεδο Ασράφ. Πιστέψτε με ξέρω πόσο σημαντικά είναι αυτά τα οποία κάνετε, αλλά παρά τα όσα γίνονται στι ανθρωπιστικές σα προσπάθειες, ο Γενικό Διευθυντής σα, το Ιδρυογραφείο σας, ε, έχουμε αυτή την δήλωση. Έχουμε αυτό το σχέδιο το οποίο και εγώ εξέγησα και είχαμε όμως 30 τόσους ε, νεκρούς και 300 τραυματίες στο τόπο αυτό, το είπαμε ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε και θα πρέπει να έχουμε κάποια συνέπεια και συνοχή στα όσα κάνουμε όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία τους και θα πρέπει να αναβάρουμε τους, τους κινδύνους όταν πρέπει να σώσουμε ζωές. Έχουμε τον διαφωνούντα στην Κούβα, τον Σωτογκαρθία, ο οποίος ε, συνελήφθη, ξυλοκοπήθηκε και τελικά πέθανε. Θα πρέπει να ζητηθεί έρευνα που να διαφωτίσει τα όσα παράδεκτα αποτρόπια γίνανε και θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει αιτιώδη σχέση μεταξύ ξυλοκοπήματος και θανάτου Για να προβείται στη συνέχεια στην καταδίκη του εγκλήματος. Ο κύριος Βιτζενίνη για δύο λεπτά. Πρόεδρε, κυρία παρακολούθησα μεγάλη ικανοποίηση της δηλώσεις. Συμφωνώ με κάθε λέξη τις ομιλίες σας παρά τις επικρίσεις που ακούστηκαν από μέρος της, ε, του Κοινοβουλίου και βέβαια και από την κοινή γνώμη για τη δυνατότητα να μιλάμε με μία φωνή ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική σας φωνή είναι σαφής. Όμως, ωστόσο επιτυχία μπορούμε να έχουμε μόνο εάν και οι άλλοι συμφωνήσουν σε μία φωνή και τα κράτη. Γιατί τώρα βλέπουμε ότι ακούγονται διαφορετικές και φάλτσες φωνές προς κάθε κατεύθυνση. Σας διαβεβαίω, κυρία Επατή εκπρόσωπε, ότι το Κοινοβούλιο είναι ο φυσικός σας σύμμαχος και χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας. Γι' αυτό σας συνιστώ να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τη δική μας υποστηρίξη αλλά και ε, με την ευκαιρία της νέας έκθεσης του, για την ε, ΕΠΑ να αναλάβετε την πρωτοβουλία για να συγυρίσετε αυτές τις σχέσεις τις εξωτερικές χωρίς βραδιπορία. Είναι ξεκάθαρο ότι η Αίγυπτος και η Τινησία θα χρειαστούν βοήθεια σε δύο φάσεις. Στην πρώτη αυτή φάση χρειάζονται άμεση βοήθεια και στήριξη. Υπάρχει ανάγκη στα αραβικά κράτη εν γέννη για δημοκρατία και ελευθερίες, αλλά και μακροπρόθεσμα κοινωνικές προοπτικές. Εμείς, οι σοσιαλιστές, οι σοσιαλδημοκράτες Ευρώπης, έχουμε κάνει μια μεγάλη συνεδρίαση όπου καλέσαμε την Ευρώπη να τακτοποιήσει τα του οίκο της και να εκφράσει μια απερίφραστη υποστήριξη προ τι δημοκρατικέ δυνάμει στι περιοχέ αυτέ. Την προηγούμενη εβδομάδα θεσπίστηκε γύρω στην κοινοβουλευτική συνέλευση που αποτελεί μια σαφή ένδειξη της βούλησής μας για δημοκρατικό διάλογο με τους εταίρους μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Νέιτσε ο Ιτεμπρούκ για 1,5 λεπτό. Κυρία, είπατε εκπρόσωπε, κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι. Τα λόγια είναι εργαλεία, τα λόγια είναι μέσα και τα λόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως όπλα στην εξωτερική πολιτική και γι' αυτό θα πρέπει με φιδό να τα χρησιμοποιούμε και με σύνεση. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να χρησιμοποιηθούν με αποφασιστικότητα. Κυρία, είπατε εκπρόσωποι, πραγματικά η φωνή σας δεν ακούστηκε τα τις πρώτες μέρες ε, της ε, των φρικαλαιοτήτων που, στις οποίες πρέβησαν οι Συριακές Αρχές και πιστεύω ότι θαραλέοι οι πολίτες που διαδήλωσαν και εξακολουθούν να διαδηλώνουν στη Συρία θέτοντα τη ζωή τους σε κίνδυνο αισθάνθηκαν ακόμη περισσότερο αυτή την έλλειψη από την, την ανυπαρξία σας. Ε, υπάρχουν στιγμέ όπου πρέπει κανείς να υψώσει τη φωνή του άμεσα και αυτή ήταν μια από αυτέ τι στιγμέ. Α στραφώ τώρα στην Μέση Ανατολή. Πιστεύω πως ε, η παρακράτηση φόρων ε, που συλλέγονται στην Παλαιστίνη από την Ισραηλινή κυβέρνηση είναι πραγματικά πολύ ατυχή ενέργεια και επιπλέον ε, δεν είναι και συνεπής, καταρχήν, καταρχήν να ζητά ότι τα θα πρέπει να λυθεί το θέμα της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας και τα λοιπά και όταν έχει βρεθεί η συμφωνία να λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση που είναι τόσο κοινική. Ε, είναι πολύ μάλιστα πιθανό η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρειαστεί να ναι, ναι. αποκαταστήσει τις οικονομικές, ε, τα οικονομικά ελλείμματα ούτως ή άλλως. Εγώ λοιπόν υποστηρίζω όλους τους συναδέλφους που έκαναν έκκληση και κάνω κι εγώ έκκληση για μια νέα όθηση για μια ειρηνική λύση της ισραηλινο σύγκρουσης που βεβαίως θα βασίζεται στην λύση των δύο κρατών. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πουγιοτρόφσκι για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, παρά το γεγονό ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα ε, είναι σε ισχύ και ρυθμίζει του όρου διεξαγωγή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία και άμυνα, δεν έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικά. Μπορεί να άλλαξαν όνομα οι διπλωματικέ υπηρεσίε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αναλάβει δράση ουσιαστικά, δεν έχει ενισχύσει τη θέση ω παράγον διεθνή σκηνή. Ε, θα μάλιστα αν υπάρξει πραγματικά δυνατότητα για εξωτερική πολιτική κοινή μεταξύ 27 κρατών μελών προκύπτει μια σχετική αμφισβήτηση από την έκθεση αμφισ... ότι ε, δηλαδή δεν υπάρχει βούληση ε, από πλευρά των κρατών μελών για μια κοινή εξωτερική πολιτική και μάλιστα ορισμένοι έχουν μάλλον ε, αποσχιστικέ τάσεις τάσεις φυγής δηλαδή από την κοινή αυτή πολιτική. Και διαπιστώνουμε και με την έκθεση του Γκουαλτιέρη ότι πολλά ακόμη και αμυντικά προγράμματα επικαλύπτουν το ένα το άλλο, επαναλαμβάνουν το ένα το άλλο και ουσιαστικά αποτελούν ε, σπατάλη, διασπάθηση δημόσιου χρήματο. Η μόνη πραγματικά ενωμένη δύναμη είναι το ΝΑΤΟ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και ίσως θα έπρεπε να κοιτάξουμε και αυτές τις απόψεις που εκφράζονται υπέρ της διάλυσης του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ ο κύριος Μπίτικοφερ για μισή λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Άστον πολύ καλή έκθεση του κυρίου Γκουαλτέρη για την κοινή, για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, ε, η οποία καταγράφει την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να ορίσω τις προτεραιότητες που θα πρέπει να μας καθοδηγήσουν τα επόμενα χρόνια στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Πρώτον, θα πρέπει να ε, ορίσουμε, να, αξιολογήσουμε ρεαλιστικά τους στόχους μας με μια εξωτερική αξιολόγηση και να εγγράψουμε τους στόχους αυτούς στην περιφερειακή μας πολιτική μέσα σε απλές έννοιες και ιδιαίτερα όσον αφορά το κέρας Αφρικής. Δεύτερον θα πρέπει να αναπτύξουμε ε, πρόοδο ως προς την ε, ενοποίηση και κοινή αξιοποίηση στρατιωτικού δυναμικού, στρατιωτικών δυνάμεων και οι ιδιαιτερότητες που έχουν επιλέξει, οι ιδιαίτερος δρόμος που έχουν επιλέξει η Γαλλία και η Βρετανία να εγκαταληφθούν για να ενταχθούν οι χώρες αυτές σε μια κοινή πολιτική. Αυτά θέσετε παρακαλώ στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Πρέπει να γίνει η συζήτηση, ο διάλογος και να εξασφαλιστεί η πρόοδος. Τρίτον, χρειαζόμαστε δημόσιο διάλογο για μια νέα ε, κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας. Το κείμενο του κ. Σολάνα το 2003 ήταν μια καλή πρόταση, αλλά ο κόσμος μεταξύ έχει εξελιχθεί και αυτό χρειάζεται να γίνει αυτός ο δημόσιος διάλογος. Και τέταρτον, θα πρέπει το κοινοβούλιο, τα κοινοβούλια των κρατών μελών να συμφωνήσουν ε, για, μια κοινή, για ένα κοινό κοινοβουλευτικό έλεγχο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Εάν το επιτύχουμε αυτό, εσείς κύριε Άστον, όπως και εμείς το Κοινοβούλιο, εάν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε αυτά τα τέσσερα σημεία και να τα προαγάγουμε σε μια κοινή, εξωτερική, κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας, μέσα σε ένα χρόνο θα έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Στέρο για ένα λεπτό. Ε, θα ήθελα, θα ήθελα λέγω, να συγχαρώ την κυρία Άστον για την παρουσία της και να την ευχαριστήσω. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω το λόγο εδώ και γι' αυτό χαιρετίζω και όλους τους συναδέλφους. Τώρα πρέπει να πω ότι χρειάζεται, είναι απολύτως απαραίτητο να μπορούμε να μιλήσουμε με μια φωνή γιατί είναι θέμα αξιοπιστίας της Ένωσης. Το θέμα βέβαια είναι να δούμε ποιος θα εκπροσωπεί την Ένωση ή ποια η οποία κανονικά εκπροσωπείται από τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τη δημιουργία πολλαπλών δομών και οργάνων αν δεν χρειάζονται. Πρέπει να δούμε ίσως τι πιστεύουν και οι πολίτες για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόβατς για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συνθήκη της Λισαβόνας με τις περίπλοκες τροποποίησεις της δυσχεραίνει ιδιαίτερα το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδίως λόγω των πολλών αλλαγών και τα θεσμικά όργανα δεν μπορούν να δράσουν. Ε, κυριαρχεί το χάος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε γιατί θα πρέπει να δώσουμε εξουσίες ε, στην εξωτερική υπηρεσία ε, δράση, στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, όταν ακόμα δεν έχει συσταθεί καταλήλως. Ε, τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο χρειάζονται άμεσα μέτρα. Αυτή τη στιγμή εμείς ακόμα συζητάμε την υπηρεσία και ακόμα δεν κατορθώνουμε να συμφωνήσουμε. Άρα η υπηρεσία δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Τη συστήσαμε αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να είναι εν πλήρη λειτουργία και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η λειτουργία, η σωστή δε λειτουργία της υπηρεσίας. Δυστυχώς η χώρα που έχει την Προεδρία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δώσει ένα νέο έναυσμα στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας και επομένως είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξουμε και το έργο της υπάρξης εκπροσώπου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπροκ για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Κομισιόν, κυρίες και κύριοι. Κυρία Άστον, αν θέλετε να υπάρχει μεγαλύτερη, λειτουργία, μεγαλύτερη υποστήριξη για τη λειτουργία τη υπηρεσία εξωτερική δράση, θα πρέπει να είναι πιο λειτουργική και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί η σύνθεση των αντιπροσωπιών. Δηλαδή, παρά το γεγονό ότι έχει περάσει πολύ λίγο χρόνο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα τη συμπληρώση των υπηρεσιών τη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είδε να λειτουργούν τα κράτη-μέλη ανεξάρτητα. Δεν υπήρξε η ευρωπαϊκή σημαία στην πλατεία Ταχρήρ, όπω ξέρουμε όλοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Αυτό είναι το δικό σα καθήκον, το οποίο εσεί πρέπει να φέρετε σε πέρα. Γιατί οι θέσει αυτέ οι οποίε ε, προέκυψαν από τη συνθήκη τη Λισαβόνα και εσείς φοράτε τρία καπέλα βάσει αυτών των θέσεων, θα πρέπει να οδηγήσουν και σε μια πολιτικά ηγετική αντιμετώπιση από τη δική σας πλευρά. Πρέπει να της δώσετε μια μεγάλη, μεγαλύτερη εμβέλεια και ακτινοβολία και να είσαστε πιο πιστικοί στην άσκηση των καθηκόντων σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα <clears throat> σημαντικό όταν βλέπουμε τα γεγονότα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Βλέπουμε ο κύριος Αλμπερτίνη να μιλάει για μια πολυγονική ε, ε, ένα πολυγονικό διαμερισμό της εξουσίας. Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει αυτό τον τριγωνικό χαρακτήρα που αναφέραμε και προηγουμένως. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια σωστή κατανομή ε, καθηκόντων. Αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κρίση, μια κρίση στην Ουκρανία, ένα πόλεμο Αρμενία-Αζερβαϊτζάν. Έχουμε τα τεράστια προβλήματα στον αραβικό κόσμο που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Πώ θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά όταν προκύπτουν <clears throat> ενέργειες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ανάφλεξη. Εγώ δεν είμαι εναντίον του να υπάρχει υποστήριξη παραδείγματο χάρη σε χώρες όπως το Ιράκ, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε παράλληλα θέματα όπως αυτό της επίθεσης κατά του καταβλισμού του Ασράφ. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει μια κατάσταση η οποία είναι ρευστή και πολυεδρική με έναν τρόπο ο οποίος είναι πράγματι ε, πιστικός και που θα έχει ένα πολιτικό ρόλο. Ξέρω ότι υπάρχει πολλές φορές η ανάγκη της ομοφωνίας στο Συμβούλιο των Υπουργών. Αυτό κάνει ακόμα πιο έντονη την ανάγκη να παίξετε ένα ηγετικό και πιστικό ρόλο, κυρία Άστον. Ευχαριστώ Χάουιτ για mm. λεπτό τώρα. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την ύπατη εκπρόσωπο για την προσωπική της επιτυχία στην επίτευξη συμβιβασμού στον ΟΗΕ. Οποτεδήποτε εδώ μέσα, ό,τι και να σκεφτόμαστε εδώ μέσα για την εξωτερική πολιτική, πρόκειται ούτως ή άλλως για μία επιτυχία με βάση όλα όσα είχαμε ζητήσει για τη συνθήκη της Λισαβόνας κλπ. Πρόεδρε, ως σοσιαλιστής συντονιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ήθελα επίσης να τη συγχαρώ για την στρατηγική αναθεώρηση ε, της, των, της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συμπερίληψη των θεμάτων αυτών σε όλες τις συμφωνίες στο κοινοβούλιο μας είχαμε ζητήσει τη δημιουργία μιας διεύθυνσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας. Την ευχαριστούμε λοιπόν για την προσπάθεια αυτή. Η, ξέρω ότι η κατάργηση της θανατικής ποινή θεωρείται από εκείνη προτεραιότητα όπως και για μας. Το αίτημα για μεγαλύτερη ορατότητα της Ένωσης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σημαίνει ότι η Ένωση πρέπει και να μιλά και να δρά υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον σεβασμό τους παντού. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι υποστηρίζουμε την στήριξη των Παλαιστινίων με φορολογικά έσοδα. γιατί έτσι με τέτοια βήματα θα δημιουργηθεί κάποτε η απαραίτητη κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, ο κύριος Γιατενμάκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα γεγονότα στη Βόρεια Αφρική έχουν καταδείξει πόσο σημαντική είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Βρίσκεται ενώπιον σημαντικέ προκλήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την δημοκρατία. αλλά δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδηθεί σε ένα αγώνα κατά των ανεμομήλων όπως ο Δον Κιχώτης. Έχουμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση ότι το 70% του εμπορίου όπλων περνάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πουλάμε όπλα στην Τινησία, στο Μπαχρέν, στο Σουδάν. Μήπως θα ήταν επιτέλους καιρός να σταματήσει αυτή η αντιμετώπιση και να υπάρξει μια κατά προτεραιότητα απαγόρευση της εξαγωγής όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι μια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε λοιπόν όταν υπάρχει μια ανταρσία σε ένα πλοίο να θεωρούμε υπεύθυνο μόνο τον καπετάνιο. Όλοι, όλοι μπορεί να έχουν ευθύνη, αλλά περιμένουμε από τον επικεφαλής μιας υπηρεσίας τουλάχιστον να πάρει μια πρωτοβουλία και να προσπαθήσει να αποτρέψει μια κατάσταση η οποία είναι αρνητική. Στίβενσον για ένα λεπτό κυρία Πρόεδρε. Η Λέδη Άστον μετά από την φοβερή σφαγή στις 8 Απριλίου στο Ασράφ, η κατάσταση στο Ασράφ παραμένει κρίσιμη. Μπορούσε ανα πάσα στιγμή να γίνει ακόμα μια αιματηρή επίθεση. Εγώ μόλις γύρισα από τη Βαγδάτη, όπου μετέβη μια μικρή μονάχα αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών για συζητήσεις υψηλού επίπεδου με τον πρόεδρο του Ιράκ. Προσπαθήσαμε να επιτύχουμε μια λύση για την κρίση του, του καταβλισμού Ασράφ. Την έχετε δει την πρότασή μας που εμπλέκει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Έθνη και που συνίσταται σε υποστήριξη της ε, μετακίνησης των 3.400 ε, προσφύγων του Αστράφ στον Καναδά, οι Ηνωμένε Πολιτείε, στην Ελβετία, στην Νορβηγία και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου αυτά τα άτομα έχουν κάποιες οικογενειακές σχέσεις. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αποτρέψουμε άλλη μία ανθρωπιστική καταστροφή. Και οι ίδιοι οι ευρισκόμενοι στο ΑΣΡΑΦ συμφώνησαν σε μια τέτοια λύση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δράξει αυτή την ευκαιρία να σώσει αθώες ζωές και να αποτρέψει περαιτέρω αιματοχυσία στο ΑΣΡΑΦ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάμπελ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η μέρα της Ευρώπης ε, υποτίθεται ότι θα ήταν μια εορτή για την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Δεν ήταν. Απλώς αντικαθιστούμε τα ευρωπαϊκά έθνη με έναν υπερεθνικό οργανισμό. Αυτό δεν συνάδει με τη διακυβερνητική ε, μορφή συνεργασίας όπου υπάρχει συνεργασία χωρίς να εκχωρούνται εξουσίες τα Ηνωμένα Έθνη συμφώνησαν να μην υπάρχει ζώνη απαγόρευση φτήσεων και υπήρχαν χώρε οι οποίες ηγήθηκαν όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ κάποιες άλλες χώρε, η Γερμανία για παράδειγμα, αποφάσισαν να μην συμμετέχουν στη διαδικασία. Το ΝΑΤΟ τώρα αποφάσισε να συμμετέχει. Σε αντίθεση, το η Υπερεθνική Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά της ε, περιοχής ε, ε, Απαγόρευση πτήσεων και η ίδια η Βαρόνη, η Άστον ε, ήταν κατά της απαγόρευσης ε, πτήσεων και θεωρούσε ότι ήταν μια απελπισμένη προσπάθεια. οι υπερεθνικοί οργανισμοί ε, απλώς χάνονται ενώ οι διακυβερνητικές οργανώσεις δρούν διακυβερνητικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάουρο τώρα για δύο λεπτά. Κυρία εκπρόσωπε, έχετε ένα πολύ δύσκολο έργο αναλάβει και στους ώμους σας βαραίνει ένα τεράστιο βάρος. Θα ήθελα να λάβετε τις ερωτήσεις μου όχι ως προκλήσεις, αλλά ως συνεισφορά για περισσότερη σκέψη. Στο τέλος της κοινή συζήτηση θα ψηφίσουμε την έκθεση για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ε, ε, ε διεθνείς οργανισμούς. Δύο χρόνια πριν, ε, πριν στην ακρόαση για την ε, ανάληψη των καθηκόντων σας, σας ρώτησα τι άποψη έχετε για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα νέο φορέα στον ΟΗΕ. Μου είχατε απαντήσει τότε ότι δεν είχατε προλάβει να το σκεφτείτε. Στην έκθεση μου Ορκίσα αναφέρεται η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματος. Ποια είναι η δική σας η θέση πλέον σήμερα. Είχατε χρόνο να το σκεφτείτε τα τελευταία δύο χρόνια. Κύριε Άστον, στις 17 Μαΐου θα εορταστεί στη Βαγδότη η ημέρα Ευρώπης-Ιράκ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στο Ιράκ με δύο υπαλλήλους και μία πρέσβυρα τρεις ανθρώπους οι οποίοι δρούν μέσα στο βρετανικό πλαίσιο. Εσείς θέλετε να βρείτε πόρους για να επιλύσετε την κατάσταση. Σας επισημαίνω ότι για να σας βοηθήσω ότι Στη Δαμασκό έχουμε 7 υπαλλήλους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι διαφορά υπάρχει σε σχέση με τη Βαγδάτη. Δεν θα ήταν καλύτερα να είμαστε περισσότεροι στην ε, Βαγδάτη και να είμαστε παρόντες στις 17 του μηνός, διότι θα έχουμε την πρώτη ε, εορτή μετά από την εποχή του Σαντάμ και ίσως να επιλύσουμε και τα όσα συμβαίνουν στο στρατόπεδο Ασράφ για να μπορέσουμε να βρούμε με τη συνεισφορά σας μια θετική λύση επί του θέματος. Κύριε Άστον, αναφερθήκατε και στο θέμα των Αιγυπτίων κοπτών, αλλά το στοιχείο αυτό είναι ένα στοιχείο που ανησυχεί ε, του σενάριου που αποκαλούμε άνοιξη ε, του αραβικού κόσμου. Στην Αίγυπτο πεθαίνουν μόνο χριστιανοί και καίγονται μόνο εκκλησίες, χριστιανικές εκκλησίες. Τι μας εμποδίζει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα και να πούμε τα πράγματα με το όνομά της και να δούμε ότι οι κόπτες είναι εμπλεγμένοι σε μια διαδικασία πολιτικού φονταμεταλιστικού σκοπού. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παντσέρη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι αναταραχές οι οποίες ε, διαμορφώνουν την πολιτική γεωγραφία της άλλης πλευράς της Μεσογείου με τις ανησυχίες και τις ε, ελπίδες ε, καλούν ακόμα περισσότερο να υπάρχει μια εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να βασίζεται σε μια εξωτερική πολιτική η οποία θα είναι συνεκτική και θα μπορέσει να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο μέλλον και ένα προβληματικό παρόν το οποίο θα αλλάξει εις βάθος τον κόσμο. Εν ώψη λοιπόν τη στρατηγική θέση χωρών όπω των ΗΠΑ, τη της Κίνας ε, και τη Ρωσία ε, και το γεγονό ότι υπάρχει συνεχή έλλειψη ενεργειακών πόρων, η Ευρώπη θα πρέπει να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό και αποφασιστικό ρόλο. Είναι προφανέ λοιπόν ότι είναι προετοίμαστοι για αυτά τα καθήκοντα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό οδεύουμε πάρα πολύ αργά προ ε, ένα κοινό προσανατολισμό των εξωτερικών πολιτικών των κρατών μελών, αλλά δεν έχει γίνει ουσιαστικό προ... ουσιαστική πρόεδρο Αφενός υπάρχουν μαρτυρίες από τα όσα γίνεται με τη δική σας εξωτερική πολιτική και από τα όσα κάνουν κάποιες χώρες οι οποίες νοσταλγούν μια απικιακή περίοδο στην οποία δεν μπορούμε να επανέλθουμε πλέον ποτέ και ε, ε, κάνουν τα πάντα μόνοι τους χωρίς να εκχωρούν καμία εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Εσείς έχετε ένα συγκεκριμένο καθήκον το οποίο θα πρέπει να διεξάγετε όσο το δυνατόν καλύτερα και να σας πω ότι εξαντλούνται και τα χρονικά περιθώρια πολύ σύντομα. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας επισημάνω αναλαμβάνοντας τα ενία της Προεδρίας, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι στον κατάλογο των αγορητών και δεν θα ήθελα να φτάσουμε στην κατάσταση στην οποία φτάνουμε συνήθω, το γεγονό δηλαδή ότι προβλέπονται στι 12.30 ψηφοφορίε και για να μην ακουστεί τίποτα από όσα λένε ούτε οι ομιλητέ ούτε ε, όσοι είναι εδώ παρέτηση και πρέπει να απαντήσουν ε, και δεν θα ακούγεται κανεί. Σα παρακαλώ να είστε πολύ αυστηροί με τα χρονοδιαγράμματα, αλλιώ θα σα διακόπτω. Έχει το λόγο για ένα λεπτό ο κύριο Κάτσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυριάστον, Άστον, οι πολιτικές φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινή πολιτική εξωτερικών θεμάτων και ασφάλειας είναι γνωστές. Αυτό όμω θα πρέπει να γίνει και πραγματικότητα και σα προσκαλώ να επισκεφτείτε το ταχύτερο δυνατό το Ιράκ. Είναι απαραίτητο να πάτε στο, στη Βαγδάτη, στο Κουρδιστάν. Φεύγουν οι Αμερικανοί, εγκαταλείπουν αυτέ τι τοποθεσίε μέχρι το τέλο του χρόνου. Θα έχουν φύγει, θα δημιουργηθεί ένα κενό και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόλυτα απούσα. Δηλαδή δεν είναι καν ορατοί και ούτε μπορούν να γίνουν ορατοί οι διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ. Χρειάζεται την προσωπική σας παρουσία, χρειάζεται την πολιτική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται και την οικονομική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας συγχαρώ για τη σημερινή σας δήλωση για τη Βοσνία Ζεχοβίνη. Έχετε θέσει τα πράγματα πολύ σωστά, αλλά ακόμα δεν έχετε διορίσει τον επικεφαλή τη αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σεράγεβο. Αυτό είναι μια ευκαιρία για ορισμένου που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την Βοσνία Ζεγοβίνη και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Αυτό θα σταματήσει με τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Κάουελ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υψηλή Εκπρόσωπε, η Ευρώπη αντιμετωπίζει δύο προβλήματα αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, χρειάζεται μια νέα αντιμετώπιση για την εξωτερική πολιτική. Ήμουνα στην Τινησία πρόσφατα και γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλέ προσδοκίε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι επίση σε μόνιμη επαφή με την Ουκρανία. Και η Ουκρανία αναμένει πολύ περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερε δυνατότητε θέλουν να γίνουν περισσότερα σε συνεργασία με την Ευρώπη. Δεν πρέπει να δείξουμε εγωισμό στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Ξέρω, κυρία Ήπατη, εκπρόσωπε, ότι και εσείς έχετε να αντιμετωπίσετε το ότι κάποιοι άλλοι αποφασίζουν πολλές φορές την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό σας. Σαν παιδάκια είμαστε μερικές φορές. Τη μια μέρα παίζουμε με την Λευκορωσία. Την άλλη μέρα τα έχουμε ξεχάσει και ενδιαφερόμαστε για τη Βόρεια Αφρική. Εσείς δείξατε ότι είσαστε μια στεναρή ε, προσωπικότητα και μπορεί, μπορείτε να πάρετε πρωτοβουλία, μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι έχουμε μια φιλόδοξη και συνεκτική πολιτική αντιμετώπιση. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε μόνο τα θέματα της μετανάστευσης. Δεν θα πρέπει να κάνουμε σαν τους αρχαίους Ρωμαίους οι οποίοι προστατεύανε μονάχα ένα σύνορο και όχι ένα άλλο. Δύο λεπτά ο κύριος Σάιρος Βόλσκι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Άστον μου, οι βιαιότητες που σημειώνονται μας ανησυχούν ιδιαίτερα αλλά το ερώτημά μας είναι με τι όργανα, με εργαλεία θα τις αντιμετωπίσουμε. Εμπορικά μέτρα, τι άλλους μέτρα. Μήπως υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από την πυθό η οποία φαίνεται ότι δεν καταλήγει σε τίποτα. Νομίζω ότι αυτό είναι από τα σημαντικότερα τμήματα της εντολής σας. Αν αποτύχουμε εκεί θα αποτύχουμε σε όλη την εξωτερική πολιτική. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αμυντική θέση. λέει Άστον. Οι μεγαλύτερες καταιγίδε έχουν συμβεί στην άμεση γειτονία μας. Τι μας λέει λοιπόν η πολιτική μετεωρολογία. Για τρίτη φορά καθυστερεί ε, σημειώνονται καθυστερήσεις χωρίς να φταίτε εσείς μάλλον από την υπηρεσία σας αλλά η εξωτερική πολιτική είναι κάτι που πρέπει, που υποτίθεται ότι αλλάζει τον ρου της ιστορίας όχι δεν περιορίζεται σε κενές δηλώσεις χρησιμοποιούνται και σκληρά και μαλακότερα μέτρα όπως για τη Συρία το Ασράφ ίσως χρειάζονται τα σκληρότερα Νομίζω ότι έχετε λανθασμένη προσέγγιση γενικά γιατί καταδικάζετε την πολιτική μας πάντοτε στο χαμηλότερο κοινό παρονομαστή και στην αιώνια καθυστέρηση. Εμείς θέλουμε ηγεσία, ηγετικό ρόλο, όχι ουραγού. Πολύ συχνά ικανοποιούμαστε, περιοριζόμαστε να καταδικάζουμε και να εφαρμόζουμε απλώς θεωρήσεις, μέτρο το οποίο είναι πλήρως αναποτελεσματικό. Δεν υπάρχουν επενδύσεις αραβικών χρημάτων στην, για την αραβική δημοκρατία όμως. Ευχαριστούμε κύριε Βόλσκι, Σάριους Βόλσκι, ο κύριος Ρούτσεκ. Ε, Άστον. Τι θα γίνει στη Βόρεια Αφρική. Αυτά που γίνονται στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή είναι ζωτικά Εκεί πολλά έθνη κερδίζουν την ανεξαρτησία τους αυτή τη στιγμή. Οι νέοι από την Τινησία μέχρι την Ιεμένη και τον Μπαχρέιν ζητούν περισσότερη ελευθερία, περισσότερη δημοκρατία, περισσότερα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμφέρον μας είναι λοιπόν και από άποψη ασφαλείας αλλά και ηθικά να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες αυτές των νέων για απελευθέρωση και αυτοδιαχείριση. Γιατί αυτές είναι και οι δικές μας αξίες. Η υποστήριξη των αξιών αυτών είναι βασικό στοιχείο για τη διατήρηση της ειρήνης και της ευημερίας στον κόσμο. Δεν εννοεί αυτό βέβαια ότι ζητούμε παρέμβαση, απλώς πιστεύουμε ότι η δημοκρατία και η ένωμη τάξη και το κράτος δικαίου είναι κάτι το οποίο έχουν δικαίωμα και υποχρέωση και οι ίδιοι οι αραβικοί λαοί να ζητήσουν και να εφαρμόσουν. Κυρία Ρόιτερ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Λέει Άστον, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να σα συγχαρώ, Λεδιάστον, για την μεγάλη σα επιτυχία στη Νέα Υόρκη. Είναι θετικό το γεγονό ότι το έργο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΟΗΕ ενισχύθηκε. Δημιουργούνται βέβαια κάποια ερωτηματικά. Ποιο είναι το μήνυμά μα, αλλά και το μήνυμά σα στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και πώ θα συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί να υπάρχουν και κάποιε αντίθετε απόψει πώς θα μπορέσουμε να μεταφράσουμε το μήνυμά μας σε έργα, όπως ρώτησε και ο κύριος Ντόλ. Βρισκόμαστε ενώπιον τεραστίων προκλήσεων στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Οι προκλήσεις δεν υπάρχουν μόνο στο Μπαχρέιν, στην Ιεμένη, στο Ιράν και στην Αρμενία, αλλά και στην άμεση γειτονία μας. Η Ρωσία, η Συρία, η Αίγυπτος, η Λιβύη, και είναι πολύ συγκεκριμένε οι προκλήσει. Υπάρχουν ε, καταπιεστικά καθεστώκα, τα ε, ε, επιθέσεις κατά θρησκειών, υπάρχουν ε, ροές μεταναστών στις ακτές μας και αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες αντιδράσεις βέβαια και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κράτο δικαίου σε κάποιες χώρες εσείς, ε, διάστον, Άστον, είστε ε, η φυσιογνωμία που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να είμαστε διχασμένοι και να μείνουμε ε, στα μετόπισθεν. Εσείς είστε σημαντικοί και ο ρόλος σας είναι θεμελιώδης. Ε, θα πρέπει να διεξάγετε το ρόλο σας και εντός αλλά και εκτός ε, των αιθουσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ιδίως εκτός. Πολλές φορές θα πρέπει να κάνετε ε, ταξίδια αλληλεγγύης, αλλά εμείς σας υποστηρίζουμε διότι θα πρέπει να πείσετε τα κράτη-μέλη ότι μια κοινή ευρωπαϊκή θέση αξίζει τον κόπο για να έχουμε μια συνεκτική κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Εσείς θα πρέπει να είστε ο άνθρωπος που εκπροσωπεί αυτή την πολιτική. Κύριε Πρόεδρε, Χρειαζόμαστε καλύτερους ανθρώπους ε, στην ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και τις ευρωπαϊκές θέσεις και θα πρέπει να γίνουν κάποια περισσότερα πράγματα επί παραδείγματι στη Συρία. Δεν ε, αναφερόμαστε σε οι λύσεις. Διακόπτεται η ομιλήτρια κυρία Κοπάγια. Τώρα συζητάμε τα κορυφαία θέματα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης αλλά και τρία σημαντικά κείμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο όμως το ερώτημα που όλοι θέτουν στη σημερινή συζήτηση είναι αν στην πραγματικότητα υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική. όταν στο ιστορικής σημασίας γεγονός των τελευταίων δεκαετιών που είναι η εξεγέρση στον αραβικό κόσμο η ευρώπη άργησε να βρει το βηματισμό της και υπήρξε δειλή άτολμη και για μεγάλο διάστημα άφωνη όταν στο κρίσιμο ψήφισμα 1973 του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Λιβύη οι χώρες της Ένωσης δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν ενιαία στάση, όταν η Ένωση διστάζει στη Συρία, αναρωτιέμαι μήπως το ερώτημα έχει ήδη απαντηθεί στην πράξη. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας οι ελπίδες ήταν μεγάλες. Όταν όμως το Συμβούλιο δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, όταν οι εθνικές ιδιοτέλειες και προσωπικές στρατηγικές κυριαρχούν στη λήψη των αποφάσεων το ότι η ευρώπη και η ευρωπαϊκή ιδέα έχουν χάσει άλλη μία μάχη. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κοπά. Ένα λεπτό, ένα μισή λεπτό μάλιστα, ο κύριος Γκάλερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, με, βλέποντας τη λυπηρή έλλειψη σύμπνοιας ε, πολλών κυβερνήσεων ενώπιον των τωρινών προκλήσεων, εγώ συμφωνώ με αυτά τα οποία είπαν πολλοί συνάδελφοι, αλλά και η κυρία Άστον, ότι η συζήτηση θα πρέπει να συμπεριλάβει και τις εθνικές κυβερνήσεις και θα πρέπει να δούμε γιατί κάποιες κυβερνήσεις μπλοκάρουν τις αποφάσεις ή τις στρέφουν προς τα εθνικά τους συμφέροντα. Όλα αυτά εμποδίζουν το να μπορέσει να υπάρξει μια κοινή αντιμετώπιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα τη εξωτερική πολιτική. σω θα πρέπει κάποιε κυβερνήσει να εξηγήσουν τη στάση του. Επομένω, εγώ όμω έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι βρισκόμαστε σε μια αργή αλλά θετική πορεία που διδασκόμαστε από τα λάθη μα και που θα οδηγήσει εν καιρό σε μια καλύτερη αντιμετώπιση στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Χρειαζόμαστε να συγκεντρώνουμε τι δυνατότητέ μα και να τι μοιραζόμαστε. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε νέε προκλήσει ενώπιον μα. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν θα χρησιμοποιήσετε αυτές τις ε, δυνατότητες, θα προχωρήσετε με αυτές τις πρωτοβουλίες που θέλουν πιο διαρθρωμένη συνεργασία. Θα θέσετε τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας στο κέντρο αυτών των προβουλειών. Ο κ. Μπιτικόφερ ανέφερε τέσσερις προτεραιότητες για τον επόμενο χρόνο και συμφωνώ μαζί του σε μεγάλο βαθμό. <clears throat> Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να υπάρξει και μια ε, επιτροπή σοφών για τα θέματα ασφάλεια και άμυνα. Ποια είναι η άποψή σα επίση σε σχέση με την υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία. Υπάρχει μια δυνατότητα να υπάρχει ένα ενιαίο στρατηγείο για την υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων. Ο κύριο Γιάννη, για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, κυρία Άστον, θέλω να σας συγχαρώ για το έργο που έχετε φέρει σε πέρα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι σαν Μέρμιγκας καταφέρατε να συλλέξετε όλα τα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε μια πιο επωφελή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι πρέπει να εμβαθύνω περισσότερο σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι από τη δική μου πολιτική ομάδα και θέλω να σταθώ περισσότερο σε τέσσερα, τέσσερα σημεία που νομίζω ότι είναι ένας μοχλός δράσης για σας και στοιχεία στα οποία μπορείτε να βασιστείτε για να έχετε μια εξωτερική πολιτική η οποία να είναι άξια του ονόματός σας. Ένα από αυτά είναι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Αντίθετα από άλλα ζητήματα, στο συγκεκριμένο αυτό θέμα, 65 <clears throat> ή 70% των Ευρωπαίων πολιτών υποστηρίζει μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Δεύτερο, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου μόνο μια μικρή ευρωσκεπτιστική ε, μειοψηφία δεν υποστηρίζει μια ομοσπονδιακή και κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Τρίτον, έχουμε τα κράτη-μέλη τα οποία είναι τα πιο φεδεραλιστικά, πιο ευρωπαϊστικά. Κάντε μια συμφωνία, κάντε μια συμμαχία μαζί τους, τον διακόπτη ο Πρόεδρος. Τελείωσε ο χρόνος σας. 1,5 λεπτό ο κύριος Μιγιάν Μόν. Δεν έχετε το λόγο κύριε Γιάννη. Πέρασε ο χρόνος σας. Ο κύριος Μιγιάν Μόν έχει το λόγο του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο προηγούμενε ε, παρατηρήσεις Μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά χωριστά ή από κοινού. Έχουμε χωριστά θέματα τα οποία αξίζουν το καθένα μία σε βάθο συζήτηση. Και κατά τα άλλα, εγώ θέλω να υποστηρίξω αυτά που είπε ο κύριος Σαλαφράγκα για το θάνατο του κυρίου Σότο, του κουβανού αντιφρονούντα. μερικές ακόμα παρατηρήσεις Δυστυχώ όταν θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερη ένταση στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορροφά την προσοχή μας η χρηματοοικονομική κρίση. Αλλά έχουμε πολλές ε, νέες εξελίξεις και γεγονότα στη γειτονιά μας, ιδίως στη Μεσόγειο και αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι παρούσα σε όλες τις διαδικασίες αλλαγής του αραβικού κόσμου. Χαίρομαι κυρία ε, Άστον που την προηγούμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη ενισχύθηκε η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη. Συγχαρητήρια η αποτυχία του προηγούμενου έτους είχε οδηγήσει σε ανησυχητικά ερωτηματικά για το μέλλον τη Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο και στους διεθνείς φορεί. Όλα αυτά όμως σημαίνουν ότι και η απόκληση απόψεων των ευρωπαϊκών κρατών στο ψήφισμα 1973 του ΟΗΕ δείχνουν πόσο τεράστιε είναι οι δυσκολίε που μα χωρίζουν ακόμα από την επίτευξη μια κοινή εξωτερική πολιτική. Εσεί, κύριε Άστον και ο κύριο Φαν που έχει αυτός αυτό μεγάλε αρμοδιότητες για τα εξωτερικά θέματα <clears throat> έχετε το δύσκολο ε, εγχείρημα να πείσετε τα κράτη-μέλη για μια ενωμένη και συνεκτική δράση και οι δύο πρέπει να κάνετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να πιέσετε τα κράτη-μέλη να παίξουν το ρόλο τους σε μια δύσκολη στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τα στοιχεία και τα εργαλεία της συνθήκη Λισαβόνας. Ένα λεπτό για τον κύριο Σίβιετσι. Κυρία, είπατε εκπρόσωπε, αντιλαμβανόμαστε όλοι το γεγονός ότι η κοινή εξωτερική πολιτική ε, πότε υπάρχει και πότε δεν υπάρχει. Όταν μιλάμε για πολιτική γειτονία, έχουμε κοινή πολιτική. Αλλά όταν μιλάμε για την Βόρεια Αφρική, στην πράξη η Δύση δεν έχει καμία αξιοπιστία. Την αξιοπιστία την έχουν οι χώρες οι ανατολικέ, οι οποίες έκαναν αντίστοιχε επαναστάσει. Εμεί έχουμε μια καλύτερη οπτική των πραγμάτων, αλλά υπάρχουν τα παλιά κράτη-μέλη που έχουν τα κονδύλια. Χρειάζονται λοιπόν κονδύλια για να γίνει πιο αξιόπιστη και η πολιτική γειτονία. Όταν αναφερόμαστε σε πολιτική άμυνας δε, ποια είναι αυτή η πολιτική άμυνας ε, σε μια Ευρώπη που δεν έχει όπλα. Έχουμε ευρωπαϊκά αεροσκάφη τα οποία πετούν στη Λιβύη, ε, τα οποία είναι παλιά τεχνολογία και μπορεί να, δεν μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά στην αποστολή. Αν δεν είχαν εμπλακεί οι Αμερικανοί εξ αρχή, δεν θα είχαμε κανένα αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη αποστολή. Δεν θα έχουμε λοιπόν κοινή πολιτική άμυνα αν δεν υπάρχουν όπλα, αν δεν υπάρχει και κοινή πολιτική για την ασφάλεια και την άμυνα. 1,5 λεπτό ο κύριος Ντανζάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπατή εκπρόσωπε. Αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δείχνουν ακόμη μια φορά ότι η Ευρώπη είναι ανίκανη να αντιδράσει στρατιωτικά και πολιτικά. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά που θα θέλαμε να εκφράσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης τα κράτη-μέλη φέρουν μεγάλο μέρος της ευθύνης για αυτή την ανικανότητα οικοδόμησης μιας συνεπούς και αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής ενώ και οι ίδιοι οι Αμερικανοί σε εμά έστρεψαν τα μάτια τους. Οι σημαντικές γεωπολιτικές και στρατηγικές εξελίξεις όμως μας υποχρεώνουν να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτά που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας και της οποίας εσείς είστε εκπρόσωπος και εγκυήτρια Έχουν σημειωθεί πολλές διεθνείς κρίσεις και δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από το να αναλάβουμε μόνοι μας να πάρουμε στα χέρια μας την τύχη μας οι φίλοι και σύμμαχοι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ δεν είναι ικανοί ούτε εκείνοι δεν μπόρεσαν να τερματίσουν την κρίση στη Γεωργία παραδείγματο χάρη πράγμα για το οποίο πολλά περισσότερα μπόρεσε να πράξει η Ευρώπη και για τη Λιβύη επίσης οι Αμερικανοί δεν θέλησαν να είναι στην πρώτη γραμμή αλλά δεν αρκεί γι' αυτό να αντιδράσουμε με μινιμαλιστικό τρόπο η κοινή πολιτική που θέλουμε να εφαρμόσουμε στα εξωτερικά είναι μια αναγκαιότητα, στρατηγική αναγκαιότητα και πρέπει εσείς να αναλάβετε πρωτοβουλίες στον τομέα αυτών. Ευχαριστούμε κύριε Ντανζάν. Για 1,5 λεπτό ο συνάδελφος Κοβατσέφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία μόνο τώρα έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ποιε είναι οι υποχρεώσει που επιβάλλει σε αυτά η συνθήκη τη Λισαβόνα. και είναι καιρό επιτέλου να τηρήσουν αυτές τι υποχρεώσει. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να χτυπήσει τη γροθιά τη στο τραπέζι και να απαιτήσει από τα κράτη-μέλη να κινηθούν αποκινούμε στα πλαίσια της συνδίκης Λισαβόνας. Χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική ε, ευρωπαϊκή διπλωματία και αποτελεσματική λειτουργία και σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Μόνο έτσι μπορούμε να ασκήσουμε πίεση σε διεθνές επίπεδο και να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τα τεκτενόμενα στο παγκόσμιο στη Μια κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική και χρήσιμη και για το ΝΑΤΟ και για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις συγκρούσεις που ξεσπούν στον κόσμο. Είναι όλα αυτά σημαντικά και για την σωστή χρησιμοποίηση των πόρων και για την σωστή ανάπτυξη μιας κοινή πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν όλες τις ευκαιρίες για να υπάρχει και καλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν λοιπόν ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δρά εξ ονοματός τους και χρησιμοποιεί όλες τις πληροφορίες τους. Αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει άλλους τρόπους για να φέρει σε πέρα σε αυτό το εγχείρημα. Και εσείς κυρία Άστον θα πρέπει να απαιτήσετε στα κράτη-μέλη να δεχτούν τις συμφωνίες επανεισδοχής και να τις εφαρμόσουν στην περίπτωση που δεν τις έχουν εφαρμόσει. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. 1,5 λεπτό ο κύριος Πέτερλε. Κυρία Άστον, αγαπητοί συνάδελφοι. Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, στο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε όλο και περισσότερες προκλήσεις. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είμαστε αναξιόπιστοι δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ αποτελεσματικοί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δράσουμε επί τη βάση των αξιών και αρχών μας. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Αστών ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε πώς ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από πολλά πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τον άνθρωπο στο κέντρο όλων των πραγμάτων και επομένως θα πρέπει να δώσουμε σημασία και στον διαπολιτισμικό διάλογο. Ο κόσμος περιμένει ένα πιο έντονο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν περιμένει 27 κατακαιρματισμένες εθνικές πολιτικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χάσουμε την πολυμορφία μας. Τρία πράγματα θέλω να τονίσω. Είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα στη Βοσνία ζεγοβιν για να αποτρέψουμε περαιτέρω βία. Δεύτερον, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε μια ενιαία στρατηγική στάση εναντί της Τουρκίας. Και τρίτον, χαίρομαι πάρα πολύ για τον αποφασιστικό ρόλο με τον οποίο έχετε δράσει, κυρία Άστον. Η φωνή μα πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφή. Ευχαριστούμε, κύριε Πέτερλε. Ενάμιση λεπτό τώρα για τον κύριο Βιντάλ Κουάντρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στι 29 Ιουλίου του 2009 έγινε μία ε, παρέμβαση στο στρατόπεδο του Ασράφ ε, και σκοτώθηκαν 11 ε, κάτοικοι του καταβλισμού. Είχαμε 24 θύματα στο περασμένη επίθεση και εσείς κυρία Άστον είχατε προειδοποιηθεί εδώ και μήνες ε, από μέλη του Κοινοβουλίου ότι αυτή η τελευταία σφαγή ε, ήταν επικείμενη. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε, επανειλημμένως είχαμε ζητήσει άλλωστε την παρέμβασή σας. Εσείς ε, αγνοήσατε τις προειδοποίησεις μας και κινηθήκατε μόνο μετά από την καταστροφή. Βέβαια κάνει αργά παραποτέ, αλλά η επόμενη επίθεση θα μπορούσε να είναι ένα λουτρό αίματος ε, τεραστίων διαστάσεων, εάν από ή τώρα ήδη δεν ε, θέσετε αυτή την ανθρωπιστική κρίση μεταξύ των μέγιστων προτεραιοτήτων του προγράμματός σας. Υπάρχει μια λύση, σας την εξήγησε ο κύριος Στίβενσον, περιμένουμε άμεση και αποφασιστική δράση από πλευρά σας και είμαστε θετικά διακείμενοι στη δέσμευση που αναλύεται σήμερα το πρωί. Υπάρχουν 3.000 άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, ε, ανυπεράσπιστοι, οι οποίοι περιμένουν από εμά τη βοήθειά μας και νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουμε για να σταθούμε και στο ύψος των αξιών μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του και πρέπει να ζητήσουμε δράση. Περιμένουμε τη δράση, τη δράση μας και ε, εάν δράσετε θα σας ευγνωμονούμε. Αν όχι και η συνείδησή σας αλλά και το κοινοβούλιο εδώ θα ε, σας ε, καταδιώκει. Ο κύριος Δομινίκ Μοντής για να μην Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους έχει εφαρμόσει κυρώσεις κατά της Συρίας. Δυστυχώς φαίνεται ότι το κάνει με τρεμάμενα χέρια προσπαθώντας συγχρόνως να αφήσει άμομο τον επικεφαλής του Συριακού καθεστώτος. Αυτή η έλλειψη αποφασιστικότητα καθώς και σαφήνειες προφανώ ερμηνεύεται από τους διαδηλωτέ στη Συρία ως μια εγκατάλειψή του και από την εξουσία στη Συρία ως επίοικια που θα τους επιτρέψει να εντατικοποιήσουν την καταστολή στη Συρία. Πρόκειται για μια καταστολή τόσο βία και τόσο σκληρή που δεν μπορούμε να φανταστούμε <clears throat> ότι συγχρόνως η Συρία μπορεί να συμμετέχει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Τη στιγμή που σήμερα οι αρχές της Συρίας αρνούνται να δεχτούν εκπροσώπους και παρατηρητές του ΟΗΕ στην Τέρα που ήταν το θέατρο τρομερών ε, βιοπραγιών κατά άμαχων και ανυπεράσπιστων ατόμων. Αυτό λοιπόν είναι μια προσβολή προς τα θύματα και προς τις οικογένειάς τους και μια ενθάρρυνση στην κυβέρνηση Συρίας να χρησιμοποιήσει τα όπλα καταπατώντας όλες τις αρχές τις οποίες το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών στο οποίο συμμετέχει θα έπρεπε να είναι ο θεματοφύλακας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε λοιπόν, κυρία κυρία Άστον μάλλον, τι προβλέπετε για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την καταστροφή στη Συρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και έχουμε κλείσει λοιπόν τον γύρο των ομιλητών και περνούμε τώρα στην ε, θύρα οφθαλμών. Έχουμε 24 συναδέλφους οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο και εγώ θα δεχτώ μοναχα πέντε από αυτούς, δέκα μάλλον από αυτούς, θα το κάνουμε όμως με σύντομο τρόπο και όταν κανείς καλύπτει το ένα λεπτό θα, θα τους παίρνω το λόγο. Κύριε Μπρισάζης έχει το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι εδώ. Αφού έχω μόνο ένα λεπτό, θα είμαι σύντομη και άλλοι συνάδελφοι ανέφεραν ήδη την κατάσταση στον Αγκόρνο Καραμπάχ και σημείωσαν ότι η κατάσταση εκεί αλλάζει ριζικά τις τελευταίες εβδομάδες. Ερωτώ λοιπόν την Λέδη Άστον. Μήπως ξέρετε αν σημειώνονται στρατιωτικές κινήσεις εκεί. Γνωρίζετε πώς έχει η κατάσταση και πώς εξελίσθηκε. Κάνετε τίποτε για να προλάβετε την κλιμάκωση των πραγμάτων και εκεί και στα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας. Ευχαριστώ κυρία Αναγκόμες έχει το λόγο. Can Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια δύναμη για το νόμο και την ανθρώπινη ασφάλεια χωρίς ε, να βρίσκει τους εγκληματίες και να αφήνει τους πρόσφυγες να πεθαίνουν στη Μεσόγειο. Λέει Άστον, ε, εγκλήματα σαν αυτά δεν θα πρέπει να βρίσκονται μόνο στην προτεραιότητα στους, ε, στον κατάλογο των σοβαρών αδικημάτων αλλά θα πρέπει να δικάζονται και από τα διεθνή δικαστήρια. Στη Βενγάζη θα έπρεπε να έχετε αναπτύξει την EU4 όχι μόνο για να συνδράμετε ανθρώπους κατά των επιθέσεων όπως τη Μιζηράτα αλλά και για να μπορέσετε να διαφυλάξετε και τα σύνορα όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν χρειάζονται άλλα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και άλλα εκκλήσει. Χρειάζεται απλώς πολιτική βούληση από πλευρά κρατών μελών. Αν αναλάβετε την πρωτοβουλία, κυρία μου, και θέσετε και τις ε, χώρες μέλη ενώπιον των ευθυνών τους, θα σας υποστηρίξει στεναρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διακόπτη. Ευχαριστώ, κυρία Γκόμε. Η κυρία Παρβανόβα. Thank you. Κύριε Πρόεδρε, κυρία είπατε εκπρόσωποι, παρά το γεγονό ότι ανατηρηχέ στη Βόρεια Αφρική ζητούν δράση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεσόγειο, θα ήθελα να αναφερθώ στο δεύτερο στολίσκο ο οποίο πηγαίνει στη Γάζα. Θυμόμαστε όλοι τα αποτελέσματα τη πρώτη νιοπομπή και το γεγονό ότι χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσουμε να έχουμε έναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Ελπίζω να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση και θα ήθελα να σας θέσω, κυρία Επατή Εκπρόσωπη, την εξή ερώτηση. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τις ε, παρούσες ανθρωπιστικές ανάγκες στη Γάζα και τα όσα περνούν ε, από τα ε, σημεία εισόδου στη Γάζα και στην Παλαιστίνη. Ε, σκοπεύετε να ξεκινήσετε συζητήσεις με το Ισραήλ για να προωθήσετε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και να υπάρχει και θετικό συμπέρασμα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουμε πιο θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάουταλα. very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρία Άστον, ακούσατε σαφώς σήμερα το πρωί την φωνή του Κοινοβουλίου ότι θα σας υποστηρίξει ιδιαίτερα στο ρόλο σας στο ηγετικό και ζητά από εσά να πάρετε πρωτοβουλία στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Ακούσατε όμω και τα πολλά ερωτήματα των συναδέλφων για το ποια είναι τα κράτη-μέλη τα οποία αυτή τη στιγμή εμποδίζουν τι κοινέ μα προσπάθειε. Η πρόταση προ εμά θα ήταν τώρα που η Υπηρεσία εξωτερική δράση αρχίζει να θεσπίζει κανόνε για την πρόσβαση σε πληροφορίε και σε έγγραφα, κάντε την μια σύγχρονη υπηρεσία που να είναι προσβάσιμη στους πολίτες και που δεν αντιμετωπίζει την κοινή εξωτερική πολιτική σαν απλώς υπόθεση διπλωματών. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να υποστηρίξουμε τις κοινές προσπάθειές μας για μια πραγματικά κοινή εξωτερική πολιτική. Ευχαριστώ κυρία Χάουταλα. Ο κύριος Βαντάλεν έχει το λόγο. Τα γεγονότα. Στη Μέση Ανατολή είναι κάτι που δείχνει ότι σημειώνονται δομικές αλλαγές και το, μία από αυτές είναι η διακριτική μεταχείριση κατά των χριστιανών στις μουσουλμανικές χώρες. Σε μερικές από αυτές μπορεί να αποτελούν το 50%. Στην Αίγυπτο γίνονται επιθέσεις και γενικά καθημερινές είναι πια και είναι πια δύνατον να πάει κανείς στις εκκλησίες. Εμείς έχουμε συναντήσει κόπτες πριν από λίγο καιρό και μας ζήτησαν κατεπηγόντως βοήθεια. Σκοπεύετε να καταστήσετε τους κόπτας μία από τις προτεραιότητές σας. Στις 2 Φεβρουαρίου είχαμε ήδη ζητήσει κάτι τέτοιο, μία στρατηγική πανευρωπαϊκή για την ανεξιθρησκεία Είστε διατεθειμένοι να την πραγματοποιήσετε. Θα ήθελα να μου απαντήσετε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φιγκερέντου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολιτικές άμυνας και προάσπισης γεωστρατηγικών συμφερόντων των ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων που βρίσκονται σε απόλυτη σύμπνοια με το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένε Πολιτείε και δεν τους ενδιαφέρει η ανάπτυξη του τρίτου κόσμου. Είναι πολλές φορές καταστροφική η παρεμβασή τους όπως στην Παλαιστίνη, στο Ιράκ, στη Λιβύη και στο Αφγανιστάν. Επικρατεί μια πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών που υποστηρίζει τα οικονομικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που παράγουν εξοπλισμούς και κερδίζουν δισεκατομμύρια πολλώντας όπλα σε δικτάτορες που τα χρησιμοποιούν στη συνέχεια για να κατασφάξουν τους λαούς τους και λαούς ομόρων χωρών. Γι' αυτό δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση χωρίς να ξέρουμε αν θα τροποποιηθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εξοπλισμούς και αν θα σταματήσει πια η ε, επεκτατική πολιτική του Ισραήλ. Τέλειωσε ο χρόνος σας κυρία Φιγερέδο. Ο κύριος Πάσκα έχει το λόγο. Κυρία Άστον, όλοι μας κατανοούμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τον ουρανό μετάστρα από τη στιγμή που έχετε μόλις αναλάβει τα καθηκοντά σας. Αλλά Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να προχωρήσετε σε διαπραγματεύσεις σε ορισμένους τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει επωφελώς την πολιτική της ε, επιρροή. Ένα από τα κύρια θέματα που απασχολεί σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας από τους τομείς όπου θα μπορούσε να υπάρξει μια λύση με μια στρογγυλή τράπεζα είναι η Κύπρος όπου ο τουρκικός στρατός κατέχει ένα τμήμα της χώρας αυτής. Η Τουρκία θέλει να γίνει τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι εφόσον αυτό είναι ένα θέμα που εμπλέκει άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητές σας για να υπάρξει σωστή λύση στο πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ κυρία Πάσκα. Πρόνς. Κύριε, κύριε Άστον, ο, η εξωτερική πολιτική είναι ένα από τα βασικά στοιχεία ενός κυριαρχού κράτους. Θα το κάνουμε πολιτική μιας ένωσης, ουσιαστικά κάνει τα κράτη-μέλη να μην είναι πια κυρίαρχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό με μια πολιτική της Ευρώπης να αποτρέπει τους πολέμους. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης παραχώρηση της ε, κυριαρχικότητας των κρατών μελών. Δεν πρέπει λοιπόν να διαλύσουμε τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πόλεμοι στους οποίους δεν έχει θεμητό συμφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφεύγονται και δεν πρέπει να κάνουμε και ε, προσπάθειες για να επιβάλλουμε τις λεγόμενες ευρωπαϊκές αξίες σε ξένα εδάφη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη και την συρροή ανθρώπων από τρίτες χώρες στην Ευρώπη. Ο κύριος Σκούρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να παρέμβω για να ευχαριστήσω τη Βαρόνια Άστον για τον απολογισμό που μας έκανε σήμερα το πρωί, αλλά θα ήθελα να της πω ότι δυστυχώς η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη δεν αντιλαμβάνεται την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξωτερική μας πολιτική, όπως καταδείχθηκε σήμερα από τις παρεμβάσεις πολλών συναδέλφων, είναι ακόμα στα σπάργανα. Το βλέπουμε άλλωστε σε όσα συμβαίνουν αυτέ τι ημέρε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να απουσιάζει στο στρατόπεδο Ασράφ. Πρόκειται για ένα στρατόπεδο στο οποίο ε, μετράται όχι μόνο η διεθνής πολιτική αλλά και η, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, σε αυτό το τμήμα του κόσμου θα πρέπει να παρεύουμε όπως πρέπει να παρεύουμε και στη Συρία η Συρία αυτή τη στιγμή βιώνει μια πολύ σοβαρή κατάσταση όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι δυνατότητες ε, να αντιμετωπίσουμε ένα δικτατορικό καθεστώς θα πρέπει να βοηθήσουν με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακόπτη να ολοκληρώσουμε ε, δίνοντας το λόγο στον κύριο Ζάλα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Μόνο μία παρατήρηση θα ήθελα να κάνω. Πιστεύω ότι ο ιδιαίτερα ενεργός ρόλος της Άγκυρας μας οδηγεί σε νέες ευκαιρίες αλλά και προκλήσει για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Κυρία Υπατή, εκπρόσωπε, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ένα θεσμικό διάλογο για τα κύρια στρατηγικά θέματα όπως η ενεργειακή πολιτική, η σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και στον Κάφκασο, η πυρηνική ε, πορεία του Ιράν και η δημοκρατική αφύπνιση στη Μέση Ανατολή με την Τουρκία. Η Τουρκία μπορεί να παίξει ένα σημαντικό και επικοδομητικό ρόλο για να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εδραιώσει τα κεκτημένα της αφύπνισης των αραβικών χωρών. Αλλά αυτός ο διάλογος δεν πρέπει να υποκαταστήσει, αλλά θα πρέπει να υποστηρίξει την τουρκική πορεία στην ένταξη. Ευχαριστώ Μπόρις. Με τον τρόπο αυτό έχουμε κλείσει τους 10 συναδέλφους οι οποίοι έλαβαν το λόγο στη διαδικασία αυτή και στο συγγνώμη και από τους 14 που ήμουν στα κρύα του Λουτρού και καταλαβαίνω τη ματέωση που νιώθουν αλλά αυτά είναι τα χρονικά όρια που έχουμε. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Αλμπερτίνη, καταρχήν, ο οποίος έχει το λόγο για δύο λεπτά ως εισηγητής. Κύριε Πρόεδρε, στην πρώτη παρέμβαση είχα στη διάθεση μου τέσσερα λεπτά και εκμεταλλεύτηκα τα δύο μόνον. Ζητώ τη δυνατότητα, αφού τώρα έχω δύο λεπτά, να χρησιμοποιήσω τέσσερα για την ε, τελική μου παρέμβαση. έχετε τέσσερα λεπτά, μου λέτε ότι ε, χρησιμοποιήσετε μόνο τέσσερα, άρα μας μένουν τέσσερα, αν ναι, όντω έγινε αυτό. Στην πρώτη μου παρέμβαση, λέει ο κύριος Αλμπερτίνη, μίλησα για δύο λεπτά και είχα στη διάθεσή μου τέσσερα λεπτά. Όχι, όχι, διακόπτει ο πρόεδρος. Κύριε Αλμπερτίνη, έχετε τέσσερα λεπτά για τις δύο σας παρεμβάσεις, καταρχάς. Χρησιμοποίησατε δύο, έχετε το λόγο, θα δείξουμε μια κάποια ευελιξία, αλλά δεν θα ήθελα να φτάσουμε κάποια στιγμή και να μην σας ακούνε. Εγώ θέλω να εισακουστείτε, διότι αν σας δώσουμε άλλα πέντε λεπτά δεν θα σας ακούσει κανένας. Είχα έξι, είχα τέσσερα σε δύο. Τέλος πάντων, δεν θα προλάβω να πω αυτά που ήθελα να πω στα δύο λεπτά, επομένω δεν θα παρέμβω. Ευχαριστώ κύριε Αλμπερτίνη, ε, κρίμα που δεν σας ακούμε. Έχει το λόγο για δύο λεπτά ο κύριος Γκουαλτιέρη. Δεν σας ακούω, εκτός μικροφώνου γίνεται μια παρέμβαση από τον κύριο Ντερόσα. Κύριε Ντερόσα. Δυστυχώς δεν σας ακούω, δεν λειτουργεί το μικρόφωνο σας. Θέλετε να μου πείτε, λειτουργεί το. Ποτέ δεν λειτουργεί το μικρόφωνο όταν πατάω το κουνί. Θα μπορούσα να έχω εγώ τα δύο λεπτά του κύριου Αλμπερτίνη. Ο κύριος Γκουαλτιέρη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να είμαι ειλικρινή, νομίζω ότι ο πρόεδρο Αρμπερτίνη έχει δίκιο, διότι ω εισηγητή είχε στη διάθεσή του 4 λεπτά για την αρχική του παρέμβαση και 2 λεπτά για την απάντηση. Επιτρέψτε μου να σα υπενθυμίσω ότι λογικά θα έπρεπε να του δώσετε τα 4 λεπτά του να μιλήσει. Τέλο πάντων, για τη δική μου παρέμβαση τώρα, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια χρήσιμη και σημαντική συζήτηση γεγονό που αποδεικνύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ονομένο και διατεθειμένο να προσφέρει τη συνδρομή του σε μια εξωτερική δράση της Ευρώπης που θα είναι αποτελεσματική και συνεκτική. Δεν ακούσαμε μόνο επικρίσεις ε, για τα προφανή όρια τα οποία απόδειξε η Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, αλλά και κάποιε προτάσεις. Προτάσεις οι οποίε που περιλαμβάνουν και την προσφορά μιας ε, κάποιας μορφής εταιρικής ε, στρατηγικής σχέσης ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αξιόπιστος παράγων ε, στην ασφάλεια και στην άμυνα. Πρόκειται για προτάσεις οι οποίες είναι και καθόλου επίκαιρες διότι αν θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως βασική δυνατότητα για να πτύξει αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση την εξωτερική δράση το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία ε, και να υπάρχουν και κάποιες εξουσίες και ένας κατάλληλος προϋπολογισμός. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρούμε και κάτι για μια διακευουνευουλευτική ε, συνεργασία. Κάποια από τα πράγματα τα οποία προέκυψαν σαφώς είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει η συνθήκη από τη διαρθρωμένη συνεργασία, ακόμα και για το άρθρο 44, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να χωρίσουμε καθόκοντα διεξαγωγής μιας αποστολής από ένα κράτος μέλος, αλλά να ακολουθώντας τη ε, ε, ε, διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχουν συγκεκριμένε ε, δυνατότητε σε υπηρεσίες εξωτερικής δράσης και να αναδείξουμε και τον κατάλληλο ηγετικό ρόλο. Σα ευχαριστούμε για τη δέσμευσή σα για τι προτάσει που διατυπώσατε και καλό είναι να σκεφτόμαστε, όπω είπατε και εσεί ότι μια ομάδα μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα πράγματα, αλλά η Ευρώπη είναι μια μεγάλη πολιτική δύναμη που δεν θα πρέπει να αποφύγει τι ε, ευθύνε τη. Ευχαριστώ κύριε Γουαλτιαρή. Κύριε Αλμπερτίνη, θα ήθελα να σα ζητήσω να με συγχωρέσετε, ενημερώθηκα για το πώς ακριβώς ε, έγιναν τα πράγματα. Είχατε τέσσερα συν δύο, μιλήσατε 3 λεπτά στην αρχική σας παρέμβαση. 3 λεπτά λοιπόν, έχετε άλλα 3 λεπτά και θα δείξουμε και τη δέωση ευελιξία. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το όριο των 3 λεπτών. Έγινε μια κρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και υπήρξε και μια ερώτηση από κάποιο συνάδελφο προς την υπατή εκπρόσωπο η οποία έλεγε ότι όταν ο Κίσιγκερ επικρινόταν ε, για την ε, ε, πολιτική απομόνωση των ΗΠΑ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε ότι δεν υπάρχει κάποιο υπουργό εξωτερικών, ούτε και κάποιο αριθμό τηλεφώνου, στον οποίο θα μπορούσα να τηλεφωνήσω για να συνεργαστώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συνάδελφο ρώτησε, υπάρχει τώρα υπουργό εξωτερικών και ένα αριθμό τηλεφώνου, στον οποίο μπορεί να αποτανθεί είναι, απάντησε με το κλασικό σκοπτικό βρετανικό τη ύφου και είπε ότι ναι, εγώ είμαι, δεν είμαι υπουργό εξωτερικό, εγώ διεξάγω τα καθήκοντα του υπουργού και υπάρχει ένα αριθμό τηλεφώνου και απαντά ε, μία γραμματέα στο 1 στα αγγλικά, στο 2 στα γαλλικά, στο 3 στα γερμανικά και ούτω καθεξής. Κύριε εκπρόσωπε, ακούσατε τι φωνέ όλων μα και στην έκθεση μου ε, υπάρχει το μήνυμα θα εισακουστείτε καλύτερα στον κόσμο εάν ακούσετε καλύτερα και εμάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε να προωθήσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική και όχι μια πολιτική των κρατών μελών όπως κάνει το Συμβούλιο ούτε μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, την οποία ε, κάνει όταν πηγαίνετε κι εσείς ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να ε, καλύψετε τον τρίτο σας ρόλο που είναι εδώ πίσω από το έδρανο, διότι εσείς είστε κατά κάποιο τρόπο Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταλάβει το ρόλο μας ε, η ευρωπαϊκή κοινωνία θα πρέπει να ενισχυθεί ο δικός σας ρόλο καλύτερα και θα σας συνδράμουμε ώστε να διεξάγετε σωστά τα καθήκοντά σας. Ευχαριστώ και νομίζω ότι δεν κατασπατάλησα όλο με το χρόνο. Ευχαριστώ Ευχαριστούμε για την ε, ευγένειά σας και για την συνοπτικότητά σας. Η κυρία Μουνίθ Δεουρκίσο έχει το λόγο για δύο λεπτά. Επίσης, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Στο ΑΣΦΡΑΦ για το Ασράφ μάλλον δεν μπορούμε παρά να προσυπογράψουμε την καταγγελία για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά δεν πρέπει να συγχαίουμε σε καμία στιγμή την καταδίκη αυτή για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την πολιτική υποστήριξη για την κίνηση η οποία βρίσκεται στο στρατόπεδο Ασράφ. Υπάρχει μία πολιτική αντιπολίτευση η οποία εκπροσωπείται από στοιχεία της πράσινης κίνησης εκεί και εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να συγχαίουμε την υποστήριξη προς αυτά τα άτομα με την καταδίκη της ε, βίας επίθεσης κατά του Ασράφ. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω από την ε, Αντιπρόεδρο και υψηλή εκπρόσωπο να κοιτάξει και να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις των Μουζαχεντίν. Θα πρέπει να δείτε τι γίνεται κατά του πληθυσμού και να προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε τα θέματα ε, τα οποία επισημαίνουν οργανώσεις όπως το Human Rights Watch. Ε, όσον αφορά την εκθεσή σας κυρία Άστον, θα ήθελα να σημειώσετε ιδιαίτερα το σημείο υπαριθμών 6 που ζητά την εκπόνηση μιας λευκής βίβλου το η οποία θα επικεντρώνεται στο στρατογικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς ε, με την προοπτική του 2020. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές για τη συνεργασία που είχαμε για την εκπόνηση της έκθεσης αυτής και θα ήθελα να ε, πω ότι λυπάμαι που πολιτικά ε, πνεύματα ε, κακόβουλων ε, διαστάσεων δεν μου επέτρεψαν να αναφερθώ σε μια ακαδημική έκθεση που συνεισέφερε σε μια μελέτη για να αποτελέσει τη βάση της έκθεσης αυτής. Πρόκειται για μια έκθεση που ετοίμασε το ε, ε, Πανεπιστήμιο και αποτέλεσε καλή βάση για να συνεργαστώ με τους χειώδεις εισηγητές και ε, με τη Γραμματεία για την εκπόνηση της συγκεκριμένη έκθεσης που ελπίζω να βοηθήσει για τον καλύτερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μουνή. Θα ήθελα να πω στον κύριο Στίβενσον ότι στη συζήτηση αυτή αποφασίστηκε πριν έρθω εγώ εδώ να αναλάβω την Προεδρία να μην χρησιμοποιήσουμε την μπλε κάρτα για να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους και να φτάσουμε μέχρι το τέλος της συζήτησης. Θα ολοκληρώσουμε τώρα τη συζήτηση δίνοντας το λόγο στην αγαπητή μας φίλη την κυρία Κάθριν Άστον για να ε, απαντήσει σε όλες ως, τις παρεμβάσεις που είχαμε σε αυτή την μακροσκελέστατη συζήτηση. Έχετε το λόγο κυρία Άστον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στους βουλευτές ότι τους ευχαριστώ για όλα όσα είπαν. Κύριε Αλμπερτίνη, Όποτε, όπου θέλετε μπορώ να λάβω το λόγο. Για, θα μπορούσα να μιλήσω και από την ε, θέση του κύριου μιλητή εδώ προς τη μέση, αλλά δεν έχει σημασία. Οι εισηγητές σας νομίζω κατέληξαν στη δημιουργία πολύ χρήσιμων εκθέσεων για την υπηρεσία μου. Θα ήθελα όμως επίσης να πω ότι ότι ίσως υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια από ό,τι φαίνεται από τη συζήτηση αυτή. Έχουμε μια πολιτική με συγκεκριμένες και συνεπείς θέσεις. Από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέχρι του πώς αντιμετωπίζουμε την κρίση στη Μέση Ανατολή, δράσεις για τη Βοσνία, για την Αφρική, όπως το πρόβλημα που αρχίζει να λύνεται στην ακτή του ελεφαντοστού. Όλα αυτά τα έχουμε υπόψη μας και έχουμε μια συνεπή πολιτική. Το είπα και στους υπουργούς. Υπάρχει συνέπεια γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Βέβαια, ίσως να μην είμαστε πάντα σε θέση να πραγματοποιήσουμε όλα όσα θα θέλαμε, αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτά που έχουμε ήδη πετύχει. Θα ήθελα λοιπόν να αποτίσω ένα φόρο τιμή σε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση έστω και μερικοί των στόχων μας. Δεν μπορούμε όλα να τα έχουμε από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτή τη στιγμή έχουμε στείλει εκπροσώπους μας που μεταφέρουν τα μηνύματά μας σε ολόκληρο τον κόσμο και σχεδόν πάντα είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε δηλώσεις και λέμε τι θα θέλαμε να πραγματοποιηθεί. Για τις κυρώσεις κατά της Συρίας ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε μία άτυπη ακόμη πρόταση. Και είμαστε πάντοτε οι πρώτοι που όχι μόνο δηλώνουμε αλλά και προσπαθούμε να υλοποιήσουμε τις προτάσεις μας με συνέπεια. Η συνέπεια αυτή είναι κάτι το ιδιαίτερα ζωτικό που το τονίσατε κι εσείς. Κατά τη συζήτηση μιλήσαμε για συγκεκριμένα μέρη του κόσμου αλλά στη συνέχεια τα μέλη έθεσαν και άλλα προβλήματα που πρέπει και αυτά να τα θίξουμε. Ο κύριος Αλαφράνκα μας μίλησε για τους αντιφρονούντες στην Κούβα. Φυσικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Άλλοι μίλησαν για τη Γάζα, για την διασφάλιση της χορήγησης βοήθειας στο λαό της Γάζης, πράγμα το οποίο κάνουμε, αλλά πρέπει βέβαια να βελτιωθεί. Για το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία έχουμε, βρισκόμαστε σε συζητήσεις και συνεννοήσεις και με τους δύο με τη βοήθεια και της Γαλλίας με την για την Αλβανία έχουμε συζητήσει με τον Πρωθυπουργό και με την αντιπολίτευση για να αρχίσει κάποιος διάλογος και φυσικά για την Αφρική μιλήσαμε για δύο χώρες θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πολλές ακόμη στο Σουδάν ας πούμε αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι κάτι που δεν το αγνοούμε και η Ουκρανία σημαντική χώρα που γυτνιάζει με την Ένωση έχουμε Πολλή δουλειά. Το ξέρουμε όμως. Και θα ασχοληθούμε με όλα τα θέματα. Θα ήθελα να απομυθοποιήσω ορισμένα πράγματα πάντως. Εγώ δεν ζήτησα θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά καταφέραμε αυτά που καταφέραμε στον ΟΗΕ. Το αναγνωρίσατε κι εσείς. Δεν ήμουν η μόνη, αλλά πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχουμε και θέλουμε να πετύχουμε στην πολιτική εξωτερικής δράσης. Στη Λιβύα και μόνο καταφέραμε με τη βοήθεια που χορηγούμε να βοηθήσουμε 55.000 ανθρώπους. Και εγώ δεν ζήτησα απαγόρευση πτήσεων στο Συμβούλιο, όπως είπε κάποιος, εγώ είπα ότι ό,τι και να γίνει πρέπει να γίνει γρήγορα και αποτελεσματικά. Τώρα για τις αντιπροσωπείες μας. Στη Βενγάζη και στο Ιράκ ας πούμε. Δεν είναι ίδια η κατάσταση όπως στις Μπαχάμες. Στις Μπαχάμες εφαρμόζονται από καιρό προγράμματα της Κομισιόν και δεν είναι εναλλάξιμα οι Μπαχάμες με το Ιράκ ας πούμε. Καταλήγω όπως άρχισα. Δεν περιοριζόμαστε σε φιλοδοξίες. Θέλουμε συγκεκριμένους πόρους και υλοποίηση αυτών που ζητάμε. Και θα το πετύχουμε, αλλά σιγά σιγά. Αν μας βοηθήσουν όλες οι χώρες. Πολλές φορές θα πιέζουμε περισσότερο από άλλες, αλλά πάντοτε θα επιτυχάνομεν πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Άστον. Αγαπητοί συνάδελφοι, χάρη στην κατανόηση καταφέραμε να μην πέσουμε σε, στην ε, δυσμενή κατάσταση που βρεθήκαμε σε άλλες φορές, να μην μπορούμε να ακούσουμε τους τελευταίους ομιλητές που θα μιλούσαν τα τελευταία 10-15 λεπτά. Και ευχαριστώ όλους αυτούς που μας επέτρεψαν να κλείσουμε τη συζήτηση εγκαίρως και ζητώ κατανόηση από αυτούς που έκοψα το λόγο, τους έκοψα το λόγο γιατί ξεπέρασαν το λόγο τους, το χρονομιλία τους, το έκανα ακριβώς για να μπορέσω να επιτύχω να τελειώσει εγκαίρως η συζήτηση. Θα διακόψουμε για τρία ολόκληρα λεπτά για να, για να αρχίσει η ψηφοφορία στην κατάλληλη στιγμή.